All right. Um, appear to have got a full panel of uh, members of the European Parliament who are going to speak. Ας έχουμε εδώ τον, ε, τα ονόματα των Ευρωβουλευτών που επιθυμούν να μιλήσουν. Ας αρχίσουμε πρώτα με τους βουλευτές των Εθνικών Κοινοβουλίων ώστε να έχουν αρκετό χρόνο. Αυτό λοιπόν που θα ήθελα να κάνουμε είναι να ακούσουμε τους αγορητές που είναι ήδη παρόντες, δηλαδή η σειρά θα είναι κάπως διαφορετική από αυτήν. Α, παρακαλώ η Σιλβί που είναι. Sylvie, you're supposed to be up here. Ελάτε εδώ παρακαλώ, Σιλβί. Στο, στα έδρανα του Προεδρείου δηλαδή. Καλά λοιπόν. Ε, σας καλωσορίζω και πάλι όλες και όλους. Οι κύριοι Γκαλτιέρη και Μπροκ, Γκουαλτιέρη μάλλον και Μπροκ θα είναι παρόντες σήμερα. Είναι εκ των διαπραγματευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το λεγόμενο Fiscal Compact, την δημοσιονομική αυτή συμφωνία, που ήταν παρόντες και στο Συμβούλιο της 8ης-9ης Δεκεμβρίου, που απεφάσισε αυστηρότερη δημοσιονομική πειθαρχία, και αυτό βέβαια είναι το περιεχόμενο της συμφωνίας μεταξύ των 17 χωρών μελών της Ευρωζώνης, που όμως είναι ανοιχτή και σε, άλλους, και σε άλλες χώρες δηλαδή. Και σύμφωνα με αυτήν την συμφωνία θα επιβάλλονται κυρώσεις αυτομάτως σε χώρες οι οποίες ε, ξεπερνούν το 3% του ΑΕΠ σε έλλειμμα εκτός εάν μπλοκαριστεί η πορεία αυτή από ε, ειδική πλειοψηφία που προβλέπεται από ε, των άλλων χωρών μελών. Καθώς επίσης και το 0,5 του ονομαστικού ΑΕΠ. Και οι χώρες επίσης αναλαμβάνουν να εντάξουν το λεγόμενο χρυσό κανόνα απαγόρευσης δηλαδή ε, ελλημάτων στα εθνικά τους συντάγματα. Τα δε συμβαλόμενα μέρη έχουν συμφωνήσει να συνεργαστούν προς την κατεύθυνση μεγαλύτερης δημοσιονομικής ε, πειθαρχία και σύμφωνα με τα συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα που θα ψηφίσει τον Μάρτιο 2012 το Ερνό Συμβούλιο Κορυφής. Τώρα θα προχωρήσουμε σε ανταλλαγή απόψεων. Πρώτα δε θα παρακαλέσω τον κύριο Γκουαλτιέρη να κάνει μια σύντομη παρουσίαση του θέματος. Θα είδατε και χθες ότι ανακύπτουν ερωτήματα και στην περίπτωση αυτή που συμβεί και σήμερα, δηλαδή θα επανέλθω στους συζητητές του Κοινοβουλίου για να τους παρακαλέσω να απαντήσουν σε ερωτήσεις αυτές στο τέλος ε, της συζητήσεως. Και εάν κάτι παραμείνει θα προσπαθήσω να απαντήσω εγώ η ίδια. Ρομπέρτο, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρόκειται για σημαντικό θέμα και είναι πολύ σημαντική η συζήτηση αυτή για την Δημοσιονομική Συμφωνία για το Fiscal Compact με τους βουλευτές των χωρών μελών που θα είναι δηλαδή οι βουλευτές των αντισυμβαλόμενων μερών το Ευρωκοινοβούλιο συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις ως παρατηρητής στις διαπραγματεύσεις οι οποίες οδήγησαν στην σύναψη του ε, κειμένου που θα υπογραφεί στο επόμενο Συμβούλιο Κορυφής. Από πλευράς μας είχαμε επιλέξει μια προσέγγιση της, θα έλεγα, κριτικής προσέγγισης, κριτικής ε, δέσμευσης ή εμπλοκής. Με την έννοια ότι για μας αυτό το Fiscal Compact δεν είναι η καλύτερη λύση για ορισμένους από εμάς νομικά μιλώντας δεν ήταν καν αναγκαία αυτή η συμφωνία. Η Μεγάλη Βρετανία υπέβαλε βέτο ή πρόβαλε μάλλον σωστότερα και για το πρωτόκολλο 12 με την έννοια ότι μπορεί αυτό να τροποποιηθεί και εκεί θα χρειάζεται συμφωνία και λόγω αυτού χρειαζόταν αυτή η διακρατική συμφωνία. Πάντως εμείς θεωρούσαμε ότι θα καταστεί απαραίτητη μια αναθεώρηση των συνθήκων. Τα τελευταία χρόνια δηλαδή έχει διαπιστωθεί ότι το σύμφωνο σταθερότητας είναι υπερβολικά αδύναμο. Περιλάμβανε κάποιες βασικές προϋποθέσεις, αλλά αυτές χρειάζονται ακόμα συζήτηση. Βέβαια, έχουμε ήδη τις έξι ε, οδηγίες, τα έξι μέτρα Όπως είπα λοιπόν, το Σύμφωνο Σταθερότητας και Αναπτύξεως ενισχύθηκε σημαντικά με το λεγόμενο six-pack. Γι' αυτό είναι θέμα εάν τα προβλήματα που γνωρίζουμε και από το παρελθόν, δηλαδή ότι τελικά χώρες μέλη δεν τηρούν τα συμφωνηθέντα. Αν, αν θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αυτό και έτσι τώρα. Λοιπόν, εμείς έχουμε ασκήσει σημαντική κριτική για το λόγο ότι η συμφωνία αυτή ήταν απλά διακρατική, διακυβερνητική και θεωρούμε ότι δεν είναι απαραίτητο να γίνει κάτι τι το νέο. Επικρίσεις επίσης ε, που ενισχύονται από την ιδέα ότι η ευθύνη για τον προϋπολογισμό είναι μια απαραίτητη προϋπόθεση, ένας όρος απαραίτητος αλλά όχι επαρκής. Και άρα κατά την κρίση μας υπάρχει επίγουσα ανάγκη για παρέμβαση αλλά και για ανάπτυξη και για αλληλεγγύη. Αλλά γι' αυτά δεν θα σταθώ σε αυτά μάλλον, γιατί προτιμώ να σταθώ στην συνθήκη. Γιατί η προσέγγιση μας ήταν επικριτική, αλλά ήταν και ε, η προσέγγιση μιας δέσμευσης, engagement. Παράλληλα με άλλα κοινοτικά όργανα και διάφορες κυβερνήσεις, θεωρούμε ότι συμβάλαμε στη βελτίωση του κειμένου αυτής της συνθήκης και ότι καταφέραμε να αποφύγουμε τον κίνδυνο που στο πρώτο σχέδιο ήταν πολύ έντονος μια συνθήκη που κατά κάποιο τρόπο θα όριζε ένα είδος παράλληλης διακυβέρνηση διαφορετικής από αυτήν την κοινοτική σε μια μάλλον ταυτόχρονα πιο άκαμπτη αλλά και περισσότερο, που δίνει και περισσότερη διακριτική ευχέρεια, δηλαδή ανεπαρκής. Στο τελευταίο λοιπόν κείμενο, στο τελικό κείμενο της συνθήκης παραμένει μια σειρά από προβλήματα, αλλά συνολικά πρέπει να πω ότι το τελικό κείμενο δεν καθορίζει, ε, δεν περιλαμβάνει αυτό τον κίνδυνο. Είναι ένα κείμενο το οποίο κατά κάποιο τρόπο είναι αρκετά, αν και όχι απόλυτα, αρκετά ε, συνεκτικό και συνεπές παραπληρωματικό με την υπόλοιπη νομοθεσία της Ένωσης και άρα ε, και με το ρόλο των θεσμικών οργάνων. Είναι ένας ρόλος αυτός, θα θέλω να το πω αυτό γιατί ίσως αυτό και από μόνο τον αποτελέσει θέμα συζήτησης, είναι ένας ρόλος που αυτή τη στιγμή μπορεί να θεωρηθεί νόμιμος ακριβώς επειδή δεν είναι ένας ρόλος που βασίζεται σε διαφορετικές δεσμεύσεις από αυτές που ορίζονται από την νομοθεσία. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο η συνθήκη σήμερα δεσμεύει τα εθνικά κράτη-μέλη να σέβονται την ε, κοινοτική νομοθεσία και τον τρόπο με τον οποίο ερμηνεύεται από τα ίδια τα όργανα της ε, Ένωσης ε, που, τους, ε, που έχουν αυτή την αρμοδιότητα μια αρμοδιότητα την οποία ασκούν που δεν τους αποδίδεται όμως από την ίδια τη συνθήκη. Σε σχέση με τα κράτη αυτά έχουν επιπλέον δεσμεύσεις που οφείλονται, απορρέων μάλλον από τη δική τους εσωτερική νομοθεσία. Αυτό δεν ίσχυε αρχικά ήταν ξεχωριστές αρμοδιότητες. Δεν ήταν πάντως ρόλος της κοινότητας. Μπάς περιπτώσει δεν ε, ξέραμε ακριβώ ποιο έπρεπε να υποπτεύει την ε, εφαρμογή της εσωτερικής νομοθεσίας σε σχέση με τη συνθήκη. Όπως γνωρίζετε, ο πυρήνα της συνθήκης είναι το άρθρο 3. δηλαδή το άρθρο που μας δεσμεύει να εισάγουμε κατά προτίμηση σε συνταγματικό επίπεδο και αυτή είναι επίσης ουσιαστική τροποποίηση διότι δεν πρόκειται πλέον για υποχρέωση ε, τροποποίησης του συντάγματος αλλά μόνο για μια επιλογή που θεωρείται προτιμητέα. Και από νομική άποψη δεν υπάρχει τέτοια κατηγορία προτιμά, προτιμητέο το τάδε. Μπορεί να το κάνει ή δεν μπορεί να το κάνει. Ε, αυτό σημαίνει ότι εναπόκειται στην διακριτική ευχαίρεια του κάθε κοινοβουλίου. Άρα λοιπόν υποχρεούνται ναι μεν στο ισοζύγιο, στον ισολογισμό συγγνώμη, ε, που όμως στη συνθήκη διευκρινίζεται καλύτερα. Μιλάμε για διαρθρωτικό ισολογισμό, δηλαδή όχι για λογιστικό ισολογισμό. Και άρα πλέον όχι για ετήσιο έλλειμμα, όπως προηγουμένως προβλεπόταν στα απορίσματα της διάσκεψης κορυφής της 3ης ε, Δεκεμβρίου, αλλά για μεσοπρόθεσμο στόχο, που είναι η κατηγορία που χρησιμοποιείται για την κοινοτική νομοθεσία. Άρα, Πρόκειται για ένα στόχο που ορίζεται από την Κομισιόν. Άσχετα από τη συνθήκη. Ήδη το κάνει αυτό η Κομισιόν. Άρα λοιπόν δεν πρόκειται για νέα αρμοδιότητα από αυτήν την έννοια για την Κομισιόν. Υπάρχει εκείνο το άρθρο, το, εκείνο το 0,5 που, που θεωρείται ως maximum διαρθωτικό έλλειμμα. Ενώ στην αρχή ήταν το 1% αλλά στην ουσία αυτό έχει λιγότερη σημασία από ό,τι νομίζουμε για δύο λόγους. Καταρχήν γιατί στην πράξη αυτό το 0,5 ισχύει για τις χώρε που είναι κάτω από το 60% το χρέο τους. Άρα για το six pack ούτως ή άλλως ε, μιλάμε για μείωση του χρέου περισσότερο ε, από, μάλλον κάτω από το 1%. Ενώ εδώ τώρα έχει μπει στη συνθήκη ότι για μια χώρα ε, Τη οποία το χρέο είναι... Συγγνώμη, τα διμπέρδεψα, λέει ο μιλήτης. Εκείνες που έχουν κάτω από 60% μπορούν να φτάσουν μέχρι το 1% χρέο. Ε, συγγνώμη, ε, ποσοστό του ΑΕΠ. Εδώ λέει ότι θα στηριχτεί η πρόταση της Κομισιόν να περάσει στο 0,5% το νούμερο του κοινοτικού στον κοινοτικό κανονισμό. Όταν θα γίνει αυτό θα έχουμε απόλυτη σύμπτωση ανάμεσα στις παραμέτρους του άρθρου 3 και της ε, κοινοτική νομοθεσίας. Και αυτό θα θέσει το πρόβλημα δηλαδή θα έχουμε συγκεκριμένα νούμερα, συγκεκριμένα όρια ή θα έχουμε κινητά όρια Δηλαδή διαρθωτικά ελλείμματα που ορίζονται από την κοινοτική νομοθεσία που μπορεί να αλλάξει στο μέλλον και άρα θα αλλάζουν και οι παράμετροι κάθε φορά. Και να θέσω άλλο ένα θέμα που σχετίζεται με το ε, με την αιτιολογική σκέψη που αφορά το ESM, τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Δηλαδή, ε, Δηλαδή, πότε μια χώρα δεν μπορεί να ζητήσει χρηματοδότηση από τον μηχανισμό σταθερότητας ένα χρόνο μετά από την επικύρωση και ένα χρόνο μετά από την εφαρμογή της μεταρρύθμισης της συνταγματικής νομοθεσίας ή μη συνταγματικής νομοθεσίας, ενισχυμένης νομοθεσίας και ε, από την ε, χρήση του μηχανισμού διόρθωσης. Αυτά τα δύο χρόνια είναι το ανώτατο όριο και αυτά θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όταν θα ορίζονται οι προθεσμίες για την επικύρωση φυσικά. Άρα λοιπόν σας καλώ να σκεφτείτε και αυτή την πτυχή. Θα είχα κι άλλα να πω, πολλά να πω για τις σχέσεις με τα εθνικά κοινοβούλια που διευκρινίστηκαν καλύτερα στην διατύπωση του άρθρου 13 και φυσικά για τις διατάξεις που αφορούν τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου όπου προστίθεται και μια ρύθμιση, ένα arrangement που θα εγκριθεί στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Αλλά επ' αυτού βεβαίως είμαστε έτοιμοι να επανέλθουμε στον γύρο των απαντήσεων. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, Ρομπέρτο. Πέντε λεπτά υποτίθεται έπρεπε να μιλήσεις, αλλά είναι αδύνατο να μιλήσει κανείς για όλα αυτά μέσα σε πέντε λεπτά. Θα δώσω τώρα το λόγο στον Έλμαρ Μπροκ, που ήταν ένας άλλος εκπρόσωπος του Κοινοβουλίου στις διαπραγματεύσεις. Κυρία Πρόεδρε, <clears throat> κυρίες και κύριοι, θα κάνω λίγες μόνο συμπληρωματικές παρατηρήσεις. Μία από τις παρανοήσεις που συχνά ακούγεται στην συζήτηση είναι ότι όσοι επινόησαν την ε, συνθήκη αυτή το έκαναν για να επιλύσουν την κρίση. Αυτό είναι παρανόηση διότι η συνθήκη αυτή δεν μπορεί να επιλύσει την κρίση ούτε είχε και ποτέ την πρόθεση αυτή. Δεν πρόκειται παρά μόνο για ένα ακόμη βήμα ή αν θέλετε ένα ακόμα λίθο στην προσπάθεια αυτή, στο χτίσιμο αυτό δηλαδή του δρόμου που θα οδηγήσει σε μια προσπάθεια πύλης της λύσης με τις έξι οδηγίες, με το ευρωπαϊκό εξάμεινο, με όλα τα άλλα συναφή μέτρα. Και υπήρχαν δύο ή τρία θέματα τα οποία δεν ήταν δυνατόν να επιληθούν υπό την ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας. Διότι η συνθήκη της Λισαβόνας είτε δεν λέει τίποτε, είτε λέει το αντίθετο από αυτό που πάμε να κάνουμε, σε ό,τι αφορά τις νομικές βάσεις δηλαδή. Είναι και το θέμα αυτό του golden rule, του χρυσού κανόνα, όπου πρέπει να πούμε ότι είναι η δέσμευση των χωρών μελών να μεταφέρουν τον κανόνα αυτό στις εθνικές τους νομοθεσίες. Και αυτό δεν έχει καμία σχέση καταρχήν με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Αυτό η επιθυμία εδώ είναι κάθε χώρα να είναι υποχρεωμένη κατά πόριαν του δικού της δικαίου να τηρήσει τα συμφωνηθέντα και υπεσχημένα, διότι ας μην λησμονούμε ότι η Γερμανία και η Γαλλία πρώτες παραβίασαν το σύμφωνο σταθερότητας και αναπτύξεως. Τώρα, ο αυτοματισμός των κυρώσεων. Προεκοσαετία στι διαπραγματεύσει για τη συνθήκη του Μάστριχτ δεν ήταν δυνατόν να περάσει κάτι τέτοιο. Ούτε επίση το 1997 στο Σύμφωνο Σταθερότητας και Αναπτύξεως. Αυτός ο αυτοματισμός των κυρώσεων απορρίφθηκε τότε διότι δεν είχε συνειδητοποιηθεί ακόμα πόσο μεγάλο ρόλο θα έπαιζε η εθνική κυριαρχία στο θέμα αυτό. Υποτίθεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημαίνει τις παραβιάσεις από πλευράς χωρών μελών και μπορεί να ανατραπεί ο αυτοματισμός των κυρώσεων μόνο εάν θεωρήσει μια πλειοψηφία των χωρών μελών ότι δεν πρέπει να επιβληθούν. Ωστόσο, μέχρι τώρα αυτοματισμός των κυρώσεων δεν έχει λειτουργήσει. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτός ο αυτοματισμός είναι σημαντικό βήμα πρόοδου. Επίσης, στη συνταγματική συνθήκη είχε προτείνει δική μου πολιτική ομάδα, το Λαϊκό Κόμμα, το 2002, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να είναι αρμόδιο και για θέματα της νομισματικής ένωσης. Όμως επ' αυτού δεν επετεύθη τότε το 2002 συνένεση. Εμείς τότε το είχαμε αιτιολογήσει αυτό λέγοντας ότι μόνο εφόσον μπορεί να γίνει προσφυγή ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου γίνεται αξιόπιστη τότε η τήρηση των διατάξεων του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Δεν μπορούσε κανείς βέβαια να φανταστεί ότι τα πράγματα θα πήγαιναν τόσο άσχημα που θα φτάσουμε στο σημερινό, στη σημερινή κατάσταση. Τώρα λοιπόν δίδεται και αυτή η δυνατότητα με την Δημοσιονομική Συμφωνία. Όπως δηλαδή δεν τηρεί τις δεσμεύσεις μπορεί να αχθεί ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου του ε, Λουξεμβούργου. Και βέβαια η συνθήκη την οποία μιλούμε, το Fiscal Compact, δεν είναι κοινοτική συνθήκη. Πώς είναι δυνατόν τότε κοινοτικό όργανο, όπως το δικαστήριο και η Κομισιόν βέβαια που εμπλέκεται, να δραστηριοποιηθούν για συμφωνία, για να τη, τη συμφωνία, η οποία δεν είναι κοινοτική. Αυτό εδώ θα χρειαστεί βέβαια το πρόβλημα με κάποιο τρόπο να λυθεί. Η λύση που σκέπτονται είναι στην βάση διαπιστώσεων της Κομισιόν να κινητοποιείται ένας αριθμός χωρών μελών ή μία χώρα μέλος και να προσφεύγει. Ή να ανατίθεται η εντολή στην Τρόικα του Συμβουλίου δηλαδή, προηγούμενη παρούσα και επόμενη Προεδρία, να προσφεύγουν αυτές στο δικαστήριο. Εδώ θέλω να πω καθαρά ότι τα δημοσιονομικά μέτρα εξετάσεων των προϋπολογισμών δηλαδή. Για θέματα προϋπολογισμού οφείλουν να σέβονται βέβαια την κυριαρχία των Εθνικών Κοινοβουλίων, αλλά ο σκοπός είναι η πρόληψη μελλοντικών κρίσεων και η υπέρβαση τούτης εδώ, που σημαίνει ότι θα χρειαστούν σημαντικές διαρθρωτικές αλλαγές για να ανέλθει η ανταγωνιστικότητα των εθνικών οικονομιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να υπάρξει ανάπτυξη. Αλλιώς τα ποσά που διατίθεται δεν έχουν επενδυτικό χαρακτήρα εφόσον δεν υπάρχουν απαραίτητες διαρθρώσεις. Αν λοιπόν αυτή, όταν μάλλον αυτή η δημοσιονομική συμφωνία θα είναι πλέον ασφαλής, θα έχει εγκριθεί δηλαδή, θα είναι απαραίτητο να σκεφτούμε πλέον για διαρθρωτικές αλλαγές και διαρθρωτικές αλλαγές με στόχο την ανάπτυξη. Βλέπω εδώ κοντά μας και τον πρόεδρο Αλάν Λαμασούρ που πιστεύω ότι θα συμφωνήσει μαζί μου ότι τα διαρθρωτικά πλέον ταμεία τότε πρέπει να επανέλθουν στην πραγματική τους αποστολή. Διότι προ 18 ετών επινοήθηκαν τα διορθωτικά ταμεία για να διευκολύνουν την ενιαία αγορά. Ενώ στην πραγματικότητα ήταν στην, στην αρχή η αποστολή τους να ενισχύσουν τις περιφέρειες, ώστε να γίνουν αυτές ανταγωνιστικές. Και τα χρήματα που θα προβλέπονται 350 με 360 δισεκατομμύρια, δηλαδή 50 δισεκατομμύρια το χρόνο για την επόμενη δημοσιονομική περίοδο. Είναι σημαντικά κονδύλια αυτά, είναι σημαντικό ποσό εντό εισαγωγικών ευρωπαϊκής αλληλεγγύης που θα κατευθυνθεί προς χώρες και περιφέρειες. Ορισμένα από τα ωραία πράγματα που επενδύσαμε, που χρηματοδοτήσαμε μάλλον μέχρι τώρα από τα διευθυντικά ταμεία, θα πρέπει να τα αφήσουμε. Και να φροντίσουμε ώστε μέσω αυτών να απαλληλθούν οι διαφορές και οι ανισότητες μέσα στην ενιαία αγορά, ώστε οι πιο αδύναμες χώρες να γίνουν πιο ισχυρές και να αποκατασταθεί η απαραίτητη ισορροπία εντός της Ευρωπαϊκής Ενιαίας Αγοράς. Ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε. Ευχαριστώ πολύ. Να δώσω το λόγο στον κύριο Τζένς Τζόλ της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου της Δανίας. Και θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι έχω λάβει μόνο τέσσερα έντυπα ε, αιτήματος λόγου και μάλιστα από το Ηνωμένο Βασίλειο μόνο. Εάν θέλετε να μιλήσετε, παρακαλώ συμπληρώστε τα έντυπα και υποβάλλετε τα στο Προεδρείο. Ο Τζένς έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι μεγάλη χαρά για μένα που βρίσκομαι εδώ και έχω την ευκαιρία να συμμετάσχω σε έναν, ελπίζω, επικοδομητικό διάλογο για την καινούργια συνθήκη. Έχω εργαστεί εδώ για πάρα πολλά χρόνια και είμαι υπέρμαχος της ευρωπαϊκής ιδέας. Πιστεύω όμως ότι δεν έχουν πιστεί όλοι οι Ευρωπαίοι ακόμα Βασικές μου παρατηρήσεις είναι οι εξής. Πρώτον, για να ξεπεράσουμε την κρίση χρειαζόμαστε περισσότερα από δημοσιονομική πειθαρχία και κατά δεύτερο λόγο θα πρέπει οι ευρωβουλευτές και μέλη εθνικών κοινοβουλίων να εστιάσουν την προσοχή τους ε, σε κοινούς στόχους. Ενώ θα πρέπει το Κοινοβούλιο να ε, εμπλακεί περισσότερο ε, στην διαδικασία λήψης αποφάσεων. Η Δανία δεν έχει υιοθετήσει το ευρώ, ωστόσο θα προσχωρήσει στη νέα δημοσιονομική συμφωνία, θα τηρήσει όλες τις διαστάσεις της συμφωνίας που, δεν, που είναι διαθέσιμες ε, για τα κράτη-μέλη που δεν έχουν το ευρώ, θα υιοθετήσει βεβαίως το χρυσό κανόνα και θα τον εφαρμόσει κατά γράμμα. Είμαστε κάπως διαφορετικοί, αλλά τασόμαστε δίπλα σε όλους. Έχουμε την εξάδα των μέτρων, την επόμενη διάδα των μέτρων, το Europlus Pact, τη Δημοσιονομική Συμφωνία και ακόμα δεν έχουμε οργανώσει τη συζήτηση σε εθνικό επίπεδο για τους δείκτες ε, περί μακροοικονομικών ανισορροπιών. Χρειάζεται να εστιάσουμε την προσοχή μας και στο θεσμικό πλαίσιο και στις πολιτικές πολιτικές. Η δημοσιονομική πειθαρχία είναι προϋπόθεση, αλλά δεν είναι λύση αυτή. Για να ξεπεράσουμε την κρίση θα πρέπει να δημιουργήσουμε θέσεις απασχόλησης. Πολλοί συνάδελφοι το έχουν επαναλάβει πολλές φορές. Όταν ο Τζόσεφ Στίγκλιτς, ο καθηγητής οικονομίας επισκέφθηκε στη, τη Δανία είπε ότι στην ιστορία δεν έχουμε παράδειγμα ε, που να έχει ξεπεραστεί μια κρίση χωρίς τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και χωρίς την ύπαρξη νέων επενδύσεων. Θέλουμε να εφαρμόσουμε κανόνες για δημοσιονομική πειθαρχία, αλλά θα πρέπει αυτό να πηγαίνει τέρι, με τέρι, χέρι με χέρι με τις επενδύσεις και την ανάπτυξη. Μιλήσαμε χθε για τα ομόλογα έργων. Θα πρέπει να συγκεντρωθούν νέα κεφάλαια. Χαίρομαι διότι οι αρχικοί κρατών και κυβερνήσεων στρέφουν επιτέλους την προσοχή τους ε, στο θέμα της απασχόλησης. Στα τέλη του Ιανουαρίου πρώτη φορά και συμφώνησαν να διοχετευτούν περισσότερα χρήματα για την επίλυση αυτών των προβλημάτων μπορούμε να δημιουργήσουμε θέσεις απασχόλησης χωρίς να φτιάξουμε καινούργια ταμεία και καινούργια χρηματοδοτικά εργαλεία. Έχουμε ένα σωρό οδηγίε πάνω στις οποίες μπορούμε να στηριχθούμε. Έχουμε την οδηγία για την ενεργειακή αποδοτικότητα. Θα οδηγήσει σε 2 εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης. Θα έχουμε 4% ως ποσοστό του ΑΕΠ περισσότερα έσοδα εάν προχωρήσουμε τα θέματα της ε, πράσινης ενέργειας. Έχουμε επιβάλει στους Έλληνες ε, φίλους μας πολύ αυστηρά μέτρα, αλλά μπορούμε να τσακωνόμαστε για ε, ολόκληρους μήνες για το ποια θα είναι η έδρα του Ευρωπαϊκού Γραφείου για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας. χρειάζεται περισσότερος ε, συμβιβασμός, περισσότερες προσπάθειες από όλους. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος ε, και ο μόνος δρόμος που θα πρέπει να ακολουθήσουμε. Η Προεδρία της Δανίας έχει παρουσιάσει τις προτεραιότητές της για την εσωτερική αγορά, για μια πιο πράσινη Ευρώπη, για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, το οποίο αποτελεί και ασφαλιστική δικλίδα για την επίτευξη των στόχων της Ευρώπης για το 2020 βασιζόμαστε ήδη σε υφιστάμενη νομοθεσία. Δεν χρειαζόμαστε καινούργια νομοθετικά πλαίσια ε, αλλά πρέπει να υιοθετήσουμε και να εφαρμόσουμε αυτά που έχουμε ήδη συμφωνήσει. Χρειάζεται να εκτελεχθεί ένας ε, κοινός διάλογος, δημόσιος διάλογος ε, που δεν στον οποίο δεν θα πρέπει να συμμετάσχουν μόνο τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Με την καινούργια συνθήκη θα χρειάζεται περισσότερο διάλογο μεταξύ Εθνικών Κοινοβουλίων, Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το μοντέλο ε, εφαρμογής όλων αυτών στην πράξη εξαρτάται από τις ανάγκες κάθε Εθνικού Κοινοβουλίου. Οι διαδικασίες είναι διαφορετικές. Βάσει του άρθρου 13 προβλέπεται αυτός ο διάλογος ε, όσον αφορά στη συζήτηση για τις δημοσιονομικές πολιτικές. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο. Ωστόσο, τα Εθνικά Κοινοβούλια θα πρέπει να επικοινωνούν άμεσα και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προς το θέμα της ετήσιας μελέτης ανάπτυξης και τις ειδικέ συστάσεις της Επιτροπής για την εκάστοτε χώρα. Νομίζω ότι οι συνάδελφοι στην ΚΟΣΑΚ ε, θα τα αναλάβουν όλα αυτά. Επόμενα ο βήμα μας πρέπει να είναι όχι μόνο η δημοσιονομική πειθαρχία, αλλά η προσοχή στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και η ολοκλήρωση της εξέτασης των ε, υφιστάμενων οδηγιών. Λίγο λιγότερα εθνικά συμφέροντα και λίγο περισσότερη εθνική εμπλοκή από όλους μας και συμμετοχή είναι αυτό που μας χρειάζεται, πιστεύω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η Σιλβία έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη γιατί ήδη οι συνάδελφοι με έχουν καλύψει. Τρεις εκπροσώπους ακούσαμε από, τον, ε, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο τρίτος ήταν ο Κίφερ Χόφσταπτ από το Άλντε και εγώ ήμουν εισηγήτρια για το θέμα της ε, δέσμης 6 μέτρων για το six Ο Ροπέρτο και ο Έλμαρ το το είπαν άλλωστε, δεν πρέπει να έχουμε προσδοκίες από τη συνθήκη ε, που δεν ήταν στο, στη διατύπωση του περιεχομένου όταν ο Μάριο Ντράκη ήρθε εδώ στις αρχές Δεκεμβρίου ε, για να συζητήσουμε για το θέμα της Δημοσιονομικής Συμφωνίας, θυμάμαι ε, τα λεγόμενά του. Όντως είναι χρήσιμη η Δημοσιονομική Συμφωνία για να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να συνεχίσει να λειτουργεί σωστά, ε, ειδικότερα όσον αφορά στις χώρες που δεν θέλουν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να ξεπεράσει την εντολή που της έχει δοθεί. Έχει σημασία αυτό το κείμενο αλλά δεν έχει και υπερβολικά μεγάλη σημασία. Με αυτό κλείνει ο κύκλος ε, της συζήτησης για τη δημοσιονομική πειθαρχία και μένει πολλής δρόμος να καλύψουμε. Θέλω να επιμείνω στο εξής. Καταρχάς, το θέμα της συλλογική μας αξιοπιστίας. Από τη στιγμή που βρισκόμαστε μεταξύ μας, πρόσωπο με πρόσωπο, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς, να μην μιλούμε με υπονοούμενα. Ε, σημειώνεται μια δυσκολία. Αν προσπαθούμε να πείσουμε όλους τους επενδυτές ε, παγκοσμίω ότι έχουμε νεονόμισμα, ότι είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε προς τα εμπρός, ε, ότι είμαστε έτοιμοι να πάρουμε όλες αυτές τις κοινωνικές και οικονομικές αποφάσεις που ταιριάζουν με την ύπαρξη ενός ενιαίου νομίσματος, τότε θα πρέπει να δεχθούμε μια πολύ πιο δυναμική σε όριση της έννοιας της εθνικής κυριαρχίας. Με την ε, δημιουργία του ενιαίου νομίσματος το 1992 έχουμε μπει πλέον ε, σε μια νέα πολιτική εποχή και όλα τα κράτη-μέλη που δεν έχουν ακόμα υιοθετήσει το ευρώ αλλά θέλουν να μπουν έχουν υιοθετήσει πολύ ισχυρές, πολύ έντονες πολιτικές δεσμεύσεις και θα πρέπει λοιπόν να μην κάνουμε μόνο μεταρρυθμίσεις στο θεσμικό πλαίσιο, αλλά να μεταρρυθμίζουμε και να αλλάζουμε την ε, συμπεριφορά μας. Το να έχουμε ενιαίο νόμισμα και να συζητούμε για το ότι τίποτα δεν θα αλλάξει, νομίζω ότι δεν έχει πολύ νόημα. Ε, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων θα πρέπει να μπορεί να παρέμβει για να ε, αποφανθεί επί αυτών των θεμάτων. Ε, το να λέμε ότι δεν μπορεί το Δικαστήριο να παρέμβει σε θέματα δημοσιονομικής συμφωνίας, γιατί η δημοσιονομική συμφωνία δεν είναι καθεαυτή κοινοτική, αλλά είναι διακυβερνητική, νομίζω ότι δεν βοηθάει. Δεν βοηθάει κυρίως τη συλλογική μας αξιοπιστία. Όσο πιο περίπλοκα είναι τα συστήματα αποφάσεων, τόσο λιγότερο θα πείθουμε τους ξένους επενδυτές για την αξιοπιστία μας προκειμένου να εμπιστευτούν στο δικό μας νόμισμα της αποταμιεύσης των συνταξιδοτικών ταμείων μεταξύ άλλων. Εγώ θεωρώ ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες είναι ενήλικοι. Δεν θα πρέπει ε, να τους πείσουμε ότι τα παλιά πράγματα θα μείνουν όπως έχουν απαράλεκτα. Ε, το θέμα είναι να δώσουμε σωστές απαντήσεις και να τους προσφέρουμε απασχόληση, θέσεις απασχόλησης και ανάπτυξη. Αν κάποιοι δεν θέλουν να προσχωρήσουν στο ευρώ, καλώς είναι δική τους επιλογή να μην μπουν. Αν όμως έχουν εθετήσει το ευρωπαϊκό νόμισμα θα πρέπει σίγουρα να αλλάξουν τη συμπεριφορά τους. Εκτός λοιπόν από το θέμα της συλλογική αξιοπιστίας θα ήθελα να μιλήσω και για το θέμα της δημοκρατίας. Το θεμελιώδες ερώτημα που εγείρεται αυτή τη στιγμή είναι το εξής. Πώς θα ε, πείσουμε τον πολίτη ότι η γνώμη του έχει βαρύτητα στις αποφάσεις που λαμβάνονται καθημερινά. Όταν ε, συνέρχεται το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Σίγουρα το κάθε μέλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου έχει εθνική νομιμότητα αδιαφυσβήτητη αφού είναι εκλεγμένος αρχηγός. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι το όργανο συλλογικά έχει νομιμότητα. Δεν υπάρχει επαρκής δημόσια διαβούλευση. Απουσιάζει έλεγχος αν θέλετε ε, και εποπτεία ε, τον, του θεσμικού οργάνου το οποίο αποφασίζει αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Και μπορεί να ακούγεται ταμπού αυτό, αλλά εγώ τολμώ να το θίξω αυτό το θέμα. Στη Γαλλία έχουμε μια φοβερή προεκλογική εκστρατεία αυτή τη στιγμή για τις προεδρικές εκλογές και δεν γίνεται λόγος επαρκής για την Ευρώπη. Στη Γαλλία αυτή τη στιγμή στην προεκλογική εκστρατεία μόνο οι ευρωσκεπτικιστές παίρνουν το λόγο, έχουν κυριοαρχήσει στο δημόσιο διάλογο. Μας λένε λοιπόν ότι όσοι εκλέγονται σε εθνικό επίπεδο φτάνουν μετά στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχουν την εντολή, υποτίθεται να αποφασίζουν. Από πού τους δόθηκε. Τους δόθηκε εθνική εντολή. Και άλλωστε κάποιοι από αυτούς έχουν εκλεγεί πριν ξεσπάσει η κρίση και χωρίς να έχουν λύσεις για την κρίση. Δεύτερο θέμα, ε, τρίτο θέμα μετά τη δημοκρατία είναι το θέμα της εξωτερικής διάστασης. Δηλαδή, ε, οι αποφάσεις που λαμβάνονται σε ένα κρατομέλος να μην έχουν φρικτές συνέπειες ε, ή επιρροές σε άλλο κράτος μέλος, χωρίς οι πολίτες του δεύτερου κράτους μέλους να έχουν τη δυνατότητα να εκφραστούν. Και να σας δώσω το εξής παράδειγμα ε, της μισθολογικής ανταγωνιστικότητας, αν θέλετε. Ε, οι επιπτώσεις στους μισθούς και στην απασχόληση. Είναι πράγματα που πλήττονται από αποφάσεις που μπορεί να ληφθούν σε μια άλλη χώρα τα θέματα των μισθών. Τι θα κάνουμε για να το καταπολεμήσουμε αυτό. Στην δέσμη 6 μέτρων έχουμε ένα καινοτόμο στοιχείο της μακροοικονομικής ισορροπίας π.χ. Ε, τι μπορούμε να κάνουμε περισσότερο σε αυτό το θέμα. Θα σταματήσω κάπου εδώ λέγοντας ότι ε, ε, μένει πάρα πολύ μεγάλη απόσταση να καλύψουμε. Δεν έχουμε φτάσει καθόλου στο τέλος. Στην αρχή είμαστε είχαμε την αίσθηση ότι η δημοσιονομική πειθαρχία θα αρκούσε για να μην υπάρχει ή για να ξεπεριστεί η κρίση. Αυτό βεβαίως δεν ισχύει. Ελπίζω να έχουν πιστεί όλοι γι' αυτό. Δεν έχουμε μια επαρκή δημοκρατική προσέγγιση. Και ένας δεύτερος κίνδυνος είναι ότι μπορεί τελικά να καταλήξουμε να σώσουμε το ευρώ, αλλά σε αυτή τη μάχη να έχουμε χάσει ε, όλους τους Ευρωπαίους πολίτες από, ε, και την υποστήριξή τους. Ευχαριστώ. Η Πρόεδρος, και εγώ σας ευχαριστώ να, μιλήσουμε, να ακούσουμε τώρα όσους θέλουν να υποβάλουν κάποιο ερώτημα ε, με σειρά υποβολής ερωτήματος. Θα ήθελα να ζητήσω από όλους τους ομιλητές να μην ξεπεράσουν τα τρία λεπτά. Όσοι θέλουν να υποβάλουν ερώτηση να μην ξεπεράσουν τα τρία λεπτά για να μπορέσουν να απαντήσουν στη συνέχεια και οι εισηγητές. Και ενδεχομένως να υποβληθούν και άλλα ερωτήματα στη συνέχεια. Bill Cash από το Ηνωμένο Βασίλειο, James Clatison από το Ηνωμένο Βασίλειο επίσης. Ε, είναι οι πρώτοι που μου υπέβαλαν αίτημα για ερώτηση. Ναι, λέει ε, η Σιλβία, αλλά θα μπορούσατε να λάβετε υπόψη σας ε, το θέμα ότι όσοι κάνουν ερώτηση καλό θα ήταν να ανήκουν και στη ζώνη του ευρώ επίσης. Η πρόεδρος, εγώ είμαι η πρόεδρος και καθορίζω τη σειρά, Σλοβανία, Σλοβενία, μετά Λουξεμβούργο, μετά θα ακούσουμε την Περβάνς Μπερές, Λίντα Χάρισον από το Ηνωμένο Βασίλειο, τον κύριο Τζορτζέτη από την Ιταλία και τον κύριο Ντόναχιου από την Ιρλανδία. Μπιλ Κάσου, λοιπόν, από το Ηνωμένο Βασίλειο. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ο Έλμαρ μας λέει ότι η συμφωνία θα προσφέρει τους κανόνες, δηλαδή το χρυσό κανόνα, για να τους υπακούν τους κανόνες οι διάφοροι άνθρωποι. Το κατανοώ αυτό. Ωστόσο, πάρα πολλές αμφιβολίες υπάρχουν ως προς την αμιμότητα αυτής της συμφωνίας της δημοσιονομικής. Και αν ως Ευρωπαϊκή Κοινότητα ή ως Ευρωπαϊκή Ένωση θα ξεκινήσουμε ε, με βάση μια υπόνοια ότι μπορεί να υπάρχει εξαναγκασμός τήρησης κανόνων, ε, βάση μιας διαδικασία η οποία υπονομεύει το κράτος δικαίου, τότε, ε, αν θέλετε, δυναμητίζονται τα θεμέλια της βιωσιμότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κυρία Μέρκελ είπε χθε ότι δεν ήθελε και ότι δεν, πρέπει, δεν θα ήθελε να πάρει περισσότερα ρίσκα από ό,τι χρειάζεται. Και η συνάδελφος από την Γαλλία είπε ότι η δημοκρατία είναι απαραίτητη για την όλη διαδικασία. Το κράτος δικαίου εξαρτάται από την δημοκρατία. Και για διάφορους λόγους που δεν θέλω να τους αναλύσω, να πω παρενθετικά ότι ο, κύριο, ο καθηγητής Πολ Κρέγκερ έχει κάνει μια πολύ διδακτική παρουσίαση στη δική μας Επιτροπή ως προς το θέμα της, νομοθε... της νομιμότητας αυτής της συνθήκης και λέει, παραθέτω, είναι σημαντικό ε, να εξετάσουμε κατά πόσο η συνθήκη δίδει νέες λειτουργίες σε υφιστάμενα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Εγώ πιστεύω ότι αυτό αντιβαίνει και αντίκειται στις υφιστάμενες ευρωπαϊκές συνθήκες και το τεκμηριώνει με 11 σελίδες μετά. Δηλαδή, εγείρονται σοβαρά ερωτήματα Είχαμε από πριν και το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Το βασικό ερώτημα είναι το εξής. Αυτό το οποίο συμβαίνει ε, γίνεται για λόγους ε, μετακίνησης προς μια περισσότερη Ευρωπαϊκή Ένωση όπως και το άρθρο, εξού και το άρθρο της Vivian Redding της προάλλες Wall Street, στη Wall Street Journal. Περισσότερη Ευρώπη με καταναγκασμό περί αυτού πρόκειται και είναι κάτι το οποίο ε, επηρεάζει όλους αν θέλετε. Δεν μπορεί κανείς να πει ότι ε, ε, δεν είμαστε εμείς μέλη αυτής της συμφωνίας ω Ενωμένο Βασίλειο, άρα δεν έχουμε λόγο. Βεβαίως και έχουμε λόγο και μπορούμε να σχολιάσουμε αυτή τη ε, συμφωνία, γιατί αυτή η συμφωνία αλλάζει ε, το ρόλο των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μεταξύ άλλων. Σε αυτό το πλαίσιο θα ήθελα να πω ότι είναι εξαιρετικά επικίνδυνο, είναι μια πολύ επικίνδυνη κατηφοριά ε, στην οποία θα κατρακυλήσουμε εάν πούμε ότι όλα αυτά είναι απολύτως νόμιμα, διότι η νομιμότητά τους αμφισβητείται και τίθεται εν κινδύνο. Και ε, σε μια επιστολή που συνέταξε πριν από λίγες μέρες ο πρέσβης του Ηνωμένου Βασιλείου ε, και την, απευθύνει, την στη γραμματεία του Συμβουλίου ε, τονίζει ότι εμείς είμαστε εκτός αυτής της συμφωνίας όχι μόνο για το City του Λονδίνου, όχι μόνο για θέματα ενιαίας αγοράς, αλλά γιατί αυτή η συνθήκη ε, ε, δυναμητίζει τα θεμέλια της ε, δημοκρατικής νομιμότητας. Είναι πολύ περισσότερα υπησέρχονται εκεί. Και μου φαίνεται αδιανόητο να υπάρχουν άνθρωποι σε αυτή την αίθουσα που δεν έχουν καταλάβει ότι είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που επηρεάζει την καθημερινότητά τους, τους ψηφοφόρους τους, ε, τις ζωές τους, συνταγματικές αλλαγές επιβάλλονται στην κάθε χώρα ε, και στον λαό με την υπηγραφή αυτής της ε, μη νομότυπης συμφωνίας. Ευχαριστώ. Ο Τζέιμς Κλάπισον από το Εμένο Βασίλειο. Κύριε Πρόεδρε, υπήρξαν κάποιες διαμαρτυρίες ε, όσον αφορά τη σειρά. Ε, προς το συμφέρον της, διεθνής, της αρμονίας, εγώ ευχαρίστως να υποβάλω την ερώτηση μου αργότερα, αν κάποιος άλλος θέλει να πάρει τη θέση μου. Εγώ είμαι ευχαριστημένη με τη σειρά των ερωτήσεων και εσείς είστε ο επόμενος στη σειρά. Μάλιστα, εφόσον λοιπόν δεν δημιουργείται δυσαρέσκεια και δυσαρμονία, έχω εγώ τρία ερωτήσεις. Πρώτον, θεωρείτε αυτή την συμφωνία διεθνή συμφωνία ή κοινοτική συμφωνία. Δεύτερον, για τις προτάσεις περί ρήξης, ε, νομίζω είναι το άρθρο 8 του Συμφώνου, είναι άποψή σας ότι η Κομισιόν κρύβεται πίσω από αυτές τις προτάσεις περί παράβασης και κοινή αυτές διαδικασίες ή τα μεμονωμένα κρατημέλη. Και γιατί στο άρθρο αυτό υπάρχει αυτή η παράξενη διαδικασία όπου η Κομισιόν ξεκινά, αλλά τα κράτη-μέλη στη συνέχεια θα ε, πρέπει να φέρουν ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου την υπόθεση. Ποια είναι η αιτιολόγηση για αυτήν εδώ την παράξενη μορφή. Και τέλος, τι συμβαίνει και όλοι ελπίζουμε πως θα καταφέρουμε να έχουμε τη σταθερότητα, την ανάπτυξη, τις θέσεις απασχόλησης και τα λοιπά, αλλά τι συμβαίνει σε σχέση με την εθνική δημοκρασία αν οι περιστάσεις σε μια συγκεκριμένη χώρα ή ομάδα χωρών, τη απουσία μεμονωμένης πολιτικής παρακολούθησης και υποπτίας και μεμονωμένο με ενιαίο νόμισμα δεν μπορούν να ανταγωνιστούν. Οι οικονομίες τους αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα, έχουν ελλείμματα και δεν είναι σε θέση να τηρήσουν τις απαιτήσει του συμφώνου χωρίς να δημιουργούν όλα ένα και υψηλότερα ελλείμματα με μειούμενα φορολογικά έσοδα. Υπάρχουν όρια για το πόσο ψηλά μπορεί να φτάσει η ενεργεία, πόσο ψηλά μπορεί να φτάσει η ενεργεία των νέων, πόσο θα επιβληθεί λιτότητα σε κάθε χώρα. Αυτά όλα θα σημειωθούν. Ήδη τα εξ απλά ισχύουν άσχετα από τις συνθήκες που επικρατούν σε κάθε χώρα και ποιες είναι οι απόψεις ε, του εκλογικού σώματος της εν λόγω χώρας. Ο κύριος Ιτσέλη από τη Σλοβενία. Ευχαριστώ <clears throat> κύριε Πρόεδρε. Λίγα λόγια για την δημοσιονομική αυτή συμφωνία, καθώς επίσης και τη δημοσιονομική πειθαρχία, όπως περιγράφεται στο έγγραφο που συζητούμε σήμερα. Κατά τη γνώμη μου, το κύριο μήνυμα του εγγράφου εμφανίζεται στο άρθρο 3, πρώτη παράγραφο, που λέει ότι οι χώρες μέλη οφείλουν να έχουν ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς. Δηλαδή, με άλλα λόγια, οι χώρες μέλη δεν μπορούν να δαπανούν περισσότερα από όσα παράγουν. Μάλιστα ακόμα περισσότερο. Λέει ότι ανεύθυνος δανεισμός δεν μπορεί να αποτελεί το θεμέλιο για παραπέρα ανάπτυξη. Το μόνο θεμέλιο για παραπέρα ανάπτυξη μπορεί να αποτελεί μια ανταγωνιστική οικονομία η οποία να παράγει απασχόληση, η οποία να παράγει ανάπτυξη και τίθεται και το θέμα της ανεργίας βέβαια εδώ που είναι πάρα πολύ επίκαιρο. Κατά τη γνώμη μου λοιπόν οι χώρες μέλη αντιμετωπίζουν, έχουν μπροστά τους δηλαδή μια σημαντική στρατηγική απόφαση να λάβουν που αυτή τη στιγμή βέβαια καλούνται να λάβουν χώρες πολλές οι οποίες βρίσκονται σε φάση δημοσιονομικής εξυγίανσης πως τόσο δεν μπορεί να αποτελεί αυτό σκοπό. Θα πρέπει να συνοδεύεται από καινοτομία, μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα και μάλιστα και σε σύγκριση με ασιατικές χώρες και τις ενομένες Πολιτείες. Εν συντομία δηλαδή, οι μελλοντικέ ευρωπαϊκές γενναίες δεν θα μπορούν να αναπτυχθούν στη βάση δανεισμού. Θα πρέπει να στηρίζονται στις δικέ του αναπτυξιακέ δυνάμει. Πολλές χώρες που σήμερα είναι βαθιά χρεωμένε και οφείλω να ομολογήσω ότι μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται και η Σλοβενία. Τα τελευταία χρόνια διπλασιάστηκε το χρέος μας και έχει φτάσει σχεδόν το 50% του ΑΕΠ μα, ενώ πριν από τρία χρόνια μόλις ανήρχεται στο 24%. Όλες αυτές οι χώρες λοιπόν αντιμετωπίζουν τώρα νέες προκλήσεις νέα καθήκοντα και οι επόμενες γενναίες θα πρέπει να εξηγιάνουν τα δημόσια οικονομικά. Άρα πρέπει να μειωθούν οι δημόσιες δαπάνες. Για το 2012 οι δημόσιες δαπάνες πρέπει να μειωθούν ώστε το έλλειμμά μας να κατέβει και το δικό μας δηλαδή στη Σλοβενία στο 3% που τώρα είναι στο 5,6% και βέβαια και ο χρυσός κανόνας που θα πρέπει να περιλάβουν στα, τους, στα συνταγματά τους μάλλον οι χώρες, θα αποσκοπεί στην εξισορρόπηση μεταξύ ε, χρέους και ανάπτυξης. Στρατηγικά μιλώντας πιστεύω ότι ο δρόμος αυτός είναι ο σωστός και για την χώρα μου, τη Σλοβενία και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλέξ Μποντρού από το Λουξεμβούργο. Ευχαριστώ. Δύο παρατηρήσεις. Πρώτα για τη δημοσιονομική συνθήκη και για το χρυσό κανόνα δεύτερον. Για τα δημόσια οικονομικά είναι προφανές ότι απαιτείται, απαιτούνται κοινή στόχοι καθώς επίσης και η εργαλειοθήκη που θα μας επιτρέπει να τα παρακολουθούμε αυτά και προληπτικά και κατασταλτικά. Θεωρώ πάντως ότι θα πρέπει να είναι εθνική επιλογή ο καθορισμός των τρόπων ε, της επίτευξης των στόχων αυτών. Θα πρέπει λοιπόν αυτό να παραμείνει στην εθνική αρμοδιότητα και επομένω των εθνικών βουλών. Δεν σας κρύβω κάποια ανησυχία που αισθάνομαι ότι δηλαδή αυτή η ανακατανομή καθηκόντων, αρμοδιοτήτων με την παρέμβαση της Κομισιόν και του Συμβουλίου που ρίχνουν όλο και περισσότερο βάρος ε, στους τρόπους με τους οποίους θα πρέπει να γίνει η δημοσιονομική εξυγένση. Το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρεμβαίνει στην διαδικασία αυτή δεν μειώνει ωστόσο δεν απαλύνει ας πούμε καλύτερα την μείωση της επιρροής των εθνικών βουλών. Είναι χρήσιμο να γίνουν ανταλλαγέ απόψεων μεταξύ Ευρωβουλευτών και Εθνικών Βουλευτών σχετικά με τον τρόπο που μεταφέρονται αυτά τα πράγματα στις εθνικές νομοθεσίες και από την ε, άποψη των Εθνικών Βουλών αλλά και για τα νέα κείμενα και για το ΣΥΚΣΠΑΚ αλλά και για την ε, Διακρατική Συμφωνία. Τώρα, για τον χρυσό κανόνα. Χαίρομαι που παρετήθηκαν τελικώ οι κυβερνήσει από την ιδέα τη υποχρεωτική εγγραφή στα εθνικά συντάγματα του κανόνα αυτού. Πρώτα-πρώτα, εμένα με απασχολεί πολύ η υποτιθέμενη, προστιθέμενη αξία αυτού του κανόνα. Και το Σύμφωνο Σταθερότητα και Αναπτύξεω που ήταν διεθνή συμφωνία και έχει επομένω υπερσυνταγματική ε, ισχύ ήδη καθορίζει στην ουσία τον κανόνα αυτό. Τι νόημα έχει τώρα να μπει και στα εθνικά συντάγματα. Δεύτερο, μια τέτοια προστιθέμενη αξία στη Γαλλία ή στη Γερμανία παράδειγμα. Εκεί οφείλει να γίνεται, ε, γίνεται μάλλον έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων. Δεν μπορεί τώρα να επιβάλλει νέο συνταγματικό έλεγχο η Ευρωπαϊκή Ένωση τη εφαρμογή των κανόνων αυτών δηλαδή. Χρειάζεται λοιπόν κάποια ευκαμψία για την μεταφορά των, του κανόνα αυτού στην εθνική νομοθεσία. Η, η θα προκληθεί μεγάλη σύγχυση. Χαίρομαι λοιπόν εν τέλει όπως είπα που εγκαταλείπεται η ιδέα αυτή και που επιτέλους ε, υπερισχύει η ε, λογική. Ευχαριστώ πολύ. Υποτίθεται ότι θα είχαμε παρέμβαση της, ε, του εισηγητή της ε, Επιτροπής Απασχόλησης που δυστυχώς δεν μπόρεσε να προσέλθει. Θα δώσω τώρα το λόγο ε, στον πρόεδρο της, την πρόεδρο συγγνώμη, της Επιτροπής Απασχόλησης, δηλαδή την κυρία Περβάνος Μπερές. Σας ευχαριστώ. Δεν παίρνω το λόγο ως πρόεδρος της Επιτροπής Απασχόλησης, αλλά προσωπικά. Όταν βλέπει κανείς την ιστορία της Ευρωζώνης, οι εμπειρογνώμονε και οι προσεκτικοί παρατηρητές δεν περίμεναν το 2007 και την έκρηξη της κρίσης ε, για να διαπιστώσουν ότι με τους κανόνες που είχαμε ορίσει, με το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξη, δεν λειτουργούσαν κατά την καλύτερη δυνατή κατάσταση τα πράγματα, για να τα πούμε έτσι ε, ε, ελαφριά. Από τις αρχές του 2007, δηλαδή όταν κάναμε τον απολογισμό των 10 ετών λειτουργίας του ευρώ, σαφώς ε, ορίστηκε ότι παρά το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης που θα έπρεπε να μας είχε χρησιμεύσει ως χρυσός κανόνας, ε, παρατηρούσαμε αποκλίσεις ανταγωνιστικότητας, ανταγω... αποκλίσεις μακροοικονομικές μέσα στην Ευρωζώνη που καθιστούσαν μη λειτουργική την υπόθεση αυτή. Σήμερα, αφού έχουμε αφού οι θύνοντες έχουν αποκομίσει τα διδάγματα αυτής της κατάστασης, τουλάχιστον σε όσα αποκαλούνται οικονομικό πακέτο το six pack, το εξαπλό πακέτο δηλαδή, την εξισορρόπηση του δικαιώματος στην τελειότητα. Γι' αυτό και ακριβώς πολλοί από εμά δεν υπερψηφίσαμε όλα τα στοιχεία του εξαπλού πακέτου, αλλά εν πάση περιπτώσει υπήρχε από τη μια πλευρά η ενίσχυση του κανόνα, σε μια, σε μια νέα φάση ενίσχυσης και έπειτα ε, ε πολλά στοιχεία εξισορρόπησης για να ληφθούν υπόψη μακροοικονομικές ανισορροπίες. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο, η αναγνώριση των αποκλήσεων και των δυσκολιών που είχαν διαπιστωθεί στο διάρκεια των 10 πρώτων ετών λειτουργίας του ευρώ. Έπειτα θα πρέπει να δούμε ότι υπάρχει μια νέα ισορροπία η οποία υποτίθεται μάλλον θα υπήρχε ανάμεσα στο χρυσό κανόνα και στην ε, μακροοικονομία. Ενώ εμείς τώρα θέλουμε να συνταγματικοποιήσουμε αυτό τον ε, χρυσό κανόνα. Και έπειτα, θα πρέπει να δούμε και ακούω τους ε, Βρετανούς συνάδελφους. Εγώ λυπάμαι που οι Βρετανοί δεν ε, υπογράφουν το κείμενο, αλλά να πω ότι ο όρος που είχαν θέσει οι Βρετανοί για να ε, συμμετέχουν, για να υπογράψουν το κείμενο, ήταν απαράδεκτος, γιατί αγγίζει τη λειτουργία, τη δυνητική λειτουργία του Ευρωζώνης. Δηλαδή να αποκλείονται από την νομοθεσία για τα πιστοτικά θέματα. Και έπειτα, όταν βλέπουμε σε ποιου απευθύνεται αυτό το κείμενο. Δεν νομίζω ότι αυτό το κείμενο απευθύνεται στην Ελλάδα ή στην Ιρλανδία ή στην Πορτογαλία, γιατί προφανώ κανεί δεν χρειάζεται τέτοια συνθήκη για να εφαρμόσει σε αυτέ τι χώρε κανόνε που είναι εξαιρετικά, εξαιρετικά ε, αυστηροί Άρα λοιπόν υπάρχει ένα πολιτικό διακύβευμα εδώ, πολύ σημαντικό για διάφορα Και πολλοί το είπαν χτε. Και ορισμένοι το επανέλαβαν και σήμερα το πρωί. Η ισορροπία που πρέπει να αναζητήσουμε στο πλαίσιο της Ευρωζώνης ανάμεσα σε μια απαραίτητη πειθαρχία αλλά και ένα κοινό μέλλον δεν είναι ε, ε θεσπισμένη μέσω αυτής της συνθήκης. Το άρθρο 1 αναφέρεται στην λέξη ανάπτυξη, αλλά με μια λογική πάντοτε ίδια, γιατί θα έχετε... Επειδή θα έχετε τηρήσει την δημοσιονομική πειθαρχία, επειδή θα έχετε αποκαταστήσει τους δημόσιους λογαριασμούς σας, θα έρθει και η ανάπτυξη. Ακριβώ το ίδιο είναι όπω όταν μα λέει η Κεντρική Τράπεζα ότι η καλύτερη συμβολή τη κοινωνισματική πολιτική στην πολιτική ανάπτυξη είναι η τήρηση τη σταθερότητα των τιμών. Ε, οι ευρωπαϊκές οικονομίες σε όλα μας τα κράτη και συλλογικά έχουν ήδη πληρώσει πολύ βαρύ τίμημα για αυτό το χρυσό κανόνα που δεν δημιουργεί θέσεις απασχόλησης και ανάπτυξη. Εδώ ποιο είναι το διακύβευμα για αυτήν εδώ τη συνθήκη, την επικύρωσή της και τις ε, προϋποθέσεις για την εξισορρόπησή της. Δεν έχω το χρόνο να πω παραπάνω πράγματα, θα πω ίσως κάποια στα συμπεράσματα πράγματα ακόμη, αλλά θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στο τι λέμε. Όταν χρησιμοποιούμε τις λέξεις ανάπτυξη και απασχόληση και θεσπίζουμε αυτή την, την συνθήκη, τον χρυσό κανόνα και την υποτιθέμενη ισορροπία. Υπάρχει έλλειψη ισορροπίας και το ξέρουμε αυτό εδώ και χρόνια για την Ευρωζώνη και ειδού και τα αποτελέσματα είναι προφανή. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, να φέρω και πάλι ότι η κυρία Μπερές ε, μας είπε τη δική της προσωπική άποψη και ότι δεν πρόκειται για την γενική άποψη της Επιτροπής για να αποφευθούν οι παρεξηγήσεις. Τώρα πάω στον κύριο Χάρισον από το Ηνωμένο Βασίλειο. Εγώ μιλώ εξ ονόματος τη Βουλής των Λόρδων και τη Ειδική Επιτροπής ε, Ρωμόδης για τα θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης Ότι όλα τα, εκπροσωπώ όλα τα πολιτικά κόμματα που ε, συμμετέχουν σε αυτήν την επιτροπή. Στις, το Μάρτιο του 2010 ενεγκρίθη η πρόταση για το εξαπλό πακέτο μέτρων ε, και ο Υπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων ανέκρινε και το Ευρωπαϊκό Εξάμενο που κατά τη γνώμη μου αποτελεί τη συνέχεια των Εβραίων ε, Οικονομικών Κατευθυντηρίων Γραμμών και έπειτα έχουμε και ε, σε δύο εβδομάδες ε, ε, μέσα σε δύο εβδομάδες κάνει μια άλλη έκθεση, ανάλυση της δημοσιονομικής συνθήκης που βελτιώνει την δυνατότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ανταποκριθεί στις, προτα... στις, στις ανάγκες. Και συμφωνώ με τον Έλμαρ Μπρόκ ότι θα πρέπει να επανέλθουμε στα διευθυντικά ταμεία και με τον Δανό συνάδελφο που έδειξε το παράδειγμα, έδωσε το παράδειγμα ενίσχυση της ενιαίας αγοράς σε αυτή την περίπτωση με τις, ε, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Τώρα, φυσικά συμφωνούμε με τη βοήθεια που δίνεται στην Ελλάδα. Θα θέλαμε Συμφωνούμε μάλλον με, τον, ε, με την προστασία και με την ανακεφαλοποίηση των τραπέζων, όχι όμως μέσω της ε, αντιστροφής του εισμόχλευσης, γιατί έτσι θα είχαν λιγότερες δυνατότητες για ανάπτυξη. Ε, γιατί δεν υπογράψαμε. Εμείς ε, ρωτήσαμε την κυβέρνηση στην Ειδική Επιτροπή γιατί δεν υπέγραψε την Δημοσιονομική Συμφωνία. Δεν ξέρουμε αν ήταν για την προστασία της ενιαίας αγοράς, για τις, ε, τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες στο Λονδίνο, φόβος της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής, φόβος του, για το φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Πάντως, εμείς στη Βουλή των Λόρδων καταλήξαμε στο πορίσματα ότι δεν υπήρχε λόγος να μην υπογράψουμε αυτή τη συνθήκη και θα ήθελα να το κατανοήσετε. Αυτή ήταν ε, η ομόφωνη άποψη της Επιτροπής μας ε, στην Βουλή των Λόρδων. Έχουμε δημοσιεύσει διάφορες εκθέσεις ε, και για τις, τους αξιολόγηση αξιολόγησης ικανότητα. ικανότητας. Φοβούμεθα όμως ότι και αν εκεί υπάρξει ένας ευρωπαϊκός τέτοιος οργανισμός δεν θα φτάσει για να κάνει αυτή τη δουλειά. Δημοσιεύσαμε την άποψή μας για έναν εποπτικό οργανισμό, για τον, ε, την άποψή μας για τον φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, καθώς και για το δημοσιονομικό πλαίσιο το οποίο προβλέπουμε για το 2014-2020. Πολλές ιδέες βελτιώνουν εκεί την ενιαία αγορά και αναζωογόνηση της, ε, της εσωτερικής αγοράς θα είναι πολύ σημαντική. Αυτές οι εκθέσεις είναι διαθέσιμες από τον εκπρόσωπο της Βουλής των Λόρδων εδώ, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε εκπρόσωπό μας και ελπίζω να τις ζητήσετε και να τις μελετήσετε. Σας ευχαριστώ. και τώρα εκπρόσωπος της Ιταλίας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η Ιταλία κινήθηκε προβλέποντας την Δημοσιονομική Συμφωνία, ιδιαίτερα όσον αφορά τη συνταγματική μεταρρύθμιση που, συν, που, που περιλαμβάνει τον ισοσκελισμό του προπολογισμού, τον χρυσό κανόνα δηλαδή, ε, στο Σύνταγμα και τον επόμενο μήνα θα έχει ήδη ενταχθεί στο Σύνταγμά μας αυτός ο κανόνας. Ωστόσο δεν νομίζω πως όλα τα προβλήματα έχουν λυθεί. Γι' αυτό και η πρώτη επαλήθευση θα έπρεπε να γίνει πριν ακόμα την, τον κάνουν οι, οι ευρωπαϊκές αρχές, οι εθνικές αρχές που, επαληθεύουν ε, τους προϋπολογισμούς. Ε, αλλά αυτή η πτυχή δεν είναι σαφής και γι' αυτό και ε, συνδέομαι και με την παρέμβαση του συναδέλφου από το Λουξεμβούργο. Ποια είναι τα όργανα που μπορούν να παρέμβουν σε αυτή τη φάση, δηλαδή συνταγματικό δικαστήριο και ελεγκτικό συνέδριο. Και επίση θα ήθελα να έχω την άποψή σα για το ποιο θα μπορούσε να είναι ένα ανεξάρτητο οργανισμό που στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 3 θα πρέπει να υποπτεύει, να παρακολουθεί τα μέτρα επανένταξη σε σχέση με την απόκληση από του στόχου, του συμπεφωνημένου μεσοπρόθεσμου στόχου. Είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό. Στην συνταγματική μεταρρύθμιση που εμείς εγκρίναμε προβλέπουμε τη δημιουργία ενός ε, ανεξάρτητου οργανισμού υπό την αιγίδα του Κοινοβουλίου. Μια προσωπική τώρα παρατήρηση σε σχέση με την έννοια της δημοκρατίας και της συμμετοχής ε, στις αποφάσεις. Η εμπειρία η προσωπική μου από το Ιταλικό Κοινοβούλιο εδώ και χρόνια είναι ότι ε, γενικά υπάρχει συμφωνία και υπερψήφιση των συνθηκών ε, που έρχονται από την ε, Ευρώπη, αλλά δεν γίνεται βάθυνση μέσα στο, μέσα στο Εθνικό μας Κοινοβούλιο. Όταν συζητάμε για αυτά τα θέματα, τα κάνουμε έτσι ανάμεσα στους συναδέλφους που ασχολούνται με αυτά τα θέματα. Δεν υπάρχει μεγάλη συμμετοχή από τους υπόλοιπους συναδέλφους. Ο μόνος τρόπος για να φέρουμε στη κοινή γνώμη τα σπουδαία αυτά θέματα και τα θέματα κυριαρχίας που προκύπτουν μέσω των συνθήκων είναι μέσω των δημοψηφισμάτων. Αν και στο Σύνταγμα το Ιταλικό δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο. Νομίζω πως θα πρέπει να βρούμε την μέθοδο ώστε με κάποιο τρόπο να συμμετέχουν οι λαοί στη λήψη αυτών των αποφάσεων. Διαφορετικά, θα βλέπουν ε, ε, τον Ευρωπαϊκή Ένωση μόνο όταν έρχονται και επιβάλλονται αυτά τα δρακόντια ε, μέτρα από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση ή όταν αυξάνουν τη φόρη. Σα ευχαριστώ. Ο επόμενο ομιλητή ο κ. Ντόνεχιου από την Ιρλανδία και έχω λάβει άλλα δύο αιτήματα. Οπότε μετά τον κύριο Ντόνεχιου κύριος Λία Μουόντογκ και ο κύριος Πίντ από την ε, Πορτογαλία. Ο κύριος Ντόναχιο, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Τρεις ερωτήσεις, παρακαλώ για τους ε, εισηγητές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η πρώτη μου ερώτηση έχει σχέση με τα προβλήματα των, δημοσίων, των εθνικών δημοσίων οικονομικών. Δεν είναι αλήθεια ότι τα προβλήματα των διαφόρων χωρών μελών στα δημόσια οικονομικά τους δηλαδή. Αυτά ούτως ή άλλως θα πρέπει να επιληθούν ανεξαρτήτως του αν θα υπάρχει αυτό, το fiscal compact ή όχι. Και όταν μια χώρα αντιμετωπίζει κρίση στα δημοσιονομικά της, μια μικρή οικονομία ας πούμε όπως η Ιρλανδική, προτιμώ να βρίσκομαι σε μια κατάσταση όπου οικειοθελώς μοιράζομαι την εθνική μου κυριαρχία με τα κοινοτικά όργανα παρά με τις αγορές. Νομίζω ότι είναι στρατηγική η επιλογή αυτή και μια στρατηγική επιλογή που έχει λόγο να αναλάβει κανείς. Είναι χρήσιμο να αναλάβει κανείς δηλαδή για την προστασία των συμφερόντων των πολιτών. Τώρα για τις μακροοικονομικές ανισορροπίες που ε, ε, προσπαθούν να επιλύσουν οι έξι οδηγίες. Το ίδιο σημαντικό είναι να εγκύψουμε και σε αυτά, όπως και στα μέτρα κατά του χρέους και, της, και του ελλείμματος. Γιατί σε μεγάλο βαθμό η δημοσιονομική κρίση που αντιμετωπίζουν σήμερα οι, χώρες, οι χώρες είναι λήψη ισορροπίας στις, στα ισοζύγια πληρωμών τους και μέσα στις ίδιες τις οικονομίες τους. Και εκεί έγκυται το πρόβλημα. Και το τρίτο μου ερώτημα είναι για τους μεσοπρόθεσμους στόχους, το τρίτο τμήμα της ε, συνθήκης. Εάν μια χώρα βρίσκεται σε κατάσταση όπου κινείται προς την επίτευξη του μεσοπρόθεσμου στόχου της, συμφωνεί με δράσεις και μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν, τα κάνει όλα αυτά και μετά λόγω εξωτερικών παραγόντων αποτυγχάνει στον στόχο της για το έλλειμμα. Ποιος είναι ο ρόλος τότε των κυρώσεων. Διότι πιστεύω ότι πολλές χώρες θα ανταποκριθούν, θα εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, αλλά λόγω εξωτερικών επιρροών θα είναι πολύ δύσκολο για αυτές να ε, σεβαστούν πραγματικά τον στόχο του ελλείμματος που έχουν δεχθεί και έχουν υπογράψει. Και εκεί νομίζω αυτό στερεί την νομιμότητα από το κείμενο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πολλοί Βρετανοί συναδελφοί πήραν το λόγο, γνωρίζουν ότι ε, ο χρυσός κανόνας που ήταν ενδιαφέροντας ε, μέσα στην ιστορία της οικονομίας ήταν σίγουρα ο χρυσός κανόνας της Βρετανίας που ίσχυε μέχρι το 2004 και που τότε απέκλειε τις, δαπάνες, ε, τις δημόσιες δαπάνες επενδύσεων από τον υπολογισμό του δημοσίου ελλείμματος. Και όταν θα κάνουμε το πραγματικό απολογισμό της περίοδου Τόνι Μπλερ θα διαπιστώσουμε πως ο ισολογισμός ήταν, προπολογισμό ήταν καλός, κυρίως γιατί υπήρξαν μαζικές επενδύσει στι δημόσιε ε, υποδομές, ε, ελήφθησαν δεσμεύσεις στην υγεία και στην ε, παιδεία και επιπλέον η Κεντρική Τράπεζα παρενέβη μαζικά για να νομισματοποιήσει το δημόσιο έλλειμμα και να αποφύγει τι εντάσει στις ισοτιμίες, χωρίς να, στα επιτόκια, χωρί να ξεχνάμε μια πολιτική ισοτιμιών ε, συναλλαγματικών ισοτιμιών που επέτρεψε στη Βρετανία, που δεν είναι στο ευρώ, να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά τη. Εγώ κατανοώ του Βρετανού φίλου που παραμένουν επιφυλακτικοί σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, που η Κεντρική Τράπεζα δεν μπορεί να παρέμβει με τέτοιο τρόπο. Και όπου ο χρυσό κανόνα που μα προτείνουν σήμερα είναι εξαιρετικά περιοριστικό. Και μόνο οι αγαθοί μπορεί να πιστεύουν πως ο περιοριστικός χρυσός κανόνας που περιλαμβάνεται στη συνθήκη Μερκοζή θα μας επιτρέψει να μειώσουμε τα ελλείμματα, να, ξαν... να αναζωογονήσουμε την ανάπτυξη και να αυξήσουμε την απασχόληση. Δεν φτάνει, επειδή τα λέμε αυτά δημοσιονομική εξυγίανση και απασχόληση και ανάπτυξη, επειδή λέει αυτές τις λέξεις ένα κείμενο, σημαίνει ότι μαγικά θα γίνουν όλα αυτά. Αυτά τα λένε διάφορα κείμενα εδώ και 10 χρόνια και τα είπε και η Περβάνς Μπερέζ. Εδώ και 10 χρόνια χειριστήκαμε τις δαπάνες. Εκτός από την περίοδο που συγκυριακά υποβαθμίστηκαν λόγω κρίσης το 2009, οι δημόσιες δαπάνες και οι κοινωνικές δαπάνες ήταν υπό σε όλα τα κρατημέλη. Αυτό εξηγεί την αύξηση των ελλημάτων. Αυτό που εξηγεί την αύξηση των ελλημάτων ήταν ξεκινήσαμε την αύξηση των φόρων για τις χθεσινές μελλοντικέ γενιές και αυτό οδήγησε στην βάθηση του χρέους και φτάσαμε σε αυτό που λέμε ε, διαρθωτικό έλλειμμα. Τώρα, σε σχέση με αυτή τη διαρθρωτική ε, ε, πολιτική που μας προτείνεται στη συνθήκη Μερκοζή, σας ζητώ να σταθείτε σε αυτή την έννοια που άρχισαμε να τη συζητάμε χτες. Διαρθρωτικό έλλειμμα. Αυτή η έννοια είναι αντικείμενο μεγάλη συζήτηση ανάμεσα στους οικονομολόγους. Συνδέεται με ένα δυνητικό ποσοστό ανάπτυξης οικονομίας, συμβατό με ένα σταθερό πληθωρισμό. Δηλαδή, να εξασφαλίσουμε, λένε οι πιο ορθόδοξοι οικονομολόγοι, ότι η οικονομία δεν έχει λόγο να κινηθεί από τη στιγμή που η δομή του κόστου παραγωγής παραμένει ίδια. Και σε αυτές τις περιπτώσεις μπορούμε να ανεχθούμε σε περίπτωση συγκυριακή διακύμανση ένα τρέχον έλλειμμα κάπω πιο σημαντικό μέσα σε ένα συγκεκριμένο όριο, π.χ. 3% του ΑΕΠ. Το μεγάλο πρόβλημα όμω είναι ότι αυτή η έννοια του διορθωτικού ελλείμματο δεν είναι στέρεη, δεν είναι συμπαγή, ούτε σκόπεμοι από εμπειρική άποψη, Η ίδια η Κομισιόν αναγνωρίζει ότι αυτό που ονομάζουμε διαρθρωτικό έλλειμμα εξελίσσεται βραχυπρόθεσμα. Αυτό αμφισβητεί την σκοπιμότητά του. Και άρα, εφόσον αυτό το διαρθρωτικό έλλειμμα εξελίσσεται κατά τη διάρκεια της κρίση, όπου το κόστος παραγωγής, το δομή του κόστος παραγωγής δεν έχει αλλάξει, αυτό ε, σημαίνει ότι εξαρτάται από το τρέχον έλλειμμα που το ίδιο εξαρτάται από την ανάπτυξη και άρα την πραγματική ζήτηση, η οποία έχει επιδεινωθεί αυτή τη στιγμή, δηλαδή κατανάλωση και επενδύσεις των επιχειρήσεων. Τι κάνει λοιπόν η συνθήκη Μερκοζή, μας απαγορεύει να δράσουμε για αυτές τις δαπάνες θεσμοθετώντας πολιτικές ε, δημοσιονομικής εξηγένσης. Το γεγονός λοιπόν ότι η αυτή, το διαστητικό αυτό έλλειμμα παραμένει πολύ εύθραυστο και οι πολιτικές εξυγίανσεις ε, διέπονται από μια ιδεολογία που είναι και η ίδια αμφισβητήσιμη, δεν μπορούμε παρά να στηρίξουμε αυτούς που πιστεύουν ότι πρέπει να διαπραγματευτούμε εκ νέου τη συνθήκη Μερκοζή, εάν θέλουμε ο μηχανισμός αλληλεγγύης να επιτρέψει στα κράτη-μέλη να ξαναπεράσουν σε ανάπτυξη. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Πίντο από την Πορτογαλία. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Ήθελα να, να, να πω ότι η ιδέα αυτή της καθιέρωσης ενός ορίου ελλείμματος συζητήθηκε στη χώρα μου όπου το 2010 ο, καν, ο κανόνας του προϋπολογισμού ήδη είχε εγκριθεί για να ξεκινήσει να ισχύει το 2015 ένα όριο αντίστοιχο με αυτό που προβλέπεται στη Δημοσιονομική Συμφωνία, δηλαδή για το μεσοπρόθεσμο στόχο. Ελπίζουμε ότι θα υπάρξει συνένεση για να μπει στο Σύνταγμα, εν πάση περιπτώσει να έχουμε την απαραίτητη πλειοψηφία για να αλλάξουμε αυτόν τον ε, νόμο περί προϋπολογισμού. Όπως ξέρετε η χώρα μου είναι υπό ένα πρόγραμμα προσαρμογής και έχει τηρήσει ε, εξ ολοκλήρου τους στόχους. Με μεγάλη συνένεση μάλιστα, πάνω από το 80% των δυνάμεων που αντιπροσωπεύονται στο Κοινοβούλιο και με μεγάλη κοινωνική συνένεση επίσης. Ωστόσο, η εφαρμογή κάποιων, αυτών, κάποιων μέτρων οδήγησε σε ύφεση πρέπει να σας πω ότι το οικονομικό πλαίσιο είναι λιγότερο ευνοϊκό από τότε που υπογράφηκε αυτή η ε, συμφωνία, το memorandum. Γι' αυτό και ήθελα να πω ότι η εφαρμογή αυτής της ε, δημοσιονομικής ε, συνθήκης θα τονίσει ακόμα περισσότερο τα αίτια Μία επίτευξη, μία υλοποίηση κάποιων μέτρων. Από τη στιγμή που επιθυνώνεται ολόκληρο το πλαίσιο, ολόκληρο το περιβάλλον το οικονομικό, υπάρχει γενική ύφεση στην Ένωση, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Κατά τη γνώμη μου αυτή η συνθήκη ενισχύει μια από τις πτυχές ε, την ε, δημοσιονομική πειθαρχία. Δεν γίνεται να συμπεριληφθούν εκεί όλοι οι εταίροι, δεν περιλαμβάνεται δηλαδή η κοινωνική συμφωνία. Υπάρχουν πτυχές που πιστεύω ότι τεχνικά θα είναι πιο προβληματικές από ας πούμε αυτή η έννοια του διαρθρωτικού ελλείμματος. Πολλές φορές διορθώνεται στο τέλος της ε, οικονομικής χρήση. Είναι ένα είδος κινούμενου στόχου. Θα μπορούσαμε όμως να έχουμε ξεχωριστά ταμεία ανάλογα με κράτος να, ώστε να μπορεί η Κομισιόν να επιβλέπει το τι συμβαίνει σε κάθε κράτος. Αυτή η συνθήκη προϋποθέτει με ένα σύνολο μέτρων και επίσης μιας, ε, μια υπόσχεση που υπονοείται όσον αφορά την ανάπτυξη, την εξάλληψη των ε, ε, ανισορροπιών εντός της Ένωσης και ελπίζουμε ότι αυτό θα αντικατοπιστεί και στα διαστατικά ταμεία. Δεν έχει νόημα να μιλάμε για δημοσιονομική πειθαρχία εάν δεν συνοδεύεται από πολιτικές υπέρ της ανάπτυξης. Διαφορετικά θα μείνει νεκρό γράμμα αυτή η συνθήκη. Ευχαριστώ. Ακόμη μια κάρτα. Όλε Σμιτ, Ευρωβουλευτής. Όλε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Είμαι Σουηδός φιλελεύθερος. Η Σουηδία, ως γνωρίζετε, είναι εκτός Ευρωζώνης. Θα ήθελα να τονίσω, να τονίσω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι βρισκόμαστε σήμερα εδώ και συζητούμε τα θέματα αυτά. Το επικίνδυνο σήμερα στην Ευρώπη είναι ότι χωρίζουμε πια την Ευρώπη σε διαφορετικές κατηγορίες. Αυτό είναι πραγματικά επικίνδυνο και δεν θα πρέπει να το επαναλάβουμε. Η ιστορία μας έχει αποδείξει ότι αυτό μπορεί να έχει δραματικές συνέπειες για την Ευρώπη. Γι' αυτό θεωρώ ότι συναντήσεις όπως η σημερινή είναι πολύ χρήσιμες. Και έχουν βελτιωθεί κιόλα. Οι πρώτε ίσω να μην ήταν τόσο ουσιώδει, αλλά σήμερα προχωρούμε πια σε ουσιαστικέ συζητήσει. Εγώ παρακολούθησα και χθε και ήθελα να, να και σήμερα και νόμιζα ότι θα είναι μόνο για την Ευρωζώνη. Αντιθέτω όμω, δεν αφορά μόνο τις χώρες τη Ευρωζώνης, αφορά όλους μας. Διότι όλοι είμαστε αλληλοσυνδεδεμένοι και αλληλοεξαρτώμεθα. Και βέβαια πρέπει να σεβόμαστε τις αποφάσεις των εθνικών βουλών και των πολιτών που εκπροσωπούν. Αλλά πρέπει να έχουμε υπόψη μα. Εμείς κάναμε δημοψήφισμα και Έχουμε δημοψήφισμα και η Δανία επίση και έχουμε αποκλήσει. Και η Μεγάλη Βρετανία είναι εκτό. Οι υπόλοιπε θέλουν να ενταχθούν στην Ευρωζώνη όμω. Εκτός από εμά του τρει. οι άλλε χώρε θέλουν να ενταχθούν στην Ευρωζώνη. Και όσε δεν είναι ακόμη μέσα. Και πρέπει να τα συζητήσουμε τα πράγματα αυτά. Και όλοι θα έπρεπε να αναγνωρίσουμε ότι οφείλουμε να είμαστε εδώ και να συζητούμε. Η Πρόεδρος, δεν έχω άλλους που να έχουν ζητήσει το λόγο. Βεβαίως τέθηκαν ερωτήσεις προς τους εισηγητές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχουμε χρόνο για να μπορέσουν να μας απαντήσουν. Θα τους πάρω λοιπόν αντίστροφα από ό,τι μίλησαν στην αρχή και πρώτα θα δώσω επομένως το λόγο στον Έλμαρ Μπρόκ. Ευχαριστώ. <clears throat> Κυρία Πρόεδρε. Λίγες σύντομες παρατηρήσεις. Πρώτα, χαίρομαι που δήλωσαν συμμετοχή 27 χώρες. Άρα η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν διαιρείται. Με εξαίρεση την προσωρινή απομόνωση δύο χωρών μελών. Και θα πρέπει να φροντίσουμε, να εξετάζουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση ως ενότητα, γνωρίζοντας βέβαια ότι με την εξαίρεση της Μεγάλης Βρετανίας και της Δανίας όλες οι υπόλοιπες χώρες έχουν δεσμευτεί να ενταχθούν στο ευρώ. Για να διατηρηθεί η ενότητα λοιπόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σημαντικό να δημιουργηθούν και βελτιωμένες συνθήκες συνεργασίας μεταξύ Εθνικών Κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού. Είναι σαφές και σύμφωνα με τη συνθήκη της Λισαβόνας αλλά και σύμφωνα με τα εθνικά συντάγματα ότι ο ρόλος είναι σαφέ μάλλον ποιο είναι ο ρόλο τη κάθε Εθνική Βουλή και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και για να ανταποκριθούν καλύτερα στα καθήκοντα αυτά, σωστό είναι να συζητούν, να συνομιλούν συχνά. Για να ελέγχουν τι οικίε δημόσιε διοικήσει. Απαντώ τώρα στην κυρία Μπερέση πρώτα. βρισκόμαστε ενώπιον του διλήμματος θα θεσπίσουμε και θα τηρήσουμε κανόνες ή θα αφήσουμε τις αγορές να κρίνουν το μέλλον των χωρών μας. Προτιμώ τους κανόνες. Και εσείς, Μπιλ, η Μεγάλη Βρετανία επέλεξε το opt-out για το ευρώ. Θα μπορούσε να συμμετάσχει στο Fiscal Compact χωρίς αυτό να έχει απόλυτος καμία συνέπεια για αυτήν. Έχει ένα απόλυτο ολοκληρωτικό opt-out. Όταν συζητούμε εμείς 25 τώρα και για ανταγωνιστικότητα, εκεί θα πρέπει να αποφασίσει η Μεγάλη Βρετανία. Τι θα κάνει, διότι θα βρίσκεται εκτός ορισμένων οργάνων. Και βέβαια, χώρες μέλη μπορούν από άποψη διεθνούς δικαίου να συνάπτουν συμφωνίες. Πρόκειται για συμφωνία διεθνούς δικαίου. Δεν μπορεί κανείς να το εμποδίσει αυτό. Και αυτά όλα δεσμεύουν οικειοθελώς τα συμβαλόμενα μέρη. Τα συμβαλόμενα μέρη αποφασίζουν και επιβάλλουν στους εαυτούς τους κανόνες. Και αυτά θα κυρωθούν από τις Εθνικές Βουλές ή και με δημοψηφίσματα, όπου αυτό προβλέπεται. Δεν βλέπω λοιπόν που εδώ τίθεται σε κίνδυνο η εθνική δημοκρατία, διότι πρόκειται για ελεύθερες δημοκρατικές αποφάσεις και θα επισημάνω ένα πράγμα. Όσο παραπλανητικά και να ακούγονται τα λόγια σου. Ναι, η κυρία Μέρκελ όντως θέλει να ελαχιστοποιήσει τους κινδύνους. Διότι αναλαμβάνει κινδύνους η κυρία Μέρκελ με τις υποσχέσεις, με τις εγγυήσεις που έχει αναλάβει η χώρα της απέναντι σε άλλες. Είμαστε αλληλέγγυοι μεταξύ μα. Οι 17 χώρες τη ζώνη ευρώ και άλλε που συμμετέχουν στην προσπάθεια. Και κάποιο ο οποίο δεν είναι αλληλέγγυο, δεν θα πρέπει να έρχεται να μέμφεται τους άλλους ότι θέλουν να μειώσουν, να ελαχιστοποιήσουν τους κινδύνους όταν δείχνουν αλληλεγγύη. Αυτός που δεν δείχνει καμία αλληλεγγύη βεβαίω, δεν αναλαμβάνει και απολύτω κανένα κίνδυνο. Παρόλο που εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι οικονομικά λάθο εάν πέσει η ζώνη ευρώ και το ευρώ, τότε και η Μεγάλη Βρετανία λόγω του χρέους της, λόγω της κατάστασης του τραπεζικού της συστήματος, θα βρεθεί πολύ γρηγορότερα σε δραματικές καταστάσεις, πολύ γρηγορότερα από ό,τι ορισμένες χώρες της ζώνης ευρώ. Όλα τα γεγονότα αυτό δείχνουν. Αυτή την αλήθεια ας μην την παραβλέπετε. Και στο μέλλον, με την παρούσα συνθήκη που συζητούμε τώρα, αυτό το επιβάλαμε ώστε να μπορεί να συμμετέχει και η, Ευρω... και η Μεγάλη Βρετανία να αντικατασταθούν οι κανόνες από κανόνες κοινοτικού, ώστε να μπορεί να συμμετέχει και η Μεγάλη Βρετανία και νομοθετικά. Εδώ νομίζω λοιπόν γενοδορία δείχνουν οι 25 και όχι τόσο η Μεγάλη Βρετανία. Αλλά το κάνουμε αυτό εμείς οι 25 δηλαδή, διότι θέλουμε να διατηρηθεί η ενότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν θέλουμε διαίρεση. Κυρώσεις. Οι κυρώσεις εφαρμόζονται σύμφωνα με το six και σύμφωνα με τις διατάξεις του Συμφώνου Σταθερότητας και Αναπτύξεως. Και μόνο η αντίστροφη πλειοψηφία του, ε, της συνθήκης και αυτή μπορεί να αποφασίσει την παρέμβαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Και αυτό βεβαίως εθελοντικά έχουν αναλάβει να δεσμευτούν οι χώρες μέλη. Και οι Σκοτσέζοι στο κάτω της γραφής δεν αντιτίθενται στις αποφάσεις του Λονδίνου. Έτσι λοιπόν και οι χώρες μέλη αποφασίζουν και επιβάλλουν κανόνες στους εαυτούς τους οι ερωτήσεις που έχουν σχέση με τους κανόνες τώρα. Είναι σαφές ότι η κρίση αυτή θα ξεπεραστεί μόνο εάν υπάρξει ανάπτυξη. Αλλά για να, ε, ε, για να έχουμε αξιοπιστία πρέπει να αποφασίσουμε δύο πράγματα. Πρώτον, να τηρήσουμε τους κανόνες, κάτι που δεν κάναμε την τελευταία δεκαετία και γι' αυτό φτάσαμε στα υψηλά χρέη και γι' αυτό φτάσαμε σε αυτή την εξάρτηση από τις διεθνείς αγορές αγορές που είναι ανυπόφορες, Το ΑΕΠ όλων των χωρών του πλανήτη είναι 55 τρισεκατομμύρια ευρώ. Στις αγορές όμως, χωρίς καμία απολύτως σχέση με την πραγματικότητα, κυκλοφορούν 500 τρισεκατομμύρια ευρώ στις αγορές. Προσέξτε τώρα. Χρειαζόμαστε στην Ευρώπη κανόνες για να μην στο τέλος της γραφής καταστρέψουν αυτά τα 503 εκατομμύρια ευρώ όλες τις χώρες του κόσμου. Αυτά οδήγησαν στην κρίση. Και αυτά ζητεί να μην ρυθμίσουμε η Μεγάλη Βρετανία. Όποιο είδε τι αποφάσει τώρα για το πακέτο για την Ελλάδα θα είδε ότι οι μισές τουλάχιστον αποφάσεις είναι διαρθρωτικές αλλαγέ για να οδηγήσουν σε μεγαλύτερη παραγωγικότητα. Είναι απαραίτητε οι διαρθρωτικές αλλαγέ, διότι μόνο τότε θα υπάρξουν επενδύσεις. Μόνο, επενδύσεις μόνο θα γίνουν εφόσον υπάρχει δυνατότητα αύξηση ανταγωνιστικότητα. Η δεμή πρόκειται για πίθο των Δαναίδων. Βαρέλι χωρί πάτο και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν σημαίνει μόνο δημοσιονομική πειθαρχία και σταθερότητα τιμών. Αλλά αυτή, αυτό είναι το πρώτο στο καθήκον της. Τα 500 δισεκατομμύρια με 1% θα μας δώσουν σταθερότητα τιμών για τα επόμενα χρόνια. Του Δεκεμβρίου δηλαδή. Η χώρα μου επιμένει στην ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Γι' αυτό μπορούμε να πούμε τώρα ότι υπάρχει και η άλλη πλευρά, δηλαδή να γίνει προσπάθεια για δημοσιονομική πειθαρχία. Αυτά πρέπει να κινούνται χέρι με χέρι. Δεν είναι δυνατό να ξεχνούμε ότι υπάρχει, υπάρχει αυτό το τρίπτυχο δημοσιονομική πειθαρχία, διαφθορτικές αλλαγές, ανάπτυξη. Τα αντίθετα όμως αυτά που λένε οι Βρετανοί και οι Αμερικανοί, δηλαδή θα λύσουμε το πρόβλημα τυπώνοντας, εκδίδοντας περισσότερο χρήμα, αυτό είναι λάθος. Δημοσιονομική πειθαρχία, διαρθρωτικές αλλαγές και μετά αυτές θα οδηγήσουν σε ανάπτυξη και σε λίγα χρόνια θα είμαστε ανταγωνιστικότεροι από ότι ορισμένες άλλες περιοχές του κόσμου οι οποίες δεν ασκούν τις πολιτικές αυτές. Δεν θα επανέλθω στο παράδειγμα των 55 τρισεκατομμυρίων και των 500 τρισεκατομμυρίων, όπως είπα, του πλανήτη. Οι Ευρωπαίοι προχωρούν σε έναν αγώνα εν μέσω δραματικών εξελίξεων σε ολόκληρο τον κόσμο. Αν δείτε τους Κινέζους, αν δείτε τους Αμερικανούς προχωρούν σε μια δημιουργία μιας ε, ζώνης ελεύθερων συναλλαγών του ειρηνικού, ενώ εμείς οι Ευρωπαίοι είμαστε στερημένοι από πρώτες ύλες. Αν οι Ευρωπαίοι δεν θέλουμε κάποια στιγμή να διαγραφούμε από τον χάρτη, πρέπει να αγωνιστούμε. Και γι' αυτό πρέπει να τα πει κανείς αυτά καθαρά και στους πολίτες και στις προεκλογικές εκστρατείες και όχι να τους λένε πράγματα που είπαμε στις δεκαετίες του 70, του 80, του 90 ακόμα μόνο για να τους χαϊδεύουμε τα αυτιά διότι πιστεύω ότι οι πολίτες θα αποδειχθούν στο τέλος ευφιέστεροι από πολλούς λαϊκιστές Ρομπέρτο. Καλώς ο Ρομπέρτο παρακαλώ Ευχαριστώ. Εγώ θα προσπαθήσω να απαντήσω σε κάποια ερωτήματα. Πρώτος, ομπιλικάς και άλλοι. Αμφιβολίες περί νομιμότητας. Θα προτιμούσα να είχα συγκεκριμένα παραδείγματα, γιατί αμφιβολίες περί νομιμότητας είναι πολύ γενικευμένο Σόρος. Εγώ επαναλαμβάνω αυτό που προσπάθησα να σας πω στην αρχή. Όσον αφορά την συνταγματικότητα του Golden Rule, του χρυσού κανόνα, αυτή δεν είναι υποχρεωτική. Λέει κατά προτίμηση, preferably, Ε, είναι δύσκολο λοιπόν να αναγκαστεί κάποια χώρα να κάνει δημοψήφισμα γι' αυτό. Τώρα, ο ρόλο των θεσμών τη Ένωση. Ακριβώ επειδή η συνθήκη στην οριστική τη μορφή αντικατοπτρίζει τις υποχρεώσεις όπως ορίζονται από την νομοθεσία της Ένωσης, αυτό δεν δίνει καινούριε αρμοδιότητες στα θεσμικά όργανα ή αντιφατικές ε, ε, αρμοδιότητες σε σχέση με αυτούς που ήδη έχουν. Η Κομισιόν ήδη πρέπει να ορίζει τους μεσοπρόθεσμους στόχους και πρέπει να ορίζει την έννοια του διαρθωτικού ελλείμματος που είναι σωστό να πούμε ότι δεν υπάρχει στη φύση το διαρθωτικό έλλειμμα. Είναι αυτό που ορίζει κανείς και εξαρτάται από αυτόν που το ορίζει. Αλλά η Κομισιόν είναι αυτή που επί τη βάση της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας ε, το ορίζει. Άρα λοιπόν δεν δίνεται νέα αρμοδιότητα στη Κομισιόν σε σχέση με αυτές που ήδη έχει. Επιπλέον η συνθήκη και αυτό επίσης χάρη στην ε, δέσμευση του Ευρωκοινοβουλίου και της Κομισιόν λέει ότι αυτό θα πρέπει να εφαρμόζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο με τις διαδικασίες της κοινοτικής νομοθεσίας. Όταν λοιπόν θα υπάρξουν συγκεκριμένες αρμοδιότητες που θα πρέπει να ανατεθούν στα θεσμικά όργανα, αυτό θα γίνει μέσω της εφαρμογής μιας κοινοτική νομοθεσίας. Δηλαδή αυτό το στοιχείο της ε, ε, μη νομιμότητας δεν υπάρχει. Ακριβώς διότι αυτή τη στιγμή η συνθήκη αντικατοπτρίζει την, την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία που θα ήθελα να προσθέσω προβλέπει και την περίπτωση ειδικών διατάξεων για την Ευρωζώνη. Γιατί το άρθρο 136 προβλέπει ακριβώς την ύπαρξη συγκεκριμένη νομοθεσία ή διατάξεων για την Ευρωζώνη. Α, λοιπόν, αυτό το θέμα το οποίο ε, αναφέρεται για παρανομία δεν ναι, ναι, είναι αβάσιμο από νομικής άποψης. Υπάρχει βέβαια ένα θέμα πιο λεπτό που αφορά το άρθρο 8. Το ρόλο του δικαστηρίου. Και πιο συγκεκριμένα το 8.2. Έχω εδώ κάποιες αμφιβολίες, αλλά εδώ το δικαστήριο θα πρέπει να αποφασίσει αν θα εφαρμόσει το άρθρο 8.2, δηλαδή αν θεωρεί πως είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί η νομική βάση του άρθρου 260 στην επαλήθευση της εφαρμογής μιας απόφασης του επί τη βάση του άρθρου 263, πράγμα το οποίο λέγεται, αναφέρεται στο άρθρο 8.1. Αυτό δεν μπορεί όμως να το αμφισβητήσει κανείς εξαρτάται από το δικαστήριο αν θα χρησιμοποιήσει ή όχι αυτή την παράγραφο, αυτό το εδάφιο ή όχι. Τώρα, για τις κυρώσεις, έχουμε σύμφωνα με τη συνθήκη τρεις δυνατότητες. Η μία ορίζεται από το άρθρο 8, Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, που αφορά την εφαρμογή του άρθρου 3.2 Δηλαδή, το δικαστήριο πρέπει να αξιολογήσει αν τα κράτη θα τοποθετήσουν στο σύνταγμά τους ή σε ενισχυμένη νομοθεσία την, το χρυσό κανόνα και αν θα δημιουργήσουν έναν διορθωτικό μηχανισμό. Επ' αυτού μόνο δίνει ένα ρόλο στο δικαστήριο, ε, ένα ρόλο διαιτησίας επί τη βάση του άρθρου 263 της συνθήκης. Αυτοί οι μηχανισμοί λοιπόν θα εξετάζονται και θα ελέγχονται από τις εθνικές αρχές. Εδώ λοιπόν το δικαστήριο, το ευρωπαϊκό δεν έχει σχέση. Ε, θα πρόκειται για τους ε, μηχανισμούς του, κράτους, του κάθε κράτους μέλους για την, που ελέγχουν την εφαρμογή των ε, νομοθεσιών του. Έπειτα υπάρχει ένα τρίτο επίπεδο κυρώσεων σε σχέση με την εφαρμογή του six δηλαδή, το ίδιο το περιεχόμενο το οποίο θα εποπτεύουν οι εθνικές αρχές ε, εάν δεν γίνουν σεβαστές αυτές οι παράμετροι μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο κυρώσεων επί τη βάση ενός κοινοτικού κανονισμού. Αλλά σε αυτό η συνθήκη δεν κάνει κάτι νέο. Υπήρχε ήδη, προβλεπόταν ήδη από το εξαπλό πακέτο και οι κυρώσεις του δεν προσθέτει ούτε κόμμα η νέα συνθήκη. Ένα μηχανισμός πολύ πιο αποτελεσματικός από την ίδια τη συνθήκη που ορίστηκε από έναν κοινοτικό κανονισμό. Συλλογικά λοιπόν έχουμε μια δομή με τρία διαφορετικά επίπεδα ε, μηχανισμών ελέγχου και επιβολής κυρώσεων. Τώρα, το θέμα των ανεξάρτητων ε, μηχανισμών. Σύμφωνα με το άρθρο 3, η Κομισιόν ορίζει αρχές, αλλά μετά οι χώρες, η κάστοτε χώρα, ορίζει αυτόν τον ε, ανεξάρτητο μηχανισμό ελέγχου. Είναι λοιπόν απόλυτη αρμοδιότητα εθνική, εθνικού επίπεδου. Όλα αυτά ενισχύουν την πτυχή της δημοσιονομικής, ε, δημοσιονομικής πειθαρχίας, που βεβαίως είναι μια προϋπόθεση για να διαχειριστεί κανείς ε, ένα ενιαίο νόμισμα, αλλά όχι επαρκής ε, προϋπόθεση. Και ούτε είναι το κύριο μέσο αυτό. Συμφωνώ με τους συναδέλφους που μίλησε. Υπάρχουν άλλα προβλήματα σημαντικά και το ένα αναφέρθηκε από τον Πορτογάλο, νομίζω, συνάδελφο, αυτό των μακροοικονομικών ανισορροπιών. Εκεί βεβαίω έχουμε πρόβλημα, γιατί αν στην έκθεση τη Επιτροπής λέει ότι όσον αφορά τις χώρες που έχουν έλλειμμα, 4% λέει είναι η παράμετρο. Όσον αφορά τις χώρες Σέρπλας είναι 6%. Δυστυχώ η Γερμανία είναι 5,9%. Οπότε πρέπει να γίνει πολλή δουλειά όσον αφορά την πτυχή της πραγματικής εφαρμογής ε, ε, του κανονισμού Φερέιρα όσον αφορά τις μακρονομικές ανισορροπίες. Αν δεν αντιμετωπιστεί αυτό το θέμα, δεν αντιμετωπίζεται το πρόβλημα της κρίσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν υπάρχει αμφιβολία περί τούτου, όπως δεν υπάρχει αμφιβολία περί του αν έχουμε όσο γίνεται πιο αυστηρή η δημοσιονομική πειθαρχία σε εθνικό επίπεδο, χρειάζονται πόροι και μέσα για πολιτικές επενδύσεων και απασχόληση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εδώ έρχεται το θέμα των ομολόγων έργου, του ευρωπαϊκού προπολογισμού, των ίδιων πόρων του, του φόρου για τις ε, ε, χρηματοπιστωτικές συναλλαγές που αποκτούν καθοριστική σημασία. Γιατί φορτίγα έχουμε ένα οικοδόμα το οποίο δεν στέκει γιατί δεν έχει ισορροπία. Αυτό απασχολεί τα θεσμικά όργανα αλλά και τα εθνικά κοινοβούλια που κατά τη γνώμη μου έχουν τεράστιο ρόλο να παίξουν και ίσως ο ρόλος της προηγούμενης κατεύθυνσης ε, το δράση των κυβερνήσεων μέσα στα ευρωπαϊκά όργανα είναι σημαντικός. Δηλαδή δεν μπορεί να, μόνο να υπογράφουν κατόπιν εορτής. Τώρα είτε μας αρέσει είτε όχι, στην ουσία οι κυβερνήσεις είναι μέλη μιας από τα δύο σώματα, δηλαδή ένα είδος γερουσίας του ε, Συμβουλίου. Το θέμα λοιπόν της κατεύθυνσης που θα δοθεί για το τι θα κάνουν αυτές οι κυβερνήσεις εκεί πέρα μέσα είναι ε, ένα θέμα το οποίο δίνει τεράστια δύναμη στα εθνικά κοινοβούλια. Θα πρέπει αυτό να, το, να ερμηνευθεί ε, όπως δει και να αναλάβουν τα εθνικά κοινοβούλια αυτό το ρόλο. Αυτό είναι αποκλειστικά πολιτικό ζήτημα. Δεν είναι θέμα αυτής της ε, συνεδρίας, οπότε σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ε, ευχαριστώ πολύ. Νομίζω, αν θυμάμαι καλά, ότι δύο είναι τα ζητήματα που δεν έχουμε εξετάσει, εκτός και αν κάνω λάθος. Τις ερωτήσεις του κυρίου Ντόναχιου Πρώτον, το θέμα της μακροοικονομικής ανισορροπίας που αρχικά ήταν στο εξαπλό πακέτο μέτρων και ότι χρειάζεται περισσότερη εξέταση όλων αυτών και όντως το Κοινοβούλιο προσπάθησε να σπρώξει τα πράγματα, να τα πιέσει προς αυτή την κατεύθυνση όταν γινόταν διαπραγμάτευση για τη δέσμη έξι μέτρων. Καταφέραμε ε, το συνολικό πακέτο να κλείσει ε, με αρκετά συμμετρικό τρόπο παρόλο που δεν καταλήξαμε για το πίνακα βαθμολόγησης και τους δείκτες όμως έχει προβλεφτεί αυτή η διαδικασία ε, κοινοβουλευτικής εξέτασης και ελπίζουμε ότι έτσι θα ε, αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που επισημάνατε εσείς. Τώρα, το άλλο ερώτημα για τις εξωτερικές επιπτώσεις, για τις αποφάσεις που ε, λαμβάνονται σε, ένα χώρο και ε, σε μια χώρα και αν έχουν εξωτερικές επιπτώσεις σε άλλες χώρες, νομίζω ότι υπάρχει μια ρήτρα διαφυγής εκεί. Μπορείτε να το σχολιάσετε. Ναι, είναι μια πολύ σημαντική ερώτηση, ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο αυτό. Το εξωτερικό αποτέλεσμα καθιστά ε, σαφές πόσο μεγάλη σημασία έχει να πετύχουμε εμείς. Πόσο μεγάλη σημασία έχει το γεγονός ότι το άρθρο 3 ευθυγραμμίζεται πλέον με τη νέα νομοθεσία. Αυτό ισχύει και για το άρθρο 3 και για το άρθρο 4 περί χρέους. Υπάρχει αυτή η ρήτρα η οποία θεσπίζει πιο αυστηρά στοιχεία σε επίπεδο ευρωπαϊκής νομοθεσίας και MTO έχουμε τη δυνατότητα στον ορισμό του MTO, του συγκεκριμένου στόχου αναχώρα, του ετήσιου διαρθρωτικού ελλείμματος και το καθεξής, εκεί μπορούμε να λάβουμε υπόψη μας και διαφορετικά στοιχεία, το περιραίον πλαίσιο, την αλληλεξάρτηση, την κρίση στη μία χώρα και στην άλλη ενδεχομένω. Όλα αυτά έχουν να κάνουν και με τον τρόπο με τον οποίο εκπληρώνει τα καθήκοντά της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σωστά ή λάθος. είναι η συνήθις διαδικασία ελέγχου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πώς θα ορίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το MTO, το διαρθρωτικό έλλειμμα και ποια μέτρα θα λάβει υπόψη της, ε, ποια στοιχεία θα λάβει υπόψη της, τα εξωτερικά στοιχεία σε σχέση με το κράτος. Όλα αυτά πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και μπορεί να γίνει αυτό. Το διαρθρωτικό έλλειμμα δεν είναι το έλλειμμα που προβλέπεται στη συνθήκη μέχρι 3% του ΑΕΠ. Το 3% του ΑΕΠ είναι, είναι ένας αριθμός, δεν είναι τίποτα άλλο. Το διαρθρωτικό έλλειμμα είναι ένα στοιχείο που εκπορεύεται, που είναι προϊόν, αν θέλετε, της ύπαρξης διαφόρων παραγόντων. Θεωρώ λοιπόν ότι υπάρχει χώρος για να ε, ε, λαμβάνονται υπόψη και τα εξωτερικά στοιχεία, οι εξωτερικές συνέπειες. Όλα αυτά βεβαίω θα υλοποιηθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εξού και προκύπτει ενδυνάμωση του ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Εθνικών Κοινοβουλίων, διότι τα κοινοβούλια ε, θα διαλεχθούν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε νέα νομοθεσία και είναι πολύ λεπτός ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πολύ σημαντικός. Κάθε μέρα διαβάζουμε π.χ. στις εφημερίδες ότι αποφασίστηκε ότι το Βέλγιο πρέπει να προβεί σε δημοσιονομική διόρθωση τέτοιου χι επίπεδου κτλ. Επομένως, δεν είναι μόνο αυτά αριθμοί, είναι και πολιτική ερμηνεία, πολιτική οικονομία, τρόπος ε, λήψης υπόψη διαφορετικών παραγόντων. Όλα αυτά είναι πολιτική και θα έπρεπε έτσι ακριβώς να είναι η ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση. Και εξού και να βαθμίζεται ο ρόλος των κοινοβουλίων. Και βεβαίως πρέπει να βελτιώσουμε ε, πολλά ε, τα επόμενα χρόνια. Ευχαριστώ. Η Σιλβή. Δύο λόγια για τις μακροοικονομικές ε, ανισορροπίες. Γιατί ο συνάδελφος ε, τόνισε κάτι το πολύ σημαντικό. Βρισκόμαστε στην αρχή μιας διαδικασίας η οποία είναι εντελώ καινούρια και σχεδόν επαναστατική θα έλεγα αναφορικά με το πνεύμα που μας διείπε όταν ε, συνάψαμε τη Συμφωνία Σταθερότητας. Έχουμε κανόνες που έχουν να κάνουν με τη διαχείριση δημοσίων ε, οικονομικών, έλλειμμα και χρέος και ε, υπάρχει επαρκές, αν θέλετε, θα μπορούσαμε να έχουμε επαρκή καθοδήγηση της οικονομίας. Όταν είχαμε ανισορροπίες στα ισοζύγια πληρεμών και ε, ε, ιδιωτικό έλλειμμα, ε, όλα αυτά τα είχαμε παραμελήσει. Με τα νέα αυτά εργαλεία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορέσει να λειτουργήσει. Έχουμε λοιπόν το εμβρυϊκό στάδιο μιας μακροοικονομικής πολιτικής η οποία πραγματικά μπορεί να γεννηθεί και να γίνει κοινή κοινοτική πολιτική. Και ε, υπάρχουν αυτές οι εξωτερικές ε, διαστάσεις. Ε, σε σχέση με αυτό που είπε και ο Φιλανδός συνάδελφος χθε για τα ευρωομόλογα, θέμα για το οποίο εγώ ήμουν η συνεισηγήτρια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και είχα τη στήριξη όλων των συναδέλφων βεβαίω. Κάτι που με εκπλήσει με αυτή την κρίση είναι το γεγονός ότι έχουμε μια φοβερή εσωστρέφεια. Προσπαθούμε να βρούμε φάρμακα και θεραπείες μέσα σε ένα πλαίσιο σκέψης αμυγός ευρωκεντρικό θέλουμε το αντίστοιχο του αμερικανικού ομολόγου ούτως ώστε να διασφαλίσουμε τη θέση του ευρώ ως διεθνούς νομίσματος ε, συναλλογών. Δεν, βεβαίως, ε, δεν θέλουμε τα ευρωομόλογα για να, να ε, προκύψει μετά το θέμα του ηθικού κινδύνου ε, δεν δουλεύουμε με αυτό το πνεύμα. Μιλούμε για την εξωτερική διάσταση των λύσεων. Πρέπει να φέρουμε λύσεις που να, ε, έχουν εξωτερικές διαστάσεις, ε, ούτω ώστε το ευρώ να παγιωθεί ως νόμισμα διεθνών συναλλαγών. Ευχαριστώ. Η Πρόεδρος. Κύριε Κάσο, Γνωρίζω ότι θέλατε ε, να αναφερθεί ε, μία δημοσίευση, μία έρευνα που έχει γίνει και μία μελέτη για την νομιμότητα της δημοσιονομικής αυτής συμφωνίας. Είναι γνωστό αυτό, είναι διαθέσιμη στη διαδικτυακή τοποθεσία της Βουλής των Κοινοτήτων του Ηνωμένου Βασιλείου, επομένως δεν χρειάζεται να το επαναλάβουμε εδώ ο κύριος Κάσ. Είναι θέμα ευρωπαϊκού δικαίου, όχι ε, δικαίου Ηνωμένου Βασιλείου. Ναι, λέει η Πρόεδρος, το, το καταλαβαίνω, είναι ένα πολύ ενδιαφέρον έγγραφο που αναλύει ε, τις πτυχές του ευρωπαϊκού δικαίου και όχι του δικαίου του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά υπάρχει αυτή η μελέτη διαθέσιμη στις, ε, στη διαδικτυακή τοποθεσία. Σας ευχαριστώ λοιπόν όλους ε, όσοι έχετε δώσει συμμετάσχει σε αυτή τη συζήτηση. Η επόμενη συνεδρία θα ξεκινήσει στις 11. Έχουμε 3-4 λεπτά διάρκεια διάλειμμα, ε, αλλά παρακαλώ να μην απομακρυνθείτε γιατί θα ξεκινήσουμε στις 11 ακριβώς για να μην καθυστερήσουμε. Ευχαριστώ. Chers collègues, je vous propose euh, Αγαπητοί συνάδελφοι, σας προτείνω να καθίσετε. Θα ξεκινήσουμε τη δεύτερη συνεδρία ανταλλαγής απόψεων με την κυρία Μάργκριτ Τεστάγκερ, Υπουργό της Δανίας, Υπουργό Οικονομικών της Δανίας, η οποία θα μας μιλήσει για τις εργασίες του ΕΚΟΦΗΝ και ε, τη σύνδεση με την νεαρινή Σύνοδο Κορυφής αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων. Θα ακούσουμε και τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον Επίτροπο κύριο Όλι Ρεν, αρμόδιο για δημοσιονομικά θέματα και ευρώ, και θα ακούσουμε και τον Επίτροπο Άντορ ε, με το υπεύθυνο του χαρτοφυλακίου για την απασχόληση. Να σας καλωσορίσω όλους. Βρίσκεστε ενώπιον αντιπροσωπιών από την πλειονότητα των Εθνικών Κοινοβουλίων των 27 χωρών μελών, των 24 μάλλον 25 χωρών μελών και έχουμε και μέλη τριών Επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εδώ στην αίθουσα. Από χθε διεξάγουμε διάφορες συζητήσεις ως προς την ετήσια μελέτη ε, ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ε, ε, συζητούμε επίσης τα θέματα της Δημοσιονομικής Συμφωνίας. Εάν δεν διαφωνείτε, να δώσω πρώτο το λόγο στους συναδέλφους μου και να πούμε και δύο λόγια για τις ειδικέ ε, συνεδριάσεις που οργανώσαμε εμείς χθες. Πρώτον, ε, το λόγο έχει ο κύριος Αλά Λαμασούχ, ε, πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου του Προπολογισμού. Έχετε το λόγο κύριε Λαμασούχ, για πέντε λεπτά το ανώτατο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί Επίτροποι, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα, εν συντομία, να πω ότι αυτές τις δύο ημέρες, οι οποίες δε βεβαίως δεν έχουν ολοκληρωθεί, είχαμε ε, πολύ επικοδομητικές συναντήσεις και ένα πρώτο συμπέρασμα το οποίο μπορούμε να εξάγουμε είναι η ανάγκη όχι απλής ανανέωσης ε, και επανάληψης αυτού του εγχειρήματο, αλλά η ανάγκη θεσμοθέτησής του. Ε, και νομίζω ότι η Περβάνς Μπερές θα επανέλθει στο θέμα αυτό εντός ολίγου. Δηλαδή θα πρέπει να θεσπιστεί ως ε, τρέχουσα κανονική διαδικασία αυτή η ανταλλαγή απόψεων με τα Εθνικά Κοινοβούλια, είτε βάσει του άρθρου 13, ε, είτε βάσει της υλοποίησης του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου κάθε ένα από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και κάθε ένα από τα μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων έχει ανάγκη να αποφασίζει επί της δημοσιονομικής πολιτικής λαμβάνοντας υπόψη ε, την ευρωπαϊκή διάσταση όλων αυτών των θεμάτων. Άρα είναι απαραίτητη ανάγκη να λαμβάνουν χώρα τέτοιες συζητήσεις όπου θα ε, θυγούν όλα τα θέματα που έχουν να κάνουν με την προσέγγιση του καθενός, την ανάγκη του καθενός, την άποψη του καθενός, ούτως ώστε η ευρωπαϊκή διάσταση να είναι παρούσα παντού ε, και να μπορεί ο κάθε βουλευτής στο κοινοβούλιο του στη συνέχεια να εξετάζει τα θέματα του εθνικού προπολογισμού υπό την ε, ε, οπτική γωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης επίσης. Πολλοί από εσάς χθες το απόγευμα αλλά και χθες το βράδυ στο δείπνο μας επιμείνατε στο γεγονός ότι ε, υπάρχει μια συγκεκριμένη δυσκολία στη συνεργασία μεταξύ ημών και ημών με ήττα και με ύψιλον αντιστοίχως διότι δεν έχουμε τις ίδιες βάσεις εκκίνησης ως προς τις οικονομικές προβλέψεις, για παράδειγμα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, προσφέρει προβλέψεις αδιαφυσβήτητες και έχουμε και την ετήσια μελέτη για την ανάπτυξη. Όμως, ε, ως προς την ονοματολογία των δημοσίων λογαριασμών, ως προς τους δημόσιους λογαριασμούς, ε, τους εθνικούς προϋπολογισμούς δεν ξεκινούμε από την ίδια βάση εκκίνησης και γι' αυτό δεν μπορούσαμε ε, ποτέ μέχρι σήμερα να προχωρήσουμε στην ενοποίηση των εθνικών προϋπολογισμών, των 27 εθνικών προϋπολογισμών, στους οποίους προστίθεται ο 28ος πλέον κοινοτικός προϋπολογισμός. Έχουμε λοιπόν ένα εργαλείο το οποίο θα μας επιτρέψει ε, μόλις χαράξουμε τη στρατηγική ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου έχουμε ένα εργαλείο να προχωρήσουμε προς τα εμπρός και στη συνέχεια το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Ιούνιο θα αποφασίσει για τη συνέχεια που θα δοθεί σε αυτή τη στρατηγική στρατηγική και τον ρόλο που θα η κάθε χώρα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, ως προς την επίτευξη αυτών των στόχων. Εν πάση περιπτώσει είναι ένα εργαλείο που μας ε, επιτρέπει να διαπιστώσουμε τι κάνει ο καθένας από εμάς για την Ευρώπη. Σε Γνωρίζουμε ήδη τα ε, θέματα δημοσίου ελλείμματος ή δημοσίου χρέους. Αυτά μπορούμε να τα λογιστικοποιήσουμε. Αλλά τι κάνει ο καθένας μας για την ανάπτυξη, για την κοινοτομία, για την ανταγωνιστικότητα, για τις ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια για τις νέες τεχνολογίες, για τις νέες επενδύσεις, για τα ευρωπαϊκά δίκτυα, αυτά μέχρι σήμερα δεν μπορούσαμε να τα ποσοτικοποιήσουμε ούτε να τα λογιστικοποιήσουμε και θα μπορούμε πλέον να ξέρουμε τι κάνει κάθε ένα από τα κράτη-μέλη ως προς αυτό. Πιστεύω λοιπόν ότι θα έχουμε καλύτερη οικονομική διακυβέρνηση και θα διασφαλίσουμε περισσότερο κοινοβουλευτικό, ε, κοινοβουλευτικό έλεγχο. Πράγματα για τα οποία είμαστε υπεύθυνοι. Ευχαριστώ πολύ. Η Πρόεδρος, να δώσω το λόγο στη συνάδελφο Σάρων Μπόου η υπεύθυνη ε, της πρώτης συνεδρίας, η οποία προείδρευσε κατά την πρώτη συνεδρία και θα μιλήσει η ίδια για το θέμα της δημοσιονομικής συμφωνίας. Τα κείμενα, τα κείμενα δηλαδή που εξετάζει αυτή τη στιγμή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχετε το λόγο για πέντε λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Χθες είχαμε μια πολύ επικοδομητική συζήτηση για τη δημοσιονομική πειθαρχία και την βιωσιμότητα των δημοσίων δαπανών. Αναγνωρίσαμε ότι είναι απαραίτητη ανάγκη να δημιουργηθεί ένα δημοκρατικό φόρουμ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ούτω ώστε σε αυτό το φόρουμ να εμπλέκονται και να συμμετέχουν όλοι όσοι ενδιαφέρονται να ε, κάνουν διάλογο για αυτά τα πολύ σημαντικά θέματα. Χρειαζόμαστε ε, δημοσιονομική εξυγίανση, η οποία όμως θα είναι φιλική προς την ανάπτυξη, ούτω ώστε να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη. Και δόθηκαν παραδείγματα από μέλη εθνικών κοινοβουλίων για το πώς πέτυχαν αυτή τη δημοσιονομική εξυγίαση στις χώρες τους στο πρόσφατο παρελθόν τους. Ακούσαμε και τους εισηγητές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι οποίοι αντάλλαξαν απόψεις με μέλη εθνικών κοινοβουλίων ε, ε, για διάφορα τεχνικά θέματα όπως είναι το ε, έλλειμμα στη μισή μονάδα σε σχέση με το ΑΕΠ. Από την τελευταία μια μισή μέρα κατέστησα σαφές ότι επικρατούν δύο εναλλακτικές απόψεις οι οποίες δεν είναι κατά ανάγκη ασύμβατες μεταξύ τους. Μπορούν να υλοποιηθούν ταυτόχρονα ενδεχομένως ξεχωριστά πρώτε μία μετά η μία μετά η άλλη. Αλλά εν πάση πτώση σίγουρα ε, χρειάζεται μια εξυγίανση δημοσιονομική για να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη, αλλά σίγουρα χρειάζεται και η βελτίωση της ανάπτυξης για να αυξηθούν τα φορολογικά έσοδα τα έσοδα των κρατών. Αυτές είναι οι παρατηρήσεις που επικράτησαν στη συζήτηση. Και επίσης στήξαμε και τις προκλήσεις που υψώνονται μπροστά μας ε, στο εγχείρημα ενισχυμένου συντονισμού των διαδικασιών ψήφισης του προϋπολογισμού στα διάφορα κράτη-μέλη. Ε, θίξαμε το θέμα της νομιμότητας, τα θέματα που έχουν να κάνουν με εθνικές ευαισθησίες μεταξύ άλλων. Η διαδικασία δηλαδή που ακολουθούμε εδώ είναι να προσφέρουμε ένα βήμα λόγου, μια νομιμότητα αν θέλετε σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεδομένης της ε, διασύνδεσης που μας χαρακτηρίζει Καμία χώρα ε, μέλος δεν μπορεί πλέον να λειτουργεί απομονωμένα και μεμονωμένα. Ένας από τους εισηγητές ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την δέσμη δύο μέτρων, τη διπλή δέσμη μέτρων, το Τούπακ, ε, εξέφρασε ανησυχίες για την αλληλουχία λήψης αποφάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θεωρεί ότι η δημόσια συζήτηση και η δημόσια διαβούλευση πρέπει να λαμβάνει χώρα πρώτα και στη συνέχεια να λαμβάνονται αποφάσεις και κλεισμένων των θυρών. Ενώ ο αντίστροφος δρόμος έχει ακολουθηθεί ε, μέχρι σήμερα. Εν γέννη συζητήσαμε τις θέσεις απασχόλησης, την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα, τη σημασία που έχει η ενιαία αγορά και τη σημασία που έχει η εφαρμογή όλων των μέτρων που θα οδηγήσουν στην τελειοποίηση της ενιαίας αγοράς. 20 ε, μέτρα λείπουν, δεν έχουν ακόμα εφαρμοστεί προκειμένου να ε, δημιουργηθεί μια πραγματικά ενιαία αγορά και αυτά τα μέτρα θα δρομολογηθούν βάσει της διαδικασίας fast track γιατί πράγματι είναι πήγον να εφαρμοστούν ε, το ταχύτερο δυνατό προκειμένου να εξυπηρετηθεί ο σκοπός της ανάπτυξης. Αυτά προς το παρόν σας ευχαριστώ πολύ. Η Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συνάδελφε. Τώρα θα έχουμε μία συζήτηση για την βιώσιμη ανάπτυξη της θέσης απασχόλησης και την ανταγωνιστικότητα σε δυσμενείς οικονομικές ε, συνθήκες. Ε, ο Επίτροπος Λεβαντόφσκι και ο Επίτροπος Χάν έχουν συμμετάσχει σε αυτή τη δουλειά. Τρεις εισηγητές από πλευράς Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η ε, της επικείμενης ε, κυπριακή Προεδρία του δεύτερου εξαμήνου του 12 και βεβαίως τρεις συναδέλφους ε, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η συζήτηση στράφηκε γύρω από τη γνωστή ιδέα. Θα πρέπει η Ευρώπη να επανασυμφιλειωθεί ε, με την ιδέα της ανάπτυξης, της οικονομικής μεγένθησης. Ο Επίτροπος Λεβαντόφσκι ε, ξεκίνησε τις εργασίες, ε, ξεκίνησε να μιλάει παρουσιάζοντας ε, ε, μια εικόνα πολύ ισχυρή ε, συναισθηματικά. Είχαμε την εικόνα της Ευρώπης και το βασικό μέρισμα το οποίο μπορούσαμε να απολαύσουμε όλες αυτές τις δεκαετίες ήταν το μέρισμα της ειρήνης. Αυτό πλέον έχει παγιωθεί και δεν αρκεί προκειμένου να είμαστε παρόντες στο διεθνές στερέωμα αυτό το οποίο θα κάνει τη διαφορά της Ευρώπης, αυτό το οποίο θα δημιουργήσει, θα συντάξει μια νέα αφήγηση ε, στην, ε, ε, στο, το διεθνές σκηνικό είναι οι λύσεις που μπορεί να προσφέρει η Ευρώπη για περισσότερη ανάπτυξη και για διαφυγή από την κρίση. Θα μπορούσαν λοιπόν τα διαρθρωτικά ταμεία του προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αξιοποιηθούν ως εργαλεία για την οικονομική μεγένθυνση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από πλευράς Ευρωπαϊκού ε, Κοινοβουλίου η κυρία Κόρνελίσεν ε, μίλησε για τέσσερις θεμελιώδεις αρχές. Πρώτον, η ανάγκη είτε σε εθνικό είτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο τη μία ή την άλλη στιγμή, κάποια στιγμή, εν πάση περιπτώσει, να συμπεριληφθεί η ευρωπαϊκή διάσταση στην λογική και ε, στον προβληματισμό των εγχώριων και των εθνικό, είτε πρόκειται για ε, χώρα ελληματική, είτε πρόκειται για χώρα πλεονασματική. Όταν, για παράδειγμα, γίνεται λόγο για επενδύσει σε μια συγκεκριμένη χώρα και αποφασίζει η κυβέρνηση, το κοινοβούλιο για τι επενδύσει, θα πρέπει πάντοτε να λαμβάνει υπόψη τη και την ευρωπαϊκή διάσταση του εκάστοτου ε, έργου. Δεύτερον, η ανάγκη Μακροπρόθεσμη μακροπρόθεσμης θεώρησης. Ε, το 2012 ε, απέχουν 8 χρόνια από τη στρατηγική 2020. Ε, θα πρέπει κάθε χρόνος να εξετάζεται ως το 1 ή αντίστοιχα το κλάσμα το αντίστοιχο μέχρι να ε, έρθουμε στο 2020 και να έχουμε επιτύχει όλους τους στόχους της στρατηγικής. Στη συνέχεια, πολλοί ομιλητές πήραν το λόγο, έθιξαν πολλά ζητήματα, κυρίως το θέμα της κινητικότητας. Ένας Ρουμάνος συνάδελφος έθιξε το θέμα αυτό, κατά πόσο δηλαδή οι φραγμοί στην κινητικότητα που παραμένουν σε κάποια επίπεδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κάτι το ανησυχητικό ή θα έπρεπε να ανησυχούμε περισσότερο για την διαρροή εγκεφάλων, το brain drain που παρατηρείται σε ορισμένα κράτη-μέλη. Αναφέρθηκε και το θέμα της συνεισφοράς και της φορολόγησης των διαφορετικών φορολογικών συντελεστών και την ανάγκη να εξαλειφθούν οι ανισότητες οι φορολογικές. Συνοχή λοιπόν μεταξύ στόχων του προϋπολογισμού και δυνατότητας υλοποίησης της στρατηγικής για την Ευρώπη του 2020. Πολλά επιχειρήματα προβλήθηκαν ε, υπέρ της ε, ειδικής μέρημνας για τους νέους και, όπως είπε και ο πρόεδρος Λαμασούχ, υποβλήθηκε το αίτημα ε, να υπάρχει περισσότερη συνοχή μεταξύ των προϋπολογισμών για να επιτευχθούν συνέργειες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για να δρομολογηθούν κοινέ στρατηγικές μεταξύ ευρωπαϊκών προϋπολογισμών και εθνικών προϋπολογισμών. Είναι μια εξαιρετικά σημαντική πρόταση αυτή. Ε, θα πρέπει να αξιολογήσουμε τις επιπτώσεις όταν θα κληθούμε μεθαύριο να αξιολογήσουμε τις νέες προτάσεις για τα διαρθρωτικά ταμεία, όταν θα κληθούμε να τοποθετηθούμε επί των νέων δημοσιονομικών προοπτικών. Καλό θα ήταν να ήδη έχουμε καταλήξει σε μια κοινή ονοματολογία. Από το 2005 μιλούμε για την εναρμόνιση των χρονοδιαγραμμάτων και την εναρμόνιση των μακροοικονομικών στοιχείων επί τη βάση των οποίων καταρτίζονται οι εθνικοί προπολογισμοί. Παρόλα αυτά, μετά από 7 χρόνια ε, χρειάζεται να διανύσουμε ακόμα μεγαλύτερη απόσταση. Ε, στη συνέχεια, ε, έγινε ανταλλαγή απόψεων με τους Σουηδούς συναδέλφους ε, για τον τρόπο με τον οποίο η Σουηδία ε, διέφυγε, ε, ξέφυγε από την κρίση όταν την είχε, όταν την είχε συναντήσει. Η Σουηδία δεν οδηγήθηκε στην κατάρρευση του κράτους πρόνοιας προκειμένου να ξεφύγει από την κρίση. παρόλα όλα αυτά κατάφερε να ξεφύγει από την κρίση εκείνη την εποχή Σίγουρα ε, τότε οι συνθήκες ήταν ευνοϊκές, ε, διασκεγραφήθηκε ένας θετικός ορίζοντας για το σύνολο της κοινωνίας. Και έτσι ε, κατέστη εφικτό να ξεφύγει η Σουηδία από την κρίση. Θίξαμε και το θέμα της ανάγκης βεβαίως δημιουργίας θέσεων απασχόλησης. Και τέλος, μιλήσαμε για το ρόλο του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού και τον συσχετισμό του με τους προϋπολογισμούς των κρατών μελών. Εάν τα κράτη-μέλη αντιμετωπίζουν δυσκολίες και επιβάλλουν περικοπές και λιτότητα, θα πρέπει να περικόπτεται και να γίνεται πιο λιτός και ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός. Τίθενται όλα αυτά τα ερωτήματα. Ο Επίτροπος Λεβαντόφσκι ξεκαθάρισε ότι ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να λειτουργήσει υποστηρικτικά και μπορεί για πάρα πολλές περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να λειτουργήσει ως μοχλός στρατηγικός κινητοποίησης ε, επενδύσεων, ούτως ώστε να επιτευχθούν ε, στόχοι που έχουμε θέσει όλοι από κοινού. Από τη στιγμή που κανείς δεν με διακόπτει, ε, διότι εγώ είμαι η πρόεδρος, σας έχω μακρηγορήσει. Θα πρέπει λοιπόν ε, να έχω περισσότερη πειθαρχία να δώσω το λόγο σε εσάς κυρία Υπουργέ, ε, για να μας μιλήσετε σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε εν ώψη και της Εαρινής Συνόδου Κορυφής. Θα μας πείτε ε, ποια είναι η διάγνωση που έχουν βγάλει οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Οικονομίας και Οικονομικών για την κρίση αυτή, το Συμβούλιο ΕΚΟΦΗΝ, τι φρονεί και πώς θα αντιμετωπιστούν και θα εξεταστούν τα θέματα αυτά από την ειρηνή Σύνοδο Κορυφή. Σας δίνω μέσω το λόγο, παρακαλώ. Well, thank you very much. Η Προεδρεύουσα στα αγγλικά. Ευχαριστώ πολύ πρώτα για την εισαγωγή σας αλλά και για την πρόσκληση. Πρώτα-πρώτα η έννοια της στρατηγικής Ευρώπης 2020. Τον τελευταίο ένα, ενάμιση, δύο χρόνια οι στόχοι άλλαξαν διότι για να επιτύχουμε τους στόχους 2020 η πορεία πρέπει βέβαια να γίνει μέσα σε ένα πλαίσιο οικονομικής κρίσης. Γι' αυτό και με ενδιαφέρει ιδιαίτερα η σημερινή συζήτηση, διότι νομίζω ότι συμμετέχουν οι πιο σημαντικοί φορείς εδώ, δηλαδή Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Εθνικά Κοινοβούλια, Κομισιόν, Συμβούλιο, επίσης οι κοινωνικοί εταίροι. Με ικανοποίηση ιδιαίτερα συζήτηση με τους κοινωνικούς εταίρους πρότινος, Επίσης και για τις μακροοικονομικές ανισότητες και το τι θα πρέπει να γίνει. Διότι είναι προφανές ότι σε μια κατάσταση κρίσεως πρέπει να φροντίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους να έχουμε μαζί μας. Υπάρχουν πέντε λοιπόν πράγματα που θέλω να θέσω υπόψη σας που θεωρώ ότι είναι σημαντικά στοιχεία για την διαχείριση της κρίσης και για την αναζήτηση διεξόδων. Πρώτα, πρώτα η σταθεροποίηση. Νομίζω ότι η συμφωνία που έγινε για την Ελλάδα είναι σημαντική, πολύ σημαντική. Για να μην επιταχύνουμε, αλλά ταυτόχρονα να είμαστε και πάρα πολύ προσεκτικοί, να ψάξουμε να βρούμε δηλαδή τους παράγοντες που θα μας επιτρέψουν να επιβραδύνουμε την κρίση, να σταθεροποιήσουμε τουλάχιστον την κρίση, να μην επιταχύνεται. Δεύτερο, να έχουμε ένα χρηματοπιστωτικό τομέα που να λειτουργεί. Να αποφύγουμε το credit crunch, την έλλειψη δηλαδή πιστώσεων, διότι οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ιδίω χρειάζονται τραπεζικό τομέα που να λειτουργεί. Τρίτο, κάθε χώρα να προβεί σε εξυγίανση, σε ευφυή εξυγίανση των δημοσιονομικών της με τρόπο που να είναι φιλικός προς την ανάπτυξη. Και ε, αυτά είναι και τα θεμέλια του Fiscal Compact. Εξυγίανση δηλαδή, αλλά είναι πολύ σημαντικό να εξεταστεί και ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει, που είναι πάρα πολύ σημαντικός. Τέταρτο, οι μεταρρυθμίσεις σε κάθε χώρα μέλος που θα διασφαλίσουν ότι οι πολίτες, τα κοινοβούλια, οι κυβερνήσεις θα σεβαστούν τις αλληλημένες υποχρεώσεις και ότι όσα αποφασίζονται εδώ θα εφαρμόζονται στις χώρες μέλη και ως πέμπτη διάσταση είναι τα σχέδια για την ευρωπαϊκή ανάπτυξη. Και άκουσα και στη συζήτησή σας να παίζει πολύ σημαντικό ρόλο αυτό δηλαδή ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός και για την πολιετή δημοσιονομική προοπτική να στοχεύει ιδιαίτερα στους στόχους της Ευρώπης 2020 και στην διαχείριση της κρίσης και όπου είναι δυνατόν να στηρίζει την ανάπτυξη. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει αυτή η ισορροπία αλλά και η δυναμική ανάμεσα στα εθνικά κοινοβούλια στου εθνικού προπολογισμού και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό γενικά. Βέβαια και η μεταρρύθμιση τη ενιαία αγορά που είναι πάρα πολύ σημαντική. Και πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση σε αυτούς τους παράγοντες ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λίγες παρατηρήσεις τώρα που θα επιτρέψουν να πούμε σε περισσότερο βάθος για ορισμένα άλλα πράγματα. Ένα από τα σημαντικά στη συζήτηση αυτή είναι να τονιστεί ότι η εξυγένση και τα υγιή δημόσια οικονομικά δεν είναι απαραίτητα αντιφατικά με την ανάπτυξη και τη δημιουργία απασχόλησης. Μάλιστα αντίθετα, η εξυγίανση αποτελεί προϋπόθεση για μια βιώσιμη ανάπτυξη. Αυτά είναι απλά ξεκάθαρα πράγματα ότι η δημόσια, ή μάλλον εξυγίανση των δημοσίων οικονομικών αποκαθιστά την αξιοπιστία. Επομένως και την οικονομική σταθερότητα και τα χαμηλά επιτόκια. Χαμηλά και σταθερά επιτόκια που να είναι προσιτά και που είναι σημαντικά για να ξεκινήσουν οι ιδιωτικές επενδύσεις και η κατανάλωση. Και οι θετικές επιπτώσεις της αξιοπιστίας είναι πολύ σημαντικές. Πάρα πολύ σημαντικές, ιδίως στην σημερινή κατάσταση, όπου η εμπιστοσύνη η αξιοπιστία όχι μόνο στις αγορές αλλά και στην πολιτική ηγεσία είναι κρίσιμες. Και πρέπει να φροντίσουμε όχι μόνο οι αγορές αλλά ίσως ακόμη περισσότερο οι επιχειρήσεις και οι καταναλωτές να είναι βέβαιοι ότι μπορούν να εμπιστεύονται τις πολιτικές τους ηγεσίε, είτε πρόκειται για βουλευτές, εθνικούς, ευρωβουλευτές, το Συμβούλιο και ούτω καθεξής. Έτσι λοιπόν, ναι μεν είναι προϋπόθεση η εξυγίανση, δεν είναι όμως φρένο στην ανάπτυξη. Να δοθούν επίσης προτεραιότητες στην παιδεία, στην, ε, στην περιβαλλοντική διάσταση, το πρασίνισμα δηλαδή και ούτω καθεξής. Πρέπει να εκπληρώσουμε υποχρώσεις και δεσμεύσεις που έχουν αναλυθεί για την εξυγένση και για τις μεταρρυθμίσεις. Πρέπει η μεταρρυθμιστική προσπάθεια να ενταθεί, γιατί αλλιώς καθυστερούμε και τρέχουμε λαχανιασμένοι πίσω από τις αρνητικές συνέπειες της κρίσης με αποτέλεσμα να αυξάνεται η ανεργία σε πολλές χώρες. Οι, πρόκλησεις, που αντιμετωπίζουμε μας αναγκάζουν να συνεργαστούμε ευθέως και άμεσα και ανοιχτά. Το έχουμε ξανακάνει και με την δέσμη 6 μέτρων. Εάν το ίδιο πνεύμα διέπει και τώρα τις ε, συζητήσεις μας θα μας βοηθήσει να υπερβούμε την κρίση. Όπως είπα προηγουμένως, θαυμάζω πραγματικά αυτούς που εργάστηκαν για την δέσμη των 6 μέτρων, για το six pack και για το έργο που έγινε για το Σύμφωνο Ανάπτυξης και Σταθερότητας και από τους κύριους στόχους, από τις κύριες προτεραιότητες της Δανικής Προεδρίας είναι η εφαρμογή αυτών των νέων και βελτιωμένων κανόνων της ε, Ευρωπαϊκής Οικονομικής Συνεργασίας η εφαρμογή είναι κρίσιμη, διότι αλλιώς δεν είμαστε παρά μια μηχανή που εκδίδει αποφάσεις που όμως δεν εφαρμόζονται, δεν έχουν σχέση με την καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Πρέπει λοιπόν να, υλοποιηθεί, να υλοποιηθούν οι στόχοι του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, να λάβουμε υπόψη τα όσα λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για τις ε, υπηρεσίες αλλά και για, την, για τις μακροοικονομικές ανισότητες και προς την κατεύθυνση αυτή να φροντίσουμε ώστε και οι εθνικές βουλές και οι κυβερνήσεις να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Στο ευρωπαϊκό τώρα επίπεδο περνούμε από την δέσμη 6 μέτρων και με τις επόμενες δύο προτάσεις που βεβαια six 6-pack αυτές τώρα λεγονται two 2-pack είναι καταπληκτική αυτή η ιδιαίτερη γλώσσα των ε, ευρωκρατών ουδής καταλαβαίνει απ' έξω τι εννοούμε αλλά τέλος πάντων το περιεχόμενο έχει σημασία, να γνωρίζουμε δηλαδή τι κάνει η κάθε μια χώρα. Και εάν μια χώρα αντιμετωπίζει προβλήματα, να παρακολουθούμε προσεκτικά, όπως έγινε και πριν, όπως γίνεται. Και το Συμβούλιο την προηγούμενη εβδομάδα κατέληξε σε συμφωνία για τις δύο αυτές προτάσεις και θα θέλαμε να αρχίσουμε τον τριμερή διάλογο σύντομα όταν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα είναι έτοιμο να προσέλθει στον τριμερή αυτό διάλογο. Ένα πράγμα που θα ήθελα τώρα να μας απασχολήσει να σας αναπτύξω δηλαδή με λίγα λόγια τώρα που ολοκληρώνω σιγά σιγά την ομιλία μου είναι ο ρόλος των εθνικών βουλών που πρέπει να ενισχυθεί καθώς επίσης και η συνεργασία τους με το ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι κρίσιμο οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται στην Ευρώπη να φτάνουν και μέχρι τις χώρες διότι αυτά που υπόσχεστε στο ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να είναι υποσχέσεις που θα τηρηθούν και στις χώρες σας. Αυτό άλλωστε είναι και η ιδέα που βρίσκεται μέσα στο Fiscal Compact. Αυτά δηλαδή που υποσχόμαστε στο ευρωπαϊκό επίπεδο, στο επίπεδο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, θα τα κάνουμε στις χώρες μας. Διότι τότε μόνο αποκαθίσταται ο πολύ στενό σύνδεσμος ανάμεσα σε μια ε, ευρωπαϊκή αντίληψη και στην εθνική αντίληψη. Το, η νέα Δημοσιονομική Συμφωνία, το νέο Fiscal Compact, αποτελεί μια καινοτομία, διότι προβλέπει συγκεκριμένες δημοσιονομικές δεσμεύσεις και αποτελεί επομένως μια προστιθέμενη αξία στην ευρωπαϊκή οικονομική διαχείριση. Τώρα στο εθνικό επίπεδο βέβαια η εφαρμογή σημαίνει έγκριση των συγκεκριμένων προπολογισμών που να σέβονται, ελπίζω, ελπίζω τις συμφωνημένες συστάσεις και προσαρμογές, γιατί αυτή είναι βασικά η ιδέα. Δηλαδή, συλλέγουμε όσο, όσο γίνεται περισσότερες πληροφορίες, συζητούμε στη βάση τους μαζί με τους κοινωνικούς εταίρους και με το Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο, όπως έγινε πριν από λίγες μέρες, και όλες αυτές οι πληροφορίες αποκρισταλώνονται εν τέλει σε, σε μια συμφωνημένη πορεία. Ελπίζω λοιπόν ότι η σημερινή συζήτηση και αυτή θα δείξει ότι συμφωνούμε το ποιε συστάσεις να δώσουμε σε ό,τι αφορά μια, δημόσια, μια, μια δημοσιονομικών φιλική προς την ανάπτυξη, με ανάπτυξη, με παιδεία, με περιβαλλοντική ε, διάσταση και ούτω καθεξής. Δεν υπάρχει και άλλος τρόπος. Όλοι γνωρίζετε τι κάνουμε και για την νομοθεσία για την ενιαία αγορά. Ολοκληρώνω λέγοντας ότι αναμένω με ενδιαφέρον τη συζήτηση καθώς επίσης και τη συνεργασία με τα εθνικά Κοινοβούλιο αλλά και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο υπόλοιπο του, ε, εξαμήνου, του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, δεν θέλησα να σας διακόψω. Θα παρακαλέσω όμως τον Επίτροπο που θα λάβει τώρα τον λόγο να είναι πιο σύντομος, πιο μέσα στα ευρωπαϊκά πλαίσια των χρόνων αγόρευσης και να εξηγήσει και με ποιο τρόπο βλέπει, σε ποιο πνεύμα βλέπει τον διάλογο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να εξηγήσει δηλαδή την ευρωπαϊκή διάσταση της ε, πολιτικής ανάπτυξης. Ως γνωρίζετε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κινητοποιείται μέσα στο πλαίσιο του πρώτου τριμήνου του έτους ε, να προωθήσει την εξέταση ε, και των εγγράφων προς ανατολισμού. Έχουμε δύο εκθέσεις, Jean-Paul Gauzès, Οικονομική Διάσταση, και η κυρία Κονέλσεν για την απασχόληση. Διάβασα κάπου ότι ορισμένοι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρούν ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάνοντας αυτό προσπαθεί να προκαταλάβει τα θέματα του Εαρινού Συμβουλίου. Δεν είναι αληθές αυτό. Εμείς θέλουμε να εμφυσίσουμε ζωή στην κοινοβουλευτική διάσταση της συζήτησης, της δημόσιας, της κοινής αυτής συζήτησης. Ίσως μπορείτε λοιπόν αγαπητέ κύριε Επίτροπε, να εξηγήσετε με ποιον τρόπο βλέπετε αυτή την κοινοβουλευτική διάσταση του διαλόγου και βεβαίω και σε συνεργασία με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Για πέντε λεπτά, κύριε Επίτροπε. Α, με συγχωρείτε, δέκα λεπτά. Δέκα λεπτά, Ευχαριστώ, Περιβάλλον. Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Εθνικών Κοινοβουλίων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαι ευτυχής που μπόρεσα να ακούσω τα πορίσματα από τις συζητήσεις για το Ευρωπαϊκό Εξάμενο εχθές και σήμερα. Και είμαι ευτυχής που μπορώ να τα συζητήσω μαζί σας. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Μπόουλ και τον κύριο Λαμασούρ για τι πολύ, ε, τις πολύ ουσιαστικές και σύντομες εκθέσει που έκαναν για τους διαλόγους και τις συζητήσει που κάνατε κατά τη διάρκεια αυτή τη διάσκεψης. Είναι λίγαν ενθαρρυντικό να βλέπουμε ότι αποκτά μία τακτική ε, μορφή αυτή η συνεδρίαση των, η διακοινοβουλευτική γιατί είναι πολύ σημαντικό και η λογοδοσία ιδιαίτερα σε μια περίοδο κρίσης όπως αυτή που διανύουμε. Και μόνο εσείς ως εκλεγμένοι εκπρόσωποι των Ευρωπαίων πολιτών μπορείτε να εξασφαλίσετε αυτή την λογοδοσία και τη δημοκρατική νομιμότητα. Έχουμε κάνει πολλά τα τελευταία δύο χρόνια, ολοκληρώνοντας την Οικονομική και Νομισματική Ένωση με την κατάλληλη αρχιτεκτονική, ώστε να υπάρχει ενισχυμένη οικονομική διακυβέρνηση. Οι νέες δομές σημαίνουν πως τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη θεωρούν κοινέ τις πολιτικές τους για το, καθώς και το σύμφωνο για την οικονομική ε, το σύμφωνο για την σταθεροποίηση ε, και την ανάπτυξη όπως προβλέπεται από τις ε, συνθήκες. Αυτό σημαίνει επίσης συντονισμό των πολιτικών σχεδίων πριν από τις τελικές εθνικές αποφάσεις και όχι μόνο κατόπιν μάλλον εκ των υστέρων όπως συνέβαινε παλιότερα και χωρίς επαρκή επιτυχία όσον αφορά τον αποτελεσματικό συντονισμό των πολιτικών. Ακριβώς ε, το νόημα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου είναι το να διευκολύνει αυτήν την εκ των προτέρων ε, συνεννόηση και συντονισμό και γι' αυτό και η συμμετοχή όλων είναι τόσο σημαντική σε αυτή την προσπάθεια. Το ευρωπαϊκό εξάμενο φέτος, το 2012, είναι το πρώτο πραγματικό με το εξαπλό πακέτο μέτρων που ισχύει ήδη. Είχαμε και τον προηγούμενο χρόνο εξάμεινο, αλλά πρώτη φορά ισχύει το six-pack έτσι ώστε να εντοπιστούν οι δημοσιονομικές και οικονομικές ανισορροπίες των κρατών μελών πολύ νωρίτερα από ό,τι παλιότερα. Ιδιαίτερα στην Ευρωζώνη οι οικονομικές και οι δημοσιονομικές σχέσεις είναι τόσο βαθιές ανάμεσα στα κράτη-μέλη και οι συνέπειες των αποφάσεων του ενός κράτους μέλους επί των υπολείπων τόσο άμεσες που χρειάζεται ακόμα μεγαλύτερη ολοκλήρωση για την ομαλή λειτουργία της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μετά από την ε, Δημοσιονομική Συμφωνία, την οποία συνυπέγραψαν 25 κράτη-μέλη και ελπίζω θα την επικυρώσουν και όλοι σε αυτό το χρόνο, αυτό λοιπόν συμφωνεί Μάλλον μετά από αυτή τη δημοσιονομική συμφωνία, τον Νοέμβριο φτιάξαμε άλλε δύο συμπληρωματικέ προτάσεις για να συμπληρώσουμε το εξαπλό πακέτο όσον αφορά την αυξημένη παρακολούθηση και εποπτεία για τα κράτη-μέλη του Ευρωζώνης. Η πρώτη ε, αφορά τα χρονοδιαγράμματα για την, την ευθυγράμμιση των προγραμμάτων για την προετοιμασία των προϋπο... εθνικών προϋπολογισμών και την υποβολή τους και εξέτασή τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο πριν την τελική τους έγκριση. Η δεύτερη πρόταση αφορά την αυξημένη εποπτεία στα κράτη-μέλη που αντιμετωπίζουν κινδύνους για την ε, ε, δημοσιονομική του σταθερότητα και άρα αποτελούν κίνδυνο για τη δημοσιονομική σταθερότητα άλλων κρατών μελών της Ένωσης. Είναι σαφές ότι αυτές οι προτάσεις που κάνουμε σημαίνουν ε, συντονισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο των εθνικών πολιτικών. περιλαμβάνεται δε και η δυνατότητα ε, η Κομισιόν να ζητήσει ένα αναθεωρημένο σχέδιο προπολογισμού από κάποιο κράτος μέλος σε περίπτωση ιδιαίτερα σημαντικής απόκλησης από τις υποχρεώσεις τις δημοσιονομικές. Γιατί το κάνουμε αυτό? Έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι τα κράτη-μέλη σέβονται θα σέβονται τους κανόνες τους οποίους τα ίδια αποφάσισαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όλοι αυτοί οι κανόνες αποφασίστηκαν ομόφωνα στο Συμβούλιο από τα 27 κράτη-μέλη μαζί με το Ευρωκοινοβούλιο. Και είναι δικό μας έργο της Κομισιόν να εξασφαλίσουμε τον σεβασμό αυτών των κανόνων στις χώρες μας. Είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι αυτή ο βαθύτερο συντονισμό είναι απαραίτητο για να λειτουργήσει η Οικονομική και Νομισματική Ένωση και να ε, ε, γίνει αρκετά στεναρή ώστε να μπορεί να αντισταθεί και να ξεπεράσει τις ε, κρίσεις όπως αυτήν που πρόσφατα γνωρίσαμε και εξακολουθούμε να ζούμε. Είναι σαφές ότι η πρόληψη είναι πάντοτε καλύτερη από την διόρθωση, τη θεραπεία. Και αυτός είναι και ο πυρήνας ε, του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και των νέων, νέας οικονομικής ε, διακυβέρνησης. Κυρίες και κύριοι, οι κανόνες και οι απαιτήσει ε, δεν είναι βεβαίως στόχοι. Είναι μόνο μέσα για να εξασφαλίσουμε ότι οι πολιτικές που έχουν στόχο την επίτευξη καλύτερης ανάπτυξης, περισσότερης ανάπτυξης και επασχόλησης, σταθερότητας, κοινωνικής προόδου θα εφαρμοστούν αποτελεσματικά. Είναι η ουσία των πολιτικών μας που τελικά έχει τη μεγαλύτερη σημασία και επί της οποίας θα ήθελα να εστιάσω την υπόλοιπη μου παρέμβαση. Όπως είπε η Πρόεδρος κυρία Μπερές, και αναφέρθηκε στη ΣΥΠΑ, τον παγκόσμιο πτέρο μας, γι' αυτό και θα ήθελα να αναφερθώ στην συνεδρίαση του G20 ε, που πρόκειται για τους παγκόσμιους εταίρους μας και όπου είχα την ευκαιρία να αντιπροσωπεύσω, να εκπροσωπήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μαζί με την ε, δανική κυβέρνηση και προεδρία. Συναντηθήκαμε λοιπόν στο πόλη του Μεξικό και ασχοληθήκαμε με τις συνεχιζόμενες ε, οικονομικές προκλήσεις και δυσκολίες. Και αυτή τη στιγμή ένιωσα να επικρατεί πιο ε, θετική ατμόσφαιρα στους 20 σε σχέση με την κρίση ε, και την αντιμετώπιση αυτή στην Ευρώπη. Ήταν σημαντικό οι 20 να αναγνωρίσουν την πρόοδο που έχει σημειώσει η Ευρώπη τους τελευταίους μήνες όσον αφορά την ανταπόκρισή μας στην κρίση, τον οδικό μας χάρτη για τη σταθερότητα και την ανάπτυξη, να ενισχύσουμε τη δημοσιονομική μας θέση στην Ιταλία ή στην Ισπανία ή και σε άλλες χώρες, να υιοθετήσουμε μέτρα για την μείωση του, δημοσιονομικού, ε, της δημοσιονομικής πίεσης, να οικοδομήσουμε ισχυρότερου θεσμούς σε σχέση με την μεταρρύθμιση της ε, διακυβέρνησης, την εφαρμογή διαρθρωτικών μέτρων που προωθούν την ε, ανάπτυξη και να βάλουμε και την Ελλάδα σε μια βιώσιμη πορεία. Ήταν σημαντικό λοιπόν οι 20 να αναγνωρίσουν ότι κάνουμε προσπάθειες για την ε, αντιμετώπιση της κρίσης, οι οποίες αποδίδουν καρπούς. Επίσης, ξεκινήσαμε το, εξηγήσαμε μάλλον το εξάμεινο και εξηγήσαμε και ότι η φιλική ε, δημοσιονομική εξυγίανση είναι απαραίτητη, γιατί η εμπιστοσύνη είναι το κλειδί στην ανάπτυξη για την ανάπτυξη. Όμως και η ανάπτυξη μόνη της δεν μπορεί να προωθήσει όλο μας το δυναμικό και γι' αυτό χρειάζονται στρατηγικές που θα αποτελέσουν το κλειδί για την οικονομική μας στρατηγική και για την ανταπόκριση στην κρίση. Από ό,τι φαίνεται όμως δεν έχω πολύ χρόνο, γι' αυτό και θα κλείσω, θα ολοκληρώσω λέγοντας ότι η επίτευξη της ανάπτυξης και η δημιουργία θέσεων απασχόλησης είναι πολύ μεγάλη πρόκληση σε περίοδο περιορισμών και δημοσιονομικής λιτότητας, αλλά πολλά κράτη-μέλη κατάφεραν να ξεπεράσουν την κρίση μέσω αποφασιστικής δράσης. Σκεφτείτε τις μεταρρυθμίσεις και τις προσαρμογές που έγιναν για παράδειγμα στη δεκαετία του 80 στη Δανία και στην Ολλανδία, στη Σουηδία και στη Φιλανδία τη δεκαετία του 90 ή στη Γερμανία κατά τη διάρκεια της προηγούμενης δεκαετίας. Η Ιρλανδία και η Λετωνία είναι τα πιο πρόσφατα παραδείγματα ότι η οικονομική ανάκαμψη και η επιστροφή στην ανάπτυξη μπορούν να επιτευχθούν ακόμα και σε δύσκολους καιρούς και υπό δύσκολες συνθήκες. Δεν υπάρχει λόγος αυτά τα επιτεύγματα να μην είναι δυνατά και σε άλλα κράτη-μέλη της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των χωρών των, των μνημονίων. Ε, νομίζω ότι χρειάζεται περισσότερο αποφασιστική δράση για να ε, μπούμε σε μια περίοδο σταθεροποίησης και να μπορούμε να πούμε πως έχουμε τις πιθανότητες να περάσουμε το σημείο καμπής από τη σταθεροποίηση στην ανάπτυξη και στη δημιουργία θέσεων. Πιστεύω πως αυτό το βήμα είναι ένα εξαίρετος τρόπος για να δουλέψουμε προς αυτή, την επίτευξη αυτών των στόχων, όχι μόνο μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών, αλλά και καλύτερων πρακτικών, γιατί έτσι μπορούμε να βελτιώσουμε το επίπεδο της δημόσιας στήριξης για τις κοινέ μας πολιτικές και για τις μεταρρυθμίσεις που είναι τόσο ζωτικές για όλους μας τους Ευρωπαίους ώστε να επιστρέψουμε, όπως είπα, στην ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Αυτό περιμένουν οι πολίτες μας από εμά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Επίτροπε. Να δώσω το λόγο στον Επίτροπο Άντορ που χειρίζεται το χαρτοφυλάκιο των θεμάτων απασχόλησης, κοινωνικών υποθέσεων και κοινωνικής συμπερίληψης και ένταξης να επενθυμίσω ότι όσοι θέλουν να υποβάλουν ερώτημα να το υποβάλουν γραπτός και να συμπληρώσουν το πράσινο έντυπο που έχουν μπροστά μας. Έχετε το λόγο για 10 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, πιστεύω ότι η χθεσινή συνάντηση αλλά και η σημερινή συνάντηση είναι εξαιρετικά ε, σημαντικές και επί της ουσίας αλλά και επί του συμβολισμού τους ως μια νέα διαδικασία. Πλέον υπάρχει συνένεση. Είναι ανάγκη να ξεπεράσουμε τη δημοσιονομική πειθαρχία και να μιλήσουμε και για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, για την ανάπτυξη και την συνοχή. Υπ' αυτή την έννοια, με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο ε, χρειάζεται καλύτερο συντονισμό πολιτικών απασχόλησης και κοινωνικών υποθέσεων. Πέρα από τον καλύτερο συντονισμό που χρειάζεται για θέματα ε, τα δημοσιονομικά και καλύτερη συνεργασία ε, με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Και σε αυτές τις γραμμές θα κινηθεί η παρουσίασή μου. Καταρχάς πιστεύω ότι το υφιστάμενο ε, πλαίσιο, το υφιστάμενο περιβάλλον μας καλεί περισσότερο από ποτέ να εστιάσουμε την προσοχή μας στην καταπολέμηση της ανεργίας με επίγοντο τρόπο και στην αντιμετώπιση του θέματος των θέσεων απασχόλησης ως βασική προτεραιότητα. Όλα αυτά ε, κατέστησαν σαφή στο άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στα τέλη του Ιανουαρίου και θα επιβεβαιωθούν και ε, επισήμως ε, μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Η δημοσιονομική εξυγίαση δεν θα πρέπει να υπονομεύει τις δαπάνες που ενισχύουν την ανάπτυξη, π.χ. τις δαπάνες στην εκπαίδευση, τις δαπάνε στην κατάρτιση των ανέργων. Είναι ζωτικής σημασίας να έχουμε σταθεροποιητές ε, κοινωνικούς και να δοθούν απαντήσεις στις ασυμμετρίες στην ευρωπαϊκή οικονομία. Σε αυτό το χάσμα δηλαδή που βαθαίνει μεταξύ χωρών με πολύ καλούς δείκτες επιδόσεων ε, και ε, ως προς τα, χρηματο... ως προς τα δημοσιονομικά έσοδα και την απασχόληση και χώρες με πολύ κακούς δείκτες και πολύ κακούς επιδόσεις στα θέματα αυτά. Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουμε εντοπίσει στη μελέτη μας τις βασικές προτεραιότητες που θα πρέπει για μας να υιοθετηθούν από όλους. Πρώτον, να ενισχύσουμε τις προσπάθειές μας για να δημιουργούνται περισσότερες θέσεις απασχόλησης στην Ευρώπη. Δεύτερον, ε, καταπολέμηση της ανεργίας των νέων. Ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, έχουμε αναλάβει δράση για να λυθεί το πρόβλημα αυτό βάσει της πρωτοβουλίες για τις ευκαιρίες στους νέους, μια πρωτοβουλία που υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τον περασμένο Δεκέμβριο. Τα κράτη-μέλη πρέπει να καταρτήσουν συνολικές στρατηγικές για την απασχόληση των νέων, να εντοπίσουν ανάγκες, να προτείνουν τοπικές δράσεις στα εθνικά σχέδια δράσης για την απασχόληση. Τρίτον, η μακροχρόνια άνεργη. Ε, χρειαζόμαστε συγκεκριμένα εστιασμένα μέτρα για να αποφύγουμε τη διαρθρωτική ανεργία και να αποφύγουμε τον κοινωνικό αποκλεισμό. Τέταρτον, να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα των συστημάτων κοινωνικής προστασίας, ώστε να λειτουργήσουν προφυλακτικά ως προφυλακτήρες έναντι της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, να προλάβουν αυξήσεις στις ανισότητες και να προλάβουν την αναζωπήρηση της ε, ε, κοινωνικής οργής. Και τέλος, τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης πρέπει να εξυγχρονιστούν και να καταστούν πιο αποτελεσματικά. Χρειαζόμαστε προσεγγίσεις έγκαιρης προέ προειδοποίησης και έγκαιρης παρέμβασης για να αποφευθεί το φαινόμενο της εγκατάλειψης της σχολικής αίθουσας από πλευράς των μαθητών. Έχουμε συζητήσει τις ε, εκθέσεις ε, της κυρίας ε, Κορνέλισεν και της κυρίας Μπέρες, οι οποίες εγκρίθηκαν στην τελευταία ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και έχουμε συζητήσει και τις κατευθυντήριες γραμμές του Συμβουλίου που στηρίζουν τις προτεραιότητες. Όλα αυτά μας βρίσκουν σύμφωνους όλους. Το θέμα τώρα είναι η υλοποίηση και πολλά από αυτά τα μέτρα πρέπει να τα εφαρμόσουν τα κράτη-μέλη και όχι εμείς. Έχουμε όμως κάποια κριτικά μέτρα, κάποιες πρωτοβουλίες που μπορούμε να αναλάβουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Να μιλήσω πρώτα για τα χρηματοδοτικά εργαλεία, ε, προκειμένου να βελτιώσουμε την εφαρμογή όλων αυτών ε, σε τοπικό επίπεδο. Να αναφέρω λοιπόν το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ευρωπαϊκό Ταμείο για την Προσαρμογή στην ε, Παγκοσμιοποίηση, το, το το πρόγραμμα για την μικροχρηματοδότηση των πολύ μικρών επιχειρήσεων κ.ο.κ. Ε, ε, επίσης θα γίνει συζήτηση για την επόμενη προγραμματική περίοδο για το νέο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το, το νέο Ταμείο ε, για την προσαρμογή στην παγκοσμιοποίηση και για τον επανασχεδιασμό του Eures και του Microfinancing υπό την μία και κοινή ομπρέλα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλησε όλα αυτά τα χρηματοδοτικά εργαλεία να τα συνδέσει άμεσα με την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής της Ευρώπης για το 2020 και των στόχων της απασχόλησης της στρατηγικής αυτής. Ως Επιτροπή θέλουμε να απλωστεύσουμε και να καταστήσουμε πιο σαφείς και ξεκάθαρες τις διαδικασίες. Όλα αυτά τα θέματα είναι υποσυζήτηση με το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο και έχουμε λάβει και σχόλια από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Όλα αυτά βεβαίως έχουν νόημα, δεν θα πρέπει όμως να παραμελούμε τον αληθινό μας στόχο όταν συζητούμε τις λεπτομέρειες εφαρμογής κάθε ενός από αυτά τα προγράμματα. Εάν πράγματι θέλουμε να πετύχουμε το στόχο, θέλουμε να ξαναδημιουργήσουμε δουλειές, τότε θα πρέπει να εφοδιαστούμε με τα απαραίτητα εργαλεία. Κυρίες και κύριοι, η πρωτοβουλία για τις ευκαιρίες στους νέους, Youth Opportunities Initiative, έχει ως στόχο να ενσωματώσει όλα αυτά τα συστήματα και όλα, αυτά τα προγράμματα που καταπολεμούν την ανεργία των ε, νέων. Ε, σε οχτω κράτη-μέλη η κατάσταση είναι αρκετά ε, κρίσιμη και θα ξεκινήσουμε την πρωτοβουλία από αυτές τις χώρες. Αν θέλετε μπορώ να μπω σε περισσότερες λεπτομέρειες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει μια αρχική αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίο εφαρμόστηκε η πρωτοβουλία για τις ευκαιρίες στους νέους στο άτυπο Συμβούλιο Απασχόληση και Κοινωνικών Υποθέσεων, στο άτυπο Συμβούλιο Υπουργών του Απριλίου. Χρειάζονται περισσότερες καινούριες ιδέες, περισσότερες νέες πρωτοβουλίες, περισσότερη αποφασισμένη και αποφασιστική δράση. Η βιώσιμη ανάπτυξη που θα συμπεριλαμβάνει όλους θα εξαρτηθεί από τη δυνατότητα της Ευρώπης να δημιουργεί θέσεις απασχόλησης και να ε, προβαίνει στις απαραίτητες διαρθρωτικές αλλαγές. Θα πρέπει η οικονομία μας να πρασινίσει περισσότερο, ε, στην ημερησία διάταξη να έχουμε περισσότερο την βιώσιμη ανάπτυξη. Ε, θα πρέπει να, να αντιμετωπίσουμε τη δημογραφική πρόκληση, τη γύριση του πληθυσμού και να γνωρίζουμε ότι ε, η τεχνολογία της επικοινωνίας και των πληροφοριών θα είναι πάντοτε στο προσκήνιο. Όλα αυτά σκιαγραφούν το τοπίο στο μέλλον και σε αυτό το πλαίσιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει μία δέσμη εργαλείων ε, τα οποία θα χρησιμοποιήσουμε για να στηρίξουμε την αγορά εργασίας, να αντιμετωπίσουμε ας πούμε τις, ε, ε, το λάθος τέριασμα μεταξύ θέσεων απασχόλησης από τη μία και προσόντων του ετούντα τη, τη συγκεκριμένη θέση από την άλλη πιο αυστηρή οικονομική διακυβέρνηση έχει θεσμοθετηθεί με την δέσμη 6 μέτρων. Απαιτείται περισσότερη δημοσιονομική πειθαρχία, αλλά απαιτείται και περισσότερο συντονισμό όλων αυτών των ε, πολιτικών με την πολιτική για την απασχόληση και ε, απαιτείται και διόρθωση των μακροοικονομικών ανισορροπιών. Υπό αυτή την έννοια, η εμπλοκή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η συμμετοχή των Εθνικών Κοινοβουλίων έχει, ε, είναι ζωτική σημασία για περισσότερη διαφάνεια ε, και περισσότερη δημοκρατική νομιμότητα σε αποφάσει που λαμβάνονται. Εξού και ο νέο οικονομικό διάλογο για του δύο αυτού κανονισμού είναι εξαιρετικά σημαντικό. Και θέλω να επιμείνω και σε μια άλλη διάσταση τη ευρωπαϊκή διακυβέρνηση. Χρειαζόμαστε ε, κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό ε, να υπάρχει ισορροπία στις μεταρρυθμίσεις. Οι πολιτικές για την απασχόληση και οι κοινωνικές πολιτικές πρέπει να ε, είναι καλύτερα συντονισμένες. Και όλα αυτά αναφέρονται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου Υπουργών αλλά και τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Δεν είναι εύκολα όλα αυτά. Ε, η απασχόληση εμφανίζεται στην μικροοικονομική θεωρία και η ανεργία εμφανίζεται στην μακροοικονομική θεωρία. Συχνά λένε οι πανεπιστημιακοί και είναι δύσκολο να υπάρχει συνέπεια και συνοχή μεταξύ των δύο. Ωστόσο, η απασχόληση, η παραγωγικότητα, η ανταγωνιστικότητα είναι δείκτες που εντοπίζουν εν δυνάμει μακροοικονομικές ανισορροπίες οι οποίες επηρεάζουν τις αγορές εργασίας σίγουρα. Επομένως, πρέπει ε, τα αντίστοιχα συμβούλια ε, Υπουργών Οικονομικών να ε, αναλάβουν την ευθύνη που τους αναλογεί στο συντονισμό όλων αυτών των πολιτικών. Και τέλος θα ήθελα να τονίσω ότι βεβαίως δεν αρκεί να μοιραζόμαστε τις βέλτιστες πρακτικές, πρέπει να παρακολουθούμε καλύτερα τον τρόπο εν τον οποίο εφαρμόζονται αυτά στα κράτη-μέλη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μεριμνήσει για όλα αυτά, στηριζόμενη στο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στο ρόλο των Εθνικών Κοινοβουλίων. Καλωσορίζουμε τη συμμετοχή των Εθνικών Κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε όλο αυτό το εγχείρημα. Εξού και είναι εξαιρετικά σημαντική αυτή η μερίδα για μας, αυτός ο διάλογος που εκτελήσετε αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ. Η Πρόεδρος, ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Ε, πολλοί έχουν ζητήσει το λόγο. Θα ήθελα να σας πω ότι δεν πρέπει να ξεπεράσετε τα δύο λεπτά ο καθένας. Να δώσω το λόγο στον κύριο Φιλίπ Μαρινή, ε, πρόεδρο της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Γαλλικής Γερουσίας. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Έφτασα χθες ε, κάπου, και το πνεύμα μου ήταν κάπως σκεπτικιστικό. Αναρωτιόμουν ε, ποια θα ήταν η χρησιμότητα αυτής της ε, συνεδρίασης. Και ε, αυτή τη στιγμή έχει μετριαστεί η αρνητική μου εντύπωση, αν θέλετε. Έχουμε καλά στοιχεία και κάποια λιγότερο καλά στοιχεία. Τα καλά στοιχεία είναι το γεγονός ότι δεν έχει ξαναοργανωθεί τέτοιου είδου συνάντηση. Ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Εθνικά Κοινοβούλια. Λιγότερο καλό στοιχείο είναι ότι θα έπρεπε να υπήρχε καλύτερη προετοιμασία επί συγκεκριμένων ε, ε, πτυχών. Ε, ε, επί συγκεκριμένων σημείων της ημερήσιας διάταξης, να αποφύγουμε τη γενικότερη κοινοβουλευτική συζήτηση και το ε, διαλέγεστε επί αφηρημένων ενιών. Είναι πολύ ενδιαφέρον να ακούμε την άποψη των Βρετανών συναδέλφων που δεν είναι καν στο ευρώ. Όμως δεν έχει και πολύ μεγάλη σχέση αυτό με τις παρατηρήσεις του Ευρωπαίου Επιτρόπου ε, οι οποίες ε, κοιμάθηκαν στη σφαίρα των γενικών πολιτικών παρατηρήσεων. Αυτά ε, δεν συμβάλλουν όλα αυτά στις εργασίες μας. Πρέπει να είμαστε πιο συγκεκριμένοι για να είμαστε και πιο χρήσιμοι. Να ορίσουμε συγκεκριμένους όρους. Six pack, two pack, δέσμοι 6 μέτρων, δέσμοι 2 μέτρων, νέα δημοσιονομική συμφωνία, Europlus Pact. Όλα αυτά θα αλλάξουν δραματικά τον τρόπο, τη μεθοδολογία δουλειά των εθνικών κοινοβουλίων κοινοβουλίων. Ε, αυτό σημαίνει να είναι κανείς κοινοβουλευτικός. Δεν είναι κοινοβουλευτικός για να αγορεύει ε, μόνο και μόνο για να εκφράζει πολιτικώς ορθές απόψεις, ε, τις οποίες άλλωστε η κοινή γνώμη δεν ακούει. Η κοινοβουλευτική δραστηριότητα είναι μια τεχνική δραστηριότητα μεταξύ άλλων και θα πρέπει λοιπόν να είμαστε πιο συγκεκριμένοι. Και εκφράζω αυτή την τοποθέτηση για να βελτιωθεί η οργάνωση των εργασιών μας. Ευχαριστώ, λέει η πρόεδρος, να δώσω το λόγο στον ε, Ιρλανδό συνάδελφο από την ε, Επιτροπή ε, του Ιρλανδικού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε. Thank you, Madam Thank you for the opportunity. Σας ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία να σας απευθύνω το λόγο είναι ένα πολύ καλό διδακτικό εγχείρημα. Εμείς ακούμε και μαθαίνουμε τις εμπειρίες των άλλων ε, κοινοβουλευτικών των άλλων κρατών μελών, από τα κοινοβούλια των άλλων κρατών μελών και αυτό με βοηθάει ιδιαιτέρως. Με ανησυχεί ωστόσο ε, το ότι δεν έχουμε θίξει το θέμα της τραπεζικής κρίσης, της κρίσης του τραπεζικού τομέα. Δεν έχουμε μιλήσει αρκετά για όλο αυτό. 23 εκατομμύρια μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 23 εκατομμύρια άνθρωποι είναι άνεργοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Ιρλανδία, για να σας παρουσιάσω την ε, εικόνα, έχουμε έλλειμμα 10% σε σχέση με το ΑΕΠ. Έχουμε τεράστιο εθνικό χρέος, το οποίο ε, δημιουργήθηκε διότι εμείς αφομοιώσαμε το τραπεζικό ε, χρέος και ε, θα φτάσουμε στο 119% ε, του ΑΕΠ φέτος. 15% του ΑΕΠ μας αυτή τη χρονιά αφιερώθηκε ως διαρθρετικά μέτρα. 25 δις ευρώ δηλαδή βγήκαν από την οικονομία για να μειωθεί το χρέος ο τραπεζικός τομέας παρά την ανακεφαλαιοποίηση δεν μπαίνει ενεργητικά στην οικονομία. Επομένως θέτω αυτά τα ερωτήματα. Ποιος είναι ο ρόλος της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Πώς θα βοηθήσει για να λυθεί, ε, να ξεπεραστεί η τραπεζική κρίση. Βεβαίως ήμασταν υπεύθυνοι για το χρέος μας. Όμω η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δάνεισε πολύ φτηνό χρήμα στι ε, τράπεζε και τελικά οι οικονομίε δεν βοηθήθηκαν και ε, εθνικοποιήσαμε πολύ τοξικές τράπεζες με ένα κόστος τεράστιο για το φορολογούμενο και διασώσαμε ε, τους, τραπε... Ε, τους τραπεζίτες ενδεχομένως ή τους προφυλάξαμε από το να καταβάλουν μεγάλη προσπάθεια. θα ήθελα ένα σχολιασμό γι' αυτό, όπως επίσης θα ήθελα και να σχολιαστεί γιατί για σε να σχολιαστεί το θέμα του πώς κάποιες χώρες μέλη κατάφεραν να ξεπεράσουν την κρίση. Η Σουηδία στη δεκαετία του 90, για παράδειγμα, χωρίς την κατάρρευση του κοινωνικού της κράτος. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει η εκπρόσωπος από την Κύπρο. Παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, ε, συμμεριζόμαστε τις ανησυχίες που έχουν διατυπωθεί από διάφορες κατευθύνσεις σε σχέση με τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί τον περασμένο Δεκέμβριο από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για δημοσιονομική πειθαρχία. Πρόκειται για αλλαγές που στο όνομα της νομισματικής σταθερότητας οδηγούν σε περαιτέρω εκχώρηση της κρατικής κυριαρχίας των μελών της Ένωσης ενώ η ρήτρα για μόνιμα ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς οδηγεί σε περαιτέρω υποχώρηση των κοινωνικών πολιτικών διολίσθηση των εργασιακών σχέσεων και δικαιωμάτων, αύξηση του χάσματος μεταξύ πλουσίων και φτωχών, όξιση της ανεργίας και ειδικά της, γυναικείας και της, νεανικής και της γυναικείας ανεργίας. Η δραματική κατάσταση που βιώνει σήμερα ο ελληνικός λαός δεν είναι αποτέλεσμα της έμφυτης τεμπελιάς του, ούτε υπάρχει κάποια αθεληνική συνωμοσία. Είναι δυστυχώς το αποτέλεσμα της λειτουργίας των νόμων της αγοράς, που ισοπεδώνουν στο πέρασμά τους. Η δημοσιονομική πειθαρχία και νομισματική αυστηρότητα δεν πρέπει να αποτελεί αυτό σκοπό και περαιτέρω θα πρέπει το επίκεντρο να είναι η ανάπτυξη που αποτελεί προϋπόθεση για την αύξηση των θέσεων εργασίας. Οι προπολογισμοί σε επίπεδο κρατών μελών θα πρέπει να δίνουν έμφαση στι δημόσιε επενδύσει σε τομεί όπω την έρευνα και την καινοτομία, την πράσινη ανάπτυξη, τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Έχω ακούσει τώρα τον κύριο Νάντορ για τις ε, εισηγήσεις του σε σχέση με την ε, απασχόληση και τα θεωρούμε όλα πολύ σημαντικά. Αυτό που ήθελα να τονίσω είναι ότι χρειαζόμαστε ένα νέο σύμφωνο εργασίας και ανάπτυξης που θα επιτρέπει στα κράτη να ακολουθούν ένα μοντέλο ανάπτυξης που θα είναι αποτέλεσμα των συνθηκών που ισχύουν σε κάθε χώρα και σίγουρα όχι αποτέλεσμα επιβολή άλλων ισχυρών κρατών ή των μονομερών επιταγών της αγοράς και του συστήματος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Ζων Αρτούς από την Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Γαλλικής ε, Γερουσίας. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να εκφράσω την ε, ευχαρίστησή μου ε, διότι διοργανώθηκε αυτή η πολύ χρήσιμη συνάντηση μεταξύ εθνικών κοινοβουλευτικών και ευρωπαίων μελών του Κοινοβουλίου. Θα ήθελα όμως να επιμείνω στα ειδικά χαρακτηριστικά της ζώνης του ευρώ. Όπως όλοι μας, ε, εγώ τρέφω ιδιαίτερη συμπάθεια στην αποκαλούμενη κοινοτική μέθοδο. Ε, το πέρασμα στο ευρώ άλλαξε τα δεδομένα ε, για τα κράτη-μέλη που προσχώρησαν στο ευρώ. Από τη στιγμή που προσχωρεί ένα κράτος μέλος στο ευρώ, δεν έχει πλέον τη δυνατότητα νομισματικής προσαρμογής. Βεβαίως το ευρώ είναι το κοινό μας νόμισμα, αλλά τα κράτη που δεν ανήκουν στο ευρώ, που δεν έχουν το ευρώ ως κοινό νόμισμα, μπορούν να προσαρμοστούν, να αλλάξουν τη συναλλαγματική ισοτιμία και αυτό δεν μπορούν να το κάνουν ε, τα κράτη-μέλη του ευρώ και έτσι... Ε, συμμορφώθηκαν με μια πολύ αυστηρή απέτηση. Όταν ε, ε, προσχωρήσαμε στο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, δεν είχαμε προβλέψει τι θα συμβεί σε περίπτωση ατυχήματος. Και σε περίπτωση ατυχήματο, αν θέλετε, η επίπτωση στον εθνικό προπολογισμό είναι εξαιρετικά μεγάλη. Ε, κάθε φορά που θα πρέπει να έχουμε ένα ευρωπαϊκό μηχανισμό σταθερότητα. και κάθε φορά που θα πρέπει να τροφοδοτηθεί με χρήματα αυτό ο μηχανισμό σταθερότητα, τα κονδύλια θα πρέπει να τα προσφέρουν τα μέλη τη ζώνη του ευρώ, θα πρέπει να εισφέρουν, να συμβάλλουν και αυτό έχει τεράστια συνέπεια στον εθνικό του προπολογισμό. Εξού και τεκμηριώνεται η ανάγκη, κατά την άποψή μου, ε, για μια ειδική διακυβέρνηση αποκλειστικά και μόνο για τη ζώνη του ευρώ, πόσο μάλλον που και οι υπόλοιπε χώρες έχουν την τάση να συγκλίνουν και να έρθουν κοντά στο ευρώ και οι Κίνες, οι υπόλοιπε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και βεβαίως δεν θα πρέπει να περιοριστούμε στην ε, παράθεση μόνο ενός ε, ε, ε, την παρουσίαση, αν θέλετε, ενός δημοκρατικού άλοθη. Θα πρέπει οι κοινοβουλευτικοί να εξετάζουν, να ελέγχουν ε, τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η διαχείριση της ζώνης του ευρώ. Ευχαριστώ να δώσω το λόγο στην Ισπανίδα συνάδελφο από την Αρμόδια Επιτροπή του Ισπανικού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ξεκινήσω καταρχάς ε, την παρέμβασή μου ευχαριστώντας σας για τη διοργάνωση αυτής της ημερίδας ε, στην οποία συμμετέχουν μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων, ε, μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου. Ήταν πολύ επικοδομητική αυτή η συνάντηση για την εκ των προτέρων συνεργασία που θα πρέπει εμείς να έχουμε εμείς τα Εθνικά Κοινοβούλια βάσει του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Και θα ήθελα να σας εκφράσω δύο προβληματισμούς. Πρώτον, αναφορικά με τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης οποίος αποκαλείται προϋπολογισμός επένδυσης, όπου το Ευρωπαϊκό Διαρθρωτικό Ταμείο και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο τρατεματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο για, την, ε, για τα κράτη-μέλη. Και απευθύνω το ερώτημα στον Επίτροπο Όλη Ρεν. Βοήθεια για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων. Είπατε μάλιστα και προχθές ότι εξετάζεται αυτά τα χρηματικά δοτικά εργαλεία ε, ε, για να τα χρησιμοποιήσετε στην Ισπανία, παρόλο που τυπικά δεν είμαστε επιλέξιμοι γιατί έχουμε περάσει σε στόχο ε, διαφορετικό. Και δεύτερον, ήθελα να μιλήσω για το ευρωομόλογο για θέματα μεταφορών ενέργειας και ψηφιακού, ψηφιακού κόσμου. Θα δίδεται προτεραιότητα στα ευρωομόλογα όταν θα έχουμε να κάνουμε με υποδομές τόσο σημαντικές όπως είναι ο ευρωμεσογειακός διάδρομος, κάτι το εξαιρετικά σημαντικό για την ανταγωνιστικότητα της Ισπανίας και των χωρών που βρίσκονται στη λεκάνη της Μεσογείου. Και από εκεί και πέρα, η δημοσιονομική ε, εξυγίανση και πειθαρχία σίγουρα είναι παράγοντες ανάπτυξης γιατί εγγυώνται την ε, χρηματοοικονομική σταθερότητα αν θέλετε. Όμως δεν αρκούν, θα πρέπει να έχουμε μέτρα αναπτυξιακά. Η δημοσιονομική εξυγίαση υπάρχει. Ερωτώ λοιπόν, εάν στην περίπτωση της Ισπανίας, όπου χθες μάθαμε ότι το έλλειμμα ανέρχεται στο 8,5 και όχι στο 6 ως ποσοστό του ΑΕΠ, έτσι όπως είχε προβλεφθεί. Έχουμε απόκληση δηλαδή 2,5 μονάδων σε σχέση με τις προβλέψεις. Το έλλειμμα είχε προβλεφθεί θα ήταν 6% του ΑΕΠ και είναι 8,5% του ΑΕΠ. Αυτό ε, έχει ε, ε, επίπτωση 4 δις στον προϋπολογισμό. Θα ληφθούν υπόψη αυτά τα κριτήρια ή θα τηρηθεί δημοσιονομική πειθαρχία σε κατά γράμμα, διότι η Ισπανική κυβέρνηση δεν θα μπορέσει έτσι να δρομολογήσει τις απαραίτητες αλλαγές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ να δώσω το λόγο στον ε, συνάδελφο από την Ιρλανδία. Κύριε White, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολλά λέχθηκαν για την αναγκαιότητα της δημοσιονομικής πειθαρχίας και του διεισμού μεταξύ δημοσιονομικής πειθαρχίας και ανάπτυξη. Πολλοί είπαν ότι είναι απαραίτητη η δημοσιονομική εξυγίαση αλλά όχι επαρκή. Και θα συμφωνούσα μάλλον. Ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζω εγώ μετά από αυτέ τι δύο ημέρε συζητήσεων είναι το εξή. Υπάρχει ένα διαφορετικό επίπεδο σαφήνεια όταν μιλούμε για δημοκρατική λογοδοσία, για ε, όλα αυτά να βγούμε, να τα πούμε δηλαδή στο εκλογικό σώμα, που για μας θα σημαίνει και δημοψήφισμα ή μέσω από την συνήθη κοινοβουλευτική διαδικασία, θα πρέπει να έχουμε τα εργαλεία που θα μας επιτρέψουν να τα πούμε πολύ πιο καθαρά στον κόσμο για, το, για τη δεύτερη πτυχή, δηλαδή για τις πολιτικές ανάπτυξης. Διότι περιστρεφόμαστε γύρω από το θέμα αυτό και χθε και σήμερα. Αλλά εάν σας ρωτήσουν ποιες είναι οι πολιτικές ανάπτυξης, αλλά αυτό θα εξαρτηθεί από το ποιον ερωτάτε. Εγώ δεν λέω ότι δεν υπάρχουν πολιτικές ανάπτυξης, άλλωστε ο κύριος Άντορ ανέπτυξε και πριν από λίγο ορισμένες από τις πολιτικές αυτές. Ορισμένοι μιλούν για απαραίτητες διαρθρωτικές αλλαγές. Άλλοι μιλούν για την χρήση οσμοχλών των διαρθρωτικών ταμείων, που δεν είναι το ίδιο πράγμα. Ο πρόεδρος τη Επιτροπή εχθές μίλησε για το 2020. Ο ίδιος όμως είπε ότι έλαβε πρόσφατα επιστολή από 12 χώρες με κοινή επιστολή, σε σχέση δηλαδή με την ανάπτυξη και την αναγκαιότητα τη ανάπτυξη και δεν μίλησε και καθόλου για 2020. Αν βγω εγώ να πάω στους Ιρλανδούς ψηφοφόρους, είτε ευθέως με δημοψήφισμα, είτε μέσω του Ιρλανδικού Κοινοβουλίου, εδώ έχω εγώ το χαρτί αυτό στα χέρια μου, 11 σελίδες ε, fiscal treaty, που μάλλον μπορώ να τους εξηγήσω, γιατί προσφέρει κάποια σαφήνεια, αν και όχι χωρίς αμφιλεγόμενα σημεία. Έχω, ε, μπορώ να έχω στο άλλο μου χέρι και κάτι άλλο για τις πολιτικές ανάπτυξεις για να μπορώ να μιλήσω πολύ πιο ξεκάθαρα στο εκλογικό σώμα, να τους πούμε δηλαδή συγκεκριμένα τι θα κάνουμε για την ανάπτυξη. Αντί να του πούμε ότι αν υποστηρίξετε το ένα έγγραφο, τότε θα έρθει και η ανάπτυξη αργότερα. Ο κύριο Γκαρίγα Πογέδο. Ευρωβουλευτή. Προφανώ είναι απόν. Ο κύριο Ζουέλ. Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων τη Δανική Βουλή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και όλες και όλους τους συναδέλφους για την καρποφόρα συζήτηση των δύο ημερών. Πολλοί συνάδελφοι τόνισαν, το είπα και εγώ σήμερα το πρωί στο πάνελ, ότι ως εθνικοί βουλευτές έχουμε διπλό ρόλο. Έχουμε την υποχρέωση αφενός να υπερασπιστούμε, να εξηγήσουμε το τι συμβαίνει στην Ευρώπη και σε ό,τι αφορά τη δημοσιονομική εξυγίανση αλλά και σε ό,τι αφορά τη δημιουργία απασχόληση, αλλά έχουμε και το δικαίωμα. Δικαίωμα να, συμπεριλα... να συμπεριλαμβανόμαστε στον διάλογο ω εθνικοί βουλευτέ. Και γι' αυτό είναι χρήσιμη η συνάντηση. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι ακόμα δεν έχουμε φτάσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα και γι' αυτό απευθύνω την ερώτηση αυτή προ την Επιτροπή. Διάφοροι ομιλητέ τόνισαν ότι είναι απαραίτητη η δημιουργία απασχόληση για να ξεφύγουμε από την κρίση και νομίζω συμφωνούμε όλοι. Η πραγματική ερώτηση είναι πώς να ερμηνεύσουμε τα πράγματα που περιλαμβάνονται στο Fiscal Compact με τρόπο που να επιτρέψει τη δημιουργία απασχόλησης και ε, ανάπτυξης. Και πιο συγκεκριμένα έχουμε την Annual Growth Survey και τις σχετικές συστάσεις. Νομίζω ότι πρέπει να καταστήσουμε απόλυτα σαφές ότι οι εθνικοί βουλευτές συμπεριλαμβάνονται σε αυτή τη συζήτηση και θα μεταφέρουν την συζήτηση στις εθνικές βουλές. Εγώ είμαι μέλος κυβερνότος κόμματος και είμαι βέβαιος ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κάνει τη συζήτηση με την αρμόδια υπουργό που κάθεται δίπλα σας, αλλά από τη δημοκρατική σκοπιά πιστεύω ότι σε πολλές χώρες πρέπει να διευρυνθεί η συζήτηση. Και βεβαίως ένα μέγεθος δεν ταιριάζει σε όλους και χρειαζόμαστε ε, ωστόσο παρόλα αυτά και κοινέ αρχές. Ποια είναι λοιπόν η στρατηγική απευθύνομαι τώρα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να τα εξηγήσουμε αυτά στους εθνικούς βουλευτές. Αυτή ε, την εβδομάδα γίνεται μια ευρύτατη συζήτηση για την Ευρωπαϊκή Ένωση και ρωτώ ποιος κάνει σωστούς υπολογισμούς, η κυβέρνηση ή η Κομισιόν. Και εάν οι υπολογισμοί αυτοί αποκλίνουν, τότε έχουμε ένα πρόβλημα. Ευχαριστώ λοιπόν πάντως που ήσασταν εδώ και μας επιτρέψατε να διαλεχθούμε. Ευχαριστώ. Για δύο λεπτά ο κύριος Αλεχάνδρος Σέρκας. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Αγαπητέ κύριε Επίτροπε Ερέν, έχω κάποιες ερωτήσεις να σας θέσω. Γιατί ο πολίτης, αλλά και εμείς ως μέλη Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ε, ακούμε να γίνεται λόγος για δημοσιονομική πειθαρχία ε, και μιλούμε πάντοτε για περικοπές και όχι για φόρους να μειωθούν δαπάνες, να αυξηθούν οι φορολογικοί συντελεστές, αλλά να μην διευρυνθεί η φορολογική βάση που είναι ο άλλος εναλλακτικό δρόμος. Στις χώρες που έχουν πληγεί ε, περισσότερο, κύριε Επίτροπε, από την ανάγκη δημοσιονομικής πειθαρχίας, μπορείτε να πείτε ξεκάθαρα ότι είναι ένα πρόβλημα περίκοπο, περίπλοκο. Δεν είναι μόνο θέμα περικοπών, αλλά είναι θέμα και δημιουργίας πλότου η οποία θα διευρύνει και τη φορολογική βάση και άρα θα οδηγήσει σε περισσότερα έσοδα. Και από εκεί και πέρα ήθελα να πω και το εξή. Οι χώρε που εφαρμόζουν αυτά τα προγράμματα προσαρμογή και επειδή το είπε και η Ισπανίδα συνάδελφος, θα πρέπει να μιλήσουμε για το μέλλον των νέων στις χώρες αυτές. Όχι μόνο ε, συμβόλαια και συμβάσεις ε, βραχίας χρονικής διάρκειας χωρίς δικαιώματα, συμβάσεις που χρησιμοποιούνται μόνο για να καλυφθούν, να φύγουν από τους πίνακες της ανεργίας και να μειωθούν κατ' τα ποσοστά ανεργίας. Χρειαζόμαστε δουλειές ποιότητας, δεν χρειαζόμαστε μόνο δουλειές που κάνουν κάποιον να διαγράφεται από το Μητρό Ανεργίας για λίγους μήνες για να έχουν μέλλον οι νέοι αυτοί, για να μπορέσουν να ζήσουν και να μην ε, χρησιμοποιούνται μόνο ως εργαλείο για να βελτιωθούν οι πίνακες των στατιστικών. Είναι ένα πρόβλημα διαρθρωτικό, είναι ένα πρόβλημα επί της ουσίας το οποίο δυναμετίζει τα θεμέλια των κοινωνιών μας στο μέλλον. Ε, πείτε στους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων ότι χρειαζόμαστε δουλειά για τους νέους, αλλά ποιοτική δουλειά, ποιοτικές θέσεις, ποιοτικές θέσεις απασχόλησης. Ευχαριστώ. Η Πρόεδρος, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Θα δώσω το λόγο στην Υπουργό για πέντε λεπτά για να απαντήσει ε, και στη συνέχεια στους επιτρόπους. Ευχαριστώ. Thank you very Καταρχήν σας ευχαριστώ πολύ. Πολλά υπόθηκαν. Και νομίζω πως ε, βασικά πρόκειται για την ισορροπία ανάμεσα στην ε, εξυγίανση και στην ανάπτυξη. Πώς θα λειτουργήσει αυτό. Αν δεν δαπανούμε, τότε από πού θα προέλθει η ανάπτυξη. Αυτό είναι ένα κέριο ερώτημα. Το πιο σημαντικό σε αυτή τη συζήτηση είναι να εξασφαλίσουμε ότι δεν, δεν υπάρχει άμεση φυσική σχέση ανάμεσα στις δαπάνες και στην ανάπτυξη. Γιατί αν, βλέπαμε, αν δούμε το χρέος και που, στα ύψη που έχει φτάσει, ε, τότε θα έπρεπε να είχαμε τεράστια ανάπτυξη μέχρι στιγμής. Έχουμε λοιπόν από τη μια πλευρά το, τη δημοσιονομική συμφωνία, αλλά από την άλλη τι έχουμε. Αυτό που είναι δύσκολο είναι να βρεθούν ε, να βρεθεί μια παρότρινση ε, για την ανάπτυξη Αν κάθε ευρώ μπορούσε να δαπανηθεί για την ανάπτυξη, την παιδεία, την έρευνα, θα ήταν πολύ διαφορετικό πολιτικό έργο. Έπειτα να εξασφαλίσουμε ότι η επόμενη γενιά της αγοράς θα λειτουργήσει και θα λειτουργήσει καλά, χωρίς γραφειοκρατία. Είναι τεράστιο πολιτικό έργο. Ευρωπαϊκή ευρεσιτεχνία, ψηφιοποίηση, υπηρεσίες. Αν όμως μπορέσουμε να δουλέψουμε με όλα αυτά, τότε πιστεύω ότι θα γίνουν πράγματα, γιατί η ενιαία αγορά τα έχει καταφέρει και παλιότερα. Έχει δημιουργήσει εκατομμύρια θέσεις και μπορεί να το ξανακάνει, αν καταφέρουμε να περάσουμε αυτά τα πολύ σημαντικά βήματα. Έπειτα... Δεν υπάρχει ανάπτυξη στην Ευρώπη χωρίς να γίνουν μεταρρυθμίσεις στα εκάστοτε κράτη-μέλη. Όσα μόλις εξέδωσε τις παρατηρήσεις του με μια πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη που αφορά το πώς οι διαθροτικές αλλαγές επηρεάζουν βραχυπρόθεσμα. Και κάτι στο οποίο κατέληξαν εκεί και το οποίο θεωρώ είναι πολύ ενδιαφέρον ότι είναι ότι δεν υπάρχει απαραίτητο ζημιά βραχυπρόθεσμα από μεταρρυθμίσεις που χρειάζονται για μακροπρόθεσμα όσον αφορά την αγορά εργασίας. Και κάτι το οποίο όλοι σκέφτονται, η ανεργία, συζητήθηκε στο Κοινοβούλιο πριν από λίγες εβδομάδες στο Στρασβούργο. Συζητήθηκε στη συζήτηση με τους κοινωνικούς εταίρους για τις μακροοικονομικές ανισορροπίες. Το συζητήσαμε και σήμερα εδώ. Νομίζω πως είναι πολύ σημαντικό να ακούσουμε τα όσα είπε η Κομισιόν, ότι δηλαδή το Συμβούλιο έχει κάνει πολύ έντονες συστάσεις στα κράτη-μέλη Διάφορε συναντήσεις θα γίνουν τον Απρίλιο ώστε όλα αυτά να συζητηθούν στην ημερήσια διάταξη και πάλι θα είναι δύσκολα γιατί το να δοθεί πρόσβαση στους νέους στην αγορά εργασία είναι πάρα πολύ δύσκολο. Σημαίνει κατάρτιση, επαγγελματική κατάρτιση, οτιδήποτε, ώστε να έχουν μια ευκαιρία. Το πιο σημαντικό πάντως σήμερα είναι να εξασφαλίσουμε ότι η εξυγένση δεν θα μείνει πίσω. Γιατί χωρίς την εξυγένση δεν θα υπάρξει εμπιστοσύνη και αυτοπεποίθηση που χρειάζεται ότι δηλαδή οι πολιτικοί μας έκαναν τις σωστές επιλογές και μπορούμε ε, και θα κάνουν και τις σωστές επενδύσεις στο μέλλον. Χρειαζόμαστε ένα χρηματοπιστωτικό τομέα, ο οποίος να είναι υγιής, ρυθμισμένος ε, και να έχουμε τις απαραίτητες, το απαραίτητο input με χαμηλά επιτόκια για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Χωρίς αυτές δεν θα έχουμε αύξηση των θέσεων απασχόλησης στην Ευρώπη και άρα δεν θα έχουμε και ανάπτυξη. Αυτό που χρειάζεται είναι μια συμμαχία για να κάνουμε αυτή τη δύσκολη, σκληρή δουλειά. Πολλοί ε, πολιτικοί ε, συμβιβασμοί θα χρειαστεί να γίνουν από το Συμβούλιο, την Κομισιόν, τα Εθνικά Κοινοβούλια, ώστε να εξασφαλίσουμε πώς θα λειτουργήσει όλη αυτή η προσπάθεια. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Υπουργέ, ο Επίτροπος. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. για την ερώτηση του Ισπανού, της Ισπανίδος, της Ισπανίδας βουλευτού, κυρία Σάντσες, για τους δημοσιονομικούς στόχους της Ισπανίας. Θα το απαντήσω αυτό γιατί είναι από τα κέρια θέματα για την ε, δημοσιονομική, ευρωπαϊκή δημοσιονομική πολιτική, αλλά βεβαίω και για την Ισπανία και για την οικονομική της πολιτική, την δημοσιονομική της βιωσιμότητα και οικονομική ανάπτυξη. Πρώτα, χρειαζόμαστε πλήρες πληροφορίες για όλες τις ε, δυσκολίες, ας πούμε, όλα τα ολιστήματα που υπήρξαν ε, τον προηγούμενο χρόνο. Δεύτερο, χρειαζόμαστε πλήρη πληροφορία, πλήρες, ε, πλήρες πληροφορίες για τον σχεδιαζόμενο προϋπολογισμό και για τα σχεδιαζόμενα μέτρα δημοσιονομικής εξυγίανσης για φέτος, για το 2012, καθώς συζητούμε δηλαδή τον φετινό προϋπολογισμό του 2012. Αυτή τη στιγμή θα έχουμε τις πληροφορίες αυτές και αναμένω να τις έχουμε μέσα στη διάρκεια του Μαρτίου, τις επόμενες εβδομάδες, θα καταστεί απαραίτητο να εξετάσουμε εάν είναι αποτελεσματική η δράση που αναλαμβάνει η Ισπανία για να εξασφαλίσει την βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών στην Ισπανία. Το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης δεν είναι ανόητο. Δίνει, ε, ε, στοχεύει ιδιαίτερα στην βιωσιμότητα των ε, δημοσίων οικονομικών και αυτός είναι και ο δικός μας στόχος όταν κάνουμε την αξιολόγηση. Θα σας παραπέμψω στα όσα προεβδομάδος την προηγούμενη Τρίτη δηλαδή, αποφάσισε το Συμβούλιο ΕΚΟΦΗΝ με ομοφωνία συμπεριλαμβανομένου του εκπροσώπου δηλαδή της Ισπανικής κυβερνήσεως. Το Συμβούλιο ΕΚΟΦΗΝ επανεπιβεβαιώνει ότι όλες οι χώρες μέλη θα πρέπει να συνεχίσουν να σέβονται τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τους κανόνες του Συμφώνου Σταθερότητας και Αναπτύξεως με τους αυτόματους σταθεροποιητές στην πορεία προς διαρθρωτικές προσαρμογές με ταυτόχρονη διατήρηση της βιωσιμότητας των δημόσιων οικονομικών. Αυτή είναι, αυτή, αυτή η βάση, αυτό είναι το μέτρο που θα χρησιμοποιήσει η Ευρωπαϊκή Αξιολόγηση για τα ισπανικά μέτρα και θα επανέλθουμε στο θέμα όταν θα έχουμε πλήρη πληροφόρηση για όλες τις ε, ε, δημοσιονομικές ολιστήσεις του περσινού χρόνου καθώς και για τα σχέδια του προπολογισμού φέτος. Δεύτερο, σε ό,τι αφορά την ερώτηση του κυρίου Ντέιλι, Ιρλανδού βουλευτού, σχετικά με τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αναφορικά, αν κατάλαβα καλά, με τις αποφάσεις που λήφθηκαν ή που σχεδιάζονται για τον τραπεζικό τομέα στην Ιρλανδία και το οικονομικό σύστημα της Ιρλανδίας. Βεβαίω η Κεντρική Τράπεζα θα έπρεπε να μιλήσει για λογαριασμό της, διότι εγώ σέβομαι την ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, σύμφωνα άλλωστε και με την κατανομή έργου που ακολουθούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύω πάντως ότι είναι σημαντικό, ήταν μάλιστα κρίσιμο για την επιτυχία του προγράμματος Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνού Νομισματικού Ταμείου για την Ιρλανδική Κυβέρνηση, το σχέδιο αναδιάρθρωσης του τραπεζικού τομέα στην Ιρλανδία να παίξει και κεντρικό ρόλο. Γνωρίζετε γιατί. Στην Ιρλανδία καταρχήν δεν ήταν δημοσιονομική η κρίση, ήταν τραπεζική, η οποία ωστόσο οδήγησε σε δημοσιονομική κρίση. Και γι' αυτό πρέπει να αναζητήσετε τις αιτίε του κακού. Γι' αυτό η αναδιάρθρωση και η ανακεφαλαιοποίηση του τραπεζικού τομέα πρέπει να, είναι, πρέπει να γίνει οπωσδήποτε. Από το πρόγραμμα 35 δις ευρώ με 25 δισεκατομμύρια ευρώ ως baseline σενάριο και τα τελευταία νούμερα που είδα εξακολουθούν να είναι κάτω από αυτό το βασικό σενάριο που ήταν απαραίτητο τόσο για την ανακεφαλαιοποίηση του Ιρλανδικού τραπεζικού τομέα και βέβαια για την παράλληλη αναδιάρθρωσή του. Και αυτό, είπα, ήταν ουσιώδες για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην Ιρλανδία, που ακόμα βέβαια βρίσκεται καθοδόν, αλλά σιγά σιγά έρχεται και είναι απαραίτητο για την ανάκαμψη της Ιρλανδικής οικονομίας, διότι χρειάζεστε υγιές τραπεζικό σύστημα για να μπορέσει να ανακάμψει η οικονομία. Για την εκπρόσωπο της Κύπρου που ρώτησε για το ελληνικό πρόγραμμα και συμφωνώ ότι πρέπει να ρίξουμε ε, ιδιαίτερο βάρο και στην δημοσιονομική εξυγίανση και στην πρόθεση της ανάπτυξης και της απασχόλησης. Ωστόσο, α μην λησμονούμε ότι το οικονομικό, το ελληνικό οικονομικό μοντέλο την προηγούμενη δεκαετία δεν ήταν βιώσιμο. Ήταν σαφές ότι διαρκώς δαπανόνταν παραπάνω χρήματα από όσα παράγονταν. Και ε, φτάσαμε ε, σε έλλειμμα του 15% του ΑΕΠ και έχουμε τώρα, έχετε δίκιο μάλλον τώρα, ότι τώρα δίνουμε, πρέπει να δώσουμε πολύ περισσότερο βάρος στην αύξηση της ανάπτυξης, της μεγέθυνσης της ανάπτυξης. Και γι' αυτό προσφέρει τεχνική υποστήριξη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μαζί και με άλλες χώρες μέλη, ώστε να μπορέσει η Ελλάδα να αναδιαρθρώσει τη δημόσια διοίκησή της. και για παράδειγμα σε τομείς όπως η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, η δημιουργία ενός φορολογικού συστήματος που να είναι έντιμο και δίκαιο, γιατί όπως γνωρίζετε στην Ελλάδα η φοροδιαφυγή είναι ένα υπερβολικά διαδεδομένο φαινόμενο και πρέπει να αντιμετωπιστεί μέσα στα πλαίσια του συνολικού αυτού πακέτου. Είναι πάρα πολλές οι ερωτήσεις βέβαια, δεν θα μπορέσω να απαντήσω σε όλες. Ήθελα μόνο να πω όσον αφορά τις, αιτήσεις, ε, ερωτήσεις μάλλον ε, Ιρλανδών και Δανών συναδέλφων ότι η νέα δημοσιονομική συμφωνία, η Fiscal Compact, είναι σημαντική, αλλά ταυτόχρονα εγώ θεωρώ ότι είναι και μια βαθιά πολιτική δέσμευση από πλευρά των κυβερνήσεων αλλά και των εθνικών βουλών για μια δημοσιονομική σοφροσύνη και βιωσιμότητα. Και ταυτόχρονα στην πράξη η εφαρμογή θα γίνει με την δευτερογενή νομοθεσία με το λεγόμενο six-pack με την ενισχυμένη οικονομική διακυβέρνηση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πίτροπε. Ελάχιστα λεπτά μας μένουν ακόμη με την συνδρομή των διερμηνέων και γι' αυτό θα δώσω σε εσάς κύριε Πίτροπε το τελικό λόγο. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, θα ήθελα σύντομα και εγώ να αντιμετωπίσω τα θέματα της αναπτύξης της απασχόλησης και της Ισπανίας, που είναι το πιο, η πιο σημαντική χώρα σε αυτή τη στιγμή στο χαρτοφυλάκιό μου. Αλλά η Ιρλανδία είναι πάρα πολύ δύσκολη υπόθεση, αλλά αυτή τη στιγμή η Ισπανία είναι αυτή που έχει τις χειρότερες στατιστικές και αντιμετωπίζει τις σπουδαιότερες προκλήσεις. Να εστιάσω σε λεπτό την προσοχή μου στο θέμα της ε, ανάπτυξης, διότι και το ευρύ κοινό σε αυτό εστιάζει. Είναι σημαντικό νομίζω να διαφοροποιήσουμε ανάμεσα στις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμε προκλήσεις της οικονομικής ανάπτυξης. Πώς θα αναζωογονήσουμε την οικονομία, πώς θα ξανανάψει η μηχανή και το σωστό μείγμα φορολογικής πολιτικής ε, και δικοδόμησης δυνατοτήτων παίζουν και ρόλο κλειδί. Εφόσον στην Ευρώπη έχουμε τόσο αλληλένδετες ε, οικονομικούς μηχανισμούς, είναι πολύ σωστό να λύσουμε τις προβληματικές ε, περιπτώσεις και να μην υποβαθμίσουν αυτές το δυναμικό του συνόλου της ευρωπαϊκής οικονομίας. Κατά τη γνώμη αυτές είναι οι βραχυπρόθεσμες αλλά το θέμα είναι να μην επιτρέψουμε να θυσιαστεί το μακροπρόθεσμο δυναμικό και οι ανθρώπινοι πόροι που είναι τόσο σημαντικοί για τη μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη ή προς χάρη μιας βραχυπρόθεσμης προσπάθειας σταθεροποίησης. Και γι' αυτό ταυτόχρονα ενώ δουλεύουμε για την δημιουργία βιώσιμης ανάπτυξης βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα, πρέπει ταυτόχρονα να επενδύσουμε στους ανθρώπινους πόρους και να μην επιτρέψουμε ένα υψηλό επίπεδο απασχόληση να συνεχίζεται και να μετατραπεί σε διαρθωτική ενεργεία, γιατί αυτό υποβαθμίζει τη δυνατότητα απασχόλησης των, του εργατικού δυναμικού ε, και επιφέρει τον κίνδυνο μιας χαμένης γενιάς και από αυτό θα χάσει το σύνολο της ευρωπαϊκής οικονομίας και της ευρωπαϊκής κοινωνίας. Αν λοιπόν δεν αναφερθούμε ρητά, δεν αναφέρονται μόνο ρητά αυτό, αλλά τα συγκεκριμένα σημεία συνδέονται με το πρόγραμμα που αποκαλείται Στρατηγική Ευρώπη 2020 ένα άλλο σημαντικό σημείο σε αυτό το τομέα που δεν μπορεί να απαντηθεί σε, σε εθνικό επίπεδο χωριστά, αλλά από κοινού σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να ενεργήσουμε, είναι η εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς. Είναι μια από τις πρωτοβουλίες κλειδιά που έχουμε και που θα συμβάλλει επίσης στην αποκατάσταση της ανάπτυξης. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να βελτιώσουμε την λειτουργία των διευθυντικών ταμείων ως επενδυτικών μέσων. Γι' αυτό και ε, είναι τόσο σημαντικό να συνδεθούν στενότερα τα δημοσιονομικά μας μέσα με τις επενδύσεις, γιατί χωρίς τέτοια μέσα ευρωπαϊκού επίπεδου μπορεί να υπάρξει αντίφαση ανάμεσα στην οικονομική διακυβέρνηση και τις δυνατότητες χειρισμού αντιμετώπισης των προκλήσεων της ανεργίας. Στην Ισπανία, όπως σας είπα, έχουμε την πιο, τη χώρα που βρίσκεται στην πιο κρίσιμη κατάσταση με πολύ ψηλό ποσοστό ανεργίας πάνω από το 20%. Αν τα καταφέρουμε την Ισπανία θα μπορούμε να τα καταφέρουμε και με όλε τι άλλες δύσκολες καταστάσεις στην Ευρώπη. Το θέμα είναι νομίζω πως δεν θα πρέπει απλά να πούμε ποιο είναι το ένα αίτιο για αυτή την ανεργία και να χρησιμοποιήσουμε ένα μέσο για να την αντιμετωπίσουμε, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε διάφορα μέσα. Μεταρρύθμιση τη αγορά εργασία είναι ένα μέσο, αλλά μόνο του δεν θα λύσει το πρόβλημα. Πρέπει να δούμε, βρούμε νέου τρόπου για να αναπτύξουμε τα συστήματα κατάρτιση, τη διαβίου μάθηση ε, για να έχουμε πιο ευέλικτο εργατικό δυναμικό. Επίση θα πρέπει να δούμε ότι αυτή η ύφεση οφείλεται και στη λάθος εξέλιξη της βιομηχανικής πολιτικής. Δηλαδή μια οικονομία θα πρέπει να παίξει το ρόλο της για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, όπως είπε και ο κύριος Σέρκας. Και νομίζω πως η Ισπανία πρέπει να χρησιμοποιήσει καλύτερα την δυνατότητα που έχει για ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας. Έχουμε καλά παραδείγματα για το πώς η κοινωνική οικονομία μπορεί να ε, ανταποκριθεί σε πολύ καλύτερε προδιαγραφές, να αποφύγει την ανεργία. Υπάρχουν ε, καλές πρακτικές και μέσα στην ίδια τη χώρα, αλλά που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν ευρύτερα. Ώστε οι, άτυποι, οι άτυπες δραστηριότητες να έρθουν, ε, να ανέβουν στην επιφάνεια, στην φορολογούμενη οικονομία δηλαδή και να φτιάξουν αυτό το παζλ που συμφωνώ μαζί σας είναι πολύ δύσκολο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε, ευχαριστώ όλους και όλες που παρακολουθήσατε. Είμαστε στο τέλος των εργασιών μας. Μόλις ξεκινήσαμε κάτι που θα πρέπει και θα πρέπει αμέσως ίσως να χωριστούμε. Με δύο λόγια να πω ότι τη στιγμή που το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα υιοθετήσει τους μεγάλους προσανατολισμούς που θα καθορίσουν τον προϋπολογισμό των Εθνικών Κοινοβουλίων, είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ήδη κάνει κάποια πράγματα. Μέχρι στιγμή η Επιτροπή ε, Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων διοργάνωνε τέτοιου είδους ε, κοινοβουλευτικές συναντήσεις ε, με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Πρώτη φορά αυτή τη στιγμή έγινε τέτοια διαδικασία με πολλούς ε, αγορητές, με τους προέδρους των τριών θεσμικών οργάνων της Ένωσης, τον προεδρεύοντα της ΕΚΟΦΗΝ, τέσσερις επιτρόπους. Νομίζω πως η κινητοποίηση αυτή επιτρέπει να δώσουμε σε αυτή την ευρωπαϊκή διάσταση να δώσουμε ευρωπαϊκή διάσταση στη συζήτηση που πρέπει να γίνει και να δοθεί έτσι μια νέα όθηση. Δίνουμε ραντεβού για του χρόνου. Λαμβάνουμε υπόψη τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις σας. Ίσως θα πρέπει να φτιάξουμε και ομάδες εργασίας για να δούμε πώς θα αξιοποιήσουμε ακόμη περισσότερο τις δυνατότητες που έχουμε, έτσι ώστε να κρατεθεί ζωντανή η κοινοβουλευτική διάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί τίποτα δεν θα στεφθεί με επιτυχία αν δεν ε, αν γίνεται μόνο και κλεισμένο των θυρών που δεν ε, και δεν έρχεται σε επαφή με τους, ε, τα κοινοβούλια και τους κοινωνικούς εταίρους. Το θυμήσατε και εσείς κυρία Υπουργέ. Σας εύχομαι λοιπόν ε, καλή επάνωδο και ραντεβού του χρόνου. Σας ευχαριστώ πολύ όσους μπορέσατε να μείνετε μέχρι το τέλος των εργασιών μας. Ευχαριστώ και τους ε, αγορητές υψηλού επίπεδου και φυσικά τους διερμηνείς που μας συνόδευσαν όλη την ώρα.